Καλημέρα σε αγαπητοί συνάδελφοι. Μια και το πρόγραμμά μας είναι αρκετά φορτωμένο σήμερα, θα έλεγα να μην χρονοτριβούμε άλλο. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να ευχαριστήσω και τον κύριο Δεκάστρο που με αντικατέστησε προχθές. Ε, πάμε στο πρώτο θέμα της πρωινής ημερήσιας διάταξης που προβλέπει την συνέπεια της ΚΑΠ για τους νέους ε, γεωργούς μέχρι το 2013. Χθες είχαμε μια πολύ σημαντική συνάντηση με πάνω από 500 ε, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα της ΚΟΠΑ ΚΟΖΕΚΑ και όπως υποσχεθήκαμε πριν από ένα εξάμεινο, διοργανώνουμε τη σημερινή συνεδρίαση με εξέχοντες καλεσμένους. Θα ξεκινήσω με την παρουσίαση μιας μελέτης που είχαμε αναθέσει για τους νέους γεωργούς και την εφαρμογή της πολιτικής μετά της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ μετά το 2013. Όπως ξέρετε, θα μπορέσουμε με τα πορίσματα αυτής της μελέτης να εμπλουτίσουμε ε, την ε, εφαρμοστική έκθεση του συναδέλφου Καπούτο με το ίδιο θέμα. Ε, η μελέτη αυτή εκπονήθηκε από μια κοινοπραξία καλεσμένων από τρία ιδρύματα, από το Τσεχικό Πανεπιστήμιο Επιστημών της Ζωής της Πράγας, από το Τεχνολογικό Κέντρο της Τσεχικής Ακαδημίας Επιστημών και το Ινστιτούτο James Hutton από τη Σκωτία. Ε, την μελέτη διαχειρίζεται το πολιτικό Β. Στόχος της έρευνας αυτής είναι η παροχή πληροφοριών για την κατάσταση εφαρμογής της τρέχουσας ΚΑΠ στους μηχανισμούς για τους νέους γεωργούς. Και μάλιστα η ανάλυση περιλαμβάνει και περιγράφει τα βασικά εμπόδια για την έναρξη ε, γεωργικής δραστηριότητας και εξηγεί τα διάφορα είδη εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους εμπειρογνώμονές μας, τον κύριο Λούκα Ζακάτα από το Πανεπιστήμιο της Πράγας και την κυρία Λι Αν Σάδερλαντ από το Ινστιτούτο James Χάτον της Σκωτίας. Ως συνήθως θα ακούσουμε πρώτα τους εμπειρογνώμονές μας που έχουν το λόγο για 20 λεπτά και κατόπιν θα δώσω το λόγο στην Ομίγυριστα και στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ο συνήθως ε, θα έχουμε και συζήτηση με τους ευρωβουλευτές, τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας. Πολύ σημαντικό το θέμα, θα μας το εξηγήσουν όμως καλύτερα οι καλεσμένοι μας. Επίσης, θα ήθελα να καλωσορίσω στην αίθουσα και τους ε, καλεσμένους ε, επισκέπτες ε, του καθηγητού Ντεκάστρο Πρόκειται για επισκέπτες ε, από την και Βόρεια Ιταλία, τους οποίους ε, καλωσορίζω θερμά στην Επιτροπή μας και σας καλώ να παρακολουθήσουν τις εργασίες μας. Θα δώσω τώρα το λόγο στους καλεσμένους μας. Πρώτα το λόγο έχει ο κύριος Ζακάτα. Ή μάλλον αποφασίστε εσείς με τη σειρά θα μιλήσετε. Συνολικά έχετε 20 λεπτά πάντως. Πώς θα κατανείμετε το χρόνο από σας εξαρτάται. Good Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ που μας ε, καλέσατε εδώ σήμερα. Ε, προέρχομαι από το Τσεχικό Πανεπιστημίο Επιστημών Ζωής στην Πράγα και εκπροσωπούμε και το Ινστιτούτο Λιάν στην Σκοτία. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν τα αποτελέσματα για μια έκθεση η οποία εστιάζεται στην εφαρμογή εργαλείων για τους νέους γεωργούς. Πρόκειται για το αποτέλεσμα συνεργασίας ε, πολλών κρατών ε, πάνω από τρεις χώρες. Είχαμε συγκεκριμένα επτά χώρες που συνεργάστηκαν. Ε, σε 20 λεπτά θα ήθελα πολύ γρήγορα να σας παρουσιάσω την, ε, τους στόχους της έκθεσης και τις μεθόδους τις οποίες ε, χρησιμοποίησαμε. Πρόκειται περισσότερο για μια ακαδημαϊκή έκθεση. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω τις απαραίτητες πληροφορίες. Από ακαδημαϊκή σκοπιά υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες που αφορούν σε αυτό που αποκαλούμε πρόβλημα των νέων αργιοργών. Στην έκθεση λοιπόν ε, έχουμε αρκετές σελίδε όπου περιγράφεται αυτό το πρόβλημα και θα ήθελα να σε ενημερώσω λιγάκι σχετικά με το θέμα αυτό. Και μετά ακολουθεί ε, η ουσία του θέματο είναι τα εφαρμοζόμενα εργαλεία και στο τέλο θα εξετάσουμε τα αποτελέσματα όπω ακριβώ τα αναλύουμε στην έκθεσή μα. Και τέλο θα παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν από την έρευνά μα. Και αυτά θα τα παρουσιάσει ο συνάδελφο, η συνάδελφός μου Λιάν Σάδερλαντ. Θα ήθελα λοιπόν να σα υπενθυμίσω ότι βασικό στόχο στόχος της έκθεσης είναι να δούμε πώς ακριβώς ε, τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν ε, την κοινή γεωργική πολιτική και τα εργαλεία για τους νέους γεωργούς, αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται για να δώσουν τη δυνατότητα στους νέους ε, να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στη γεωργία. Αποδώσαμε ιδιαίτερη σημασία στα δομικά αποτελέσματα. Το μεγαλύτερο θέμα που τίθεται είναι ποιε είναι οι ευκαιρίες που υπάρχουν για νέους γεωργούς και αυτούς που νέους έρχονται στη Γεωργία να αρχίσουν να ασχολούνται με τη Γεωργία. Πώ τα διάφορα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Και αυτό λοιπόν σημαίνει ότι στην πραγματικότητα πώ μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να ξεπεραστούν οι δυσκολίε και να αρχίσουν οι νέοι να ασχολούνται με τη μεγεωργία. Όσον αφορά τη μέθοδό μα, ε, διεξαγάγαμε μια ποσοτική ανάλυση χρησιμοποιώντας ε, ε, τις μεθόδους που υπάρχουν, αυτές της Eurostat και μετά εξετάσαμε και τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Και Επίσης κάναμε και μία έρευνα σε 7 επιλεγμένα κράτη-μέλη. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της απόφασής μας να φέρουμε μία ισορροπία ανάμεσα στον προπολογισμό που είχαμε και στο χρόνο για να διεξάγουμε την ανάλυση. Θα μιλήσω λιγάκι για το ιστορικό του προβλήματος των νέων γεωργών. Είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει κανείς το πρόβλημα των νέων γεωργών να το αντιμετωπίσει κάτω από ολιστική προσέγγιση που σημαίνει ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι το πρόβλημα των νέων γεωργών ε, στη Γεωργία δεν είναι μόνο η γύρανση αλλά και άλλα πολύ σημαντικά φαινόμενα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αυτά λοιπόν τα φαινόμενα αφορούν στην αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα. Βασικές τάσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Γεωργία έχουν σχέση με την συγκέντρωση μειώνονται κατά πολύ οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την τελευταία δεκαετία πάνω από 3,5 γεωργικές εκμεταλλεύσεις εξαφανίστηκαν σε αρκετούς υποτομείς της γεωργίας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι το μέσο μέγεθος μιας, μιας εκμετάλλευσης αυξάνεται μεγαλώνει και αυτό σημαίνει όμως ότι για τους νέους γεωργούς απομένει λιγότερη γη. Άρα δηλαδή η κατάσταση όλη είναι πιο ανταγωνιστική για τους νέους γεωργούς. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα έχει σχέση με τη διαδοχή στη γεωργία. Η γεωργία είναι ένα κλασικό παράδειγμα όπου ισχύει αυτή η διαδοχή, δηλαδή με βάση το τι κληρονομεί μια οικογένεια στους από Νομίζω ότι και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν εξετάζουμε το θέμα των νέων γεωργών. Για τη γύρανση έχω να σας δείξω και κάποιες άλλες διαφάνειες και νομίζω ότι υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με το πώς μπορεί να γίνει η διαφοροποίηση ανάμεσα στους νέους γεωργούς και τους νέο εισερχόμενους. Ένα από τα βασικά ερωτήματα και αυτό που βλέπετε έχει σχέση με το πρόβλημα των νέων γεωργών. Ένα πρόβλημα είναι το θέμα της γύρανσης. Βλέπετε τα στοιχεία που δείχνουν την συμμετοχή, το ποσοστό των γεωργών ε, που ε, τα, τις διαχειρίζονται, τις εκμεταλλεύσεις και είναι άνω των 55 ετών. Το ποσοστό των εκμεταλλεύσεων που έχουν η γεωργοί άνω της ηλικία των 55 ετών. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι βεβαίως ότι τα στοιχεία αλλάζουν με το χρόνο. Υπάρχει μια ελαφρά μετατόπιση στα ποσοστά ε, και αυτό κατ' ουσίαν σημαίνει ότι το πρόβλημα των νέων γεωργών κατά κάποιον τρόπο υπάρχει, επιμένει να υπάρχει στη γεωργία. Και αυτό που επίσης έχει σημασία είναι να εξετάσουμε πιο προσεκτικά τους, γεωργικούς, τους τομείς γεωργίας ε, στα διάφορα κρατημέλη. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για την αναλογία ανάμεσα σε νέους και πιο ηλικιωμένους γεωργούς. Για να κάνουμε καλή ανάλυση πρέπει να ξέρουμε πού βρίσκονται οι εκμεταλλεύσεις και πόσο μεγάλες είναι. Γιατί εξ αυτού απορρέουν σημαντικές πληροφορίες για το πώς επίγον είναι το πρόβλημα της γύρανσης. Ενδιαφέρον αυτό το γράφημα και ε, δείχνει ότι υπάρχουν τέσσερα κλάστερ, τέσσερα, τέσσερις ομάδες κρατών μελών που εκεί ποικίλει ε, το κατά πόσο είναι επίγον το πρόβλημα ή όχι. Από τη μια βλέπουμε χώρες που έχουν υψηλό ποσοστό νέων, οι πράσινες ε, χώρες που βλέπουμε δεξιά, εκεί υπάρχει μικρό ποσοστό πιο ηλικιωμένων ε, διαχειριστών εκμεταλλεύσεων. Και από την άλλη πλευρά, ακριβώ την άλλη πλευρά του γραφήματος, έχουμε εκμεταλλεύσεις όπου είναι μικρό το ποσοστό των νέων γεωργών. Σας είπα ότι για να κατανοήσει κανείς ακριβώς πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα της γύρανσης πρέπει να εξετάσει μια συγκεκριμένη κατάσταση σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ο διαχωρισμός ανάμεσα σε νέους γεωργούς και νέο εισερχόμενους. Αν δείτε λιγάκι την έκθεσή μας θα διαπιστώσετε ότι η συζήτηση, ανάμεσα, η συζήτηση που αφορά στην υποστήριξη των νέων γεωργών είναι αρκετά περίπλοκη, γιατί δεν είναι όλοι νέοι Γεωργοί εισερχόμενοι. Δηλαδή σας είπα ότι οι νέοι Γεωργοί είναι συνήθως ε, διάδοχοι, έχουν κληρονομήσει την εκμετάλλευση από την οικογένειά τους. Ε, υπάρχει λοιπόν μια τυπολογία που δείχνει τι ακριβώς συμβαίνει με όσους νεοεισέρχονται στη Γεωργία. Ποιο είναι το υπόβαθρό τους. Διαπιστώνεται ότι ε, τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα από το πώς θα ορίσουμε την ομάδα στόχο για να την υποστηρίξουμε. Πάμε στο πώς έχει αυτή τη στιγμή η κατάσταση σε σχέση με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Πυλώνας 1. Ε, πληρωμές σε νέους γεωργούς. Ε, το τι ξεκίνησε μετά το 2013, μετά τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Αυτά αφορούν τον πυλώνα υπαριθμών 1. Και υπάρχουν και μέτρα που έχουν στόχο με πέντε συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την υποστήριξη των νέων γεωργών. Στη δική μας την έρευνα προσπαθούμε να κάνουμε αναλύσεις χρησιμοποιώντας ποσοτική προσέγγιση, να βρούμε τις διαφορές και πώς τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται διαφορετικά σε επιλεγμένα κράτη-μέλη. Σε εκείνα δηλαδή τα οποία στην ανάλυση μας παρουσιάζονται στον χάρτη ε, και παρουσιάζονται επίσης και στην έκθεσή μας με περισσότερες λεπτομέρειες. Υπάρχουν βασικές πληροφορίες για τις πληρωμές σε νέους γεωργούς υπό τον πυλώνα 1. Αυτή τη στιγμή περίπου το 4% ε, των ε, ετούντων για βασικές πληρωμές έχουν υποφεληθεί από τις πληρωμές για τους νέους. 12% είναι στην Τσεχία, αυτοί έχουν υποφεληθεί οι νέοι σε εμά. Τα κράτη-μέλη έχουν δυνατότητα να αποφασίσουν μόνα τους για τις ε, προϋποθέσεις ε, που ορίζουν και οι προϋποθέσεις ε, για να καταβληθούν οι πληρωμές στους νέους γεωργούς. Στα, τα περισσότερα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν το ανώτατο όριο δηλαδή 90 εκτάρια είναι το ανώτατο όριο για να μπορεί μια γεωργική εκμετάλλευση να υποβάλει αίτηση ο ιδιοκτήτης ως νέος γεωργός. Λίγα είναι τα κράτη που προσφέρουν αυτή την ε, ενίσχυση σε μικρότερες εκμεταλλεύσεις. Βεβαίως, στην έκθεσή μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς συγκεκριμένα κρατημέλια αποφασίζουν να εφαρμόσουν αυτό το μέτρο και τι τους αλλαγές έχουν λάβει η χώρα. Ας πάμε τώρα στον δεύτερο πυλώνα. Όπως σας είπα, πρόκειται ε, η προτεραιότητα παραθυμών 2, εστιάζουμε σε νέους γεωργούς, ε, η ανάλυση που κάναμε μας κατέδειξε με απόλυτη σαφήνεια ότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετική προσέγγιση για το πώς διανέμουν και ιεραρχούν την υποστήριξη στους νέους γεωργούς πάντα σε σχέση με τα μέτρα που διατίθενται. Εδώ στον πίνακα βλέπουμε ότι κατ' ουσίαν υπάρχουν τέσσερις ομάδες κρατών μελών τις οποίες και αναλύσαμε στην έκθεσή μας. Και βλέπετε επίσης πόσο διαφορετικός είναι ο προπολογισμό τα κονδύλια που δίδονται στους νέους γεωργούς βλέπουμε ότι υπάρχει μια ομάδα κρατών μελών που αποφάσισαν να υποστηρίξουν τους νέους γεωργούς να δώσουν πάνω από 10% από τον προεπλογισμό τους της περιφερειακής πολιτικής για να τους στηρίξουν. Δεξιά βλέπετε τα κράτη-μέλη και τις περιοχές που αποφάσισαν να προσφέρουν υποστήριξη ε, στο πλαίσιο της υπάρχουσας, ε, του υπάρχοντος προπολογισμού για την περιφερειακή πολιτική. Υπάρχει βέβαια ένα στοιχείο το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι διαφορές που υπάρχουν. Ε, γιατί βλέπουμε ότι εδώ στον πίνακα υπάρχουν πάρα πολλές διαφοροποίησεις ανάμεσα και στις χώρες ε, και στις ε, περιοχές. Ε, το σημαντικότερο μέτρο είναι το επαρτμόν 6. Είναι το μέτρο εκείνο που κατ' ουσίαν αφορά στο 80% του προπλογισμού P2B, όπως βλέπουμε, και Νομίζω ότι είναι σημαντικό εργαλείο για να αντιμετωπιστεί το θέμα των νέων γεωργών στη γεωργία. Το μέτρο υπαριθμών 6.1 ε, εφαρμόζεται και αυτό διαφορετικά στα διάφορα κρατημέλη. Μπορείτε να καταφύγετε στην έκθεση να δείτε ποιες είναι ακριβώς οι λεπτομέρειες ε, ε, συνήθως οι ίδιες οι χώρες μπορούν να αποφασίσουν για τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, να ορίζουν μόνα τους τα κριτήρια, ποιο είναι το ελάχιστο μέγεθος εκμετάλλευσης που θα στηρίζεται, αλλά και το μέγιστο μέγεθος εκμετάλλευσης. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται να υπάρχει ένα επιχειρηματικό πλάνο ε, το οποίο ε, να καταδεικνύει το τι θα γίνει με την εκμετάλλευση τα επόμενα έως και πέντε χρόνια. Και πάλι σας λέω ότι τα διάφορα κρατημέλια απαιτούν διαφορετικά κριτήρια για να εφαρμόζεται το επιχειρηματικό πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα των εφαρμοστέων μέτρων. Καταρχήν έχουμε μια ομάδα στόχο και από τις συζητήσεις που κάναμε σε αυτές τις επιλεγμένες 7 χώρες Εξαιτία του γεγονότο ότι δεν έχουμε διαθέσιμα ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα, γιατί από το χρόνο εφαρμογή ε, των μέτρων αυτών δεν πέρασε αρκετό χρόνο ώστε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και ποσοτικοποιημένα. Ε, συζητήσαμε με νέους γεωργούς, άλλους γεωργούς, ε, συμβούλους πολιτικής, εκπροσώπους γεωργών στις επιλεγμένες 7 χώρες και προσπαθήσαμε να διαπιστώσουμε ποια ήταν τα αποτελέσματα των μέσων αυτών από την άποψη των συμφεροντούχων. Εντοπίσαμε λοιπόν διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι εισερχόμενοι. Μια και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι μας παρήχαν τις σχετικές πληροφορίες, πρόσβαση στη γη, διάφορες τάσεις που περιγράφονται στην έκθεση που αντιμετωπίζουν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, πρόσβαση στο κεφάλαιο, στο δανεισμό, τα θέματα της ανταγωνιστικότητας όταν ε, είναι εισερχόμενοι ε, και οι μικρές εκμεταλλεύσεις επίσης οι δεξιότητες που χρειάζονται για τη διαχείριση μιας ε, αγροτικής εκμετάλλευσης. Ποικίλουν τα προβλήματα λοιπόν, υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση. Τώρα, από την ανάλυση μας προέκυψαν ε, οι βασικές προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζουν οι Η πρόσβαση στη γη, σε ποιοτική γη είναι πολύ περιορισμένη, γιατί οι γεωργικές εκτάσεις γίνονται όλο και πιο ακριβές, οπότε οι υπάρχουσες ενισχύσεις, ε, η ενίσχυση των νέων γεωργών και τα μέτρα του πυλώνα 2 δεν ε, είναι αρκετά για να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα της ε, δύσκολης πρόσβασης στη γη. Βέβαια, η ισχύουσα ενίσχυση ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των νέων γεωργών στις εκμεταλλεύσεις. Ε, γιατί εποφελούνται από δίκτυα συμβούλων και λαμβάνουν την τεχνογνωσία για τη σωστή διαχείριση μιας αγροτικής εκμετάλλευσης. Ταυτόχρονα ε, λαμβάνουν και ε, στήριξη επενδυτική και χρηματοδοτική, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τους νέους νεαρούς γεωργούς. Τώρα, η εμπειρία των επιλεγμένων κρατών μελών. Για τους ενδιαφερομένους, η εφαρμογή των μέτρων του πυλώνα 1 και πυλώνα 2 ήταν πολύ θετική. Τα μέτρα έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό ε, και μάλιστα ειδικά οι επιδοτήσει για τους νέους γεωργούς είναι πολύ δημοφιλείς και σε μερικές χώρες ε, υπάρχει τέτοια ζήτηση που δεν ε, υπάρχουν αρκετά κονδύλια για να ικανοποιηθούν όλοι οι ετούντες που ζητούν τέτοιου είδους επιχορηγήσεις. Στην έκθεσή μας ε, και στη μελέτη μας θα βρείτε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες ε, για τα σχόλια των συμφεροντούχων σε ό,τι αφορά την διοικητική κατάσταση, διοικητικές διατυπώσεις και το πώς εφαρμόζεται εμπράκτο στα κράτη-μέλη η ενίσχυση. Αυτά εκ μέρους μου θα ήθελα να δώσω το λόγο στη συνάδελφο, στην Λι Αν Σάδερλαντ. Σε ευχαριστώ Λούκας. Εγώ θα επικεντρωθώ στο τελευταίο πεντάλεπτο που μας έμεινε στις συστάσεις μας αυτές που περιλαμβάνουμε στην έκθεση. Έχουμε συνολικά υποβάλει 14 συστάσεις. Εγώ θα επικεντρωθώ σε τρεις κατηγορίες. Το συνολικό μήνυμα, το γενικό μήνυμα μάλλον, είναι ότι οι ενισχύσεις έτυχαν ε, θερμής υποδοχής. 180.000 ε, νέοι γεωργοί ε, υποφελούνται από τις ενισχύσεις αυτές και εμείς θέλουμε να αυξηθεί ο αριθμός της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τους νεαρούς αγρότες γιατί όπως είπατε υπάρχει υπερβολική ζήτηση και σε μερικές χώρες είναι πιο επιτυχημένη ε, ε, και πολύ επιλέξιμοι οι αιτούντες, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια για να ικανοποιηθούν όλοι. Επίσης, θα πρέπει ε, να καταρρύψουμε το εμπόδιο της πρόσβασης στη γη, που είναι το μείζον πρόσκομα για τους νέους γεωργούς. Και μάλιστα και η ιδιαίτερη ομάδα που έχει συσταθεί έχει εντοπίσει το πρόβλημα αυτό της πρόσβασης στη γη. Ε, καταρχήν, ε, θα πρέπει να επανεξεταστεί η δομή των άμεσων ενισχύσεων. Ε, και αν λάβουμε υπόψη το θέμα της δύσκολης πρόσβασης της γη, θα διαπιστώσουμε ότι οι παλιότεροι γεωργοί δεν θέλουν να μεταβιβάσουν τη γη γιατί τη θεωρούν ως ένα συνταξιοδο... μια συνταξιοδοτική εγγύηση. Και η τιμή των γεωρικών εκτάσεων αυξάνεται εξαιτίας της σύνδεσής τους με τις άμεσες ε, ενισχύσεις που στηρίζονται στη στραματική ενίσχυση. Θα πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε κάποια ε, τέτοια συστήματα ε, πρόσβασης στη γη. Θέλουμε να αυξήσουμε την ε, κινητικότητα και από τους φιλαθροφικούς οργανισμούς και από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Έχουμε ε, εκολαπτήρια αγροκτημάτων, κάποιες ε, βοήθειες για την έναρξη επιχειρήσεων, τα land trusts. Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τους πιο ηλικιωμένους γεωργούς να μεταβιβάσουν τις εκμεταλλεύσεις τους. Και φυσικά θα πρέπει να εξετάσουμε και πιο ίσως άμεσες χρηματοδοτήσεις. Το δεύτερο ζήτημα που ανέφερε και ο Λούκας είναι η διάκριση μεταξύ των νεαρών, νέων γεωργών και των νέων εισερχόμενων. Ε, το ηλικιακό όριο που χρησιμοποιείται είναι τα 40 έτη. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραταθεί μέχρι τα 45 για να χαρακτηρίζεται ένας γεωργός ως νέος και χρειάζεται και δύο δεκαετίες για να συγκεντρώσει κανείς τους πόρου και να ξεκινήσει μια βιώσιμη αγροτική εκμετάλλευση. Επίσης, ε, θα πρέπει να δούμε το σκοπό των ενισχύσεων. Αν σκοπό είναι των ενισχύσεων να ενθαρρύνουν του νέου και να του προσελκύσουν στη γεωργία, τότε θεωρούμε ότι μια πενταετία δεν είναι το σωστό όριο για την πρόσβαση στις ενισχύσεις. Και το λέω αυτό γιατί ένας νέος, ιδιαίτερα όταν έχει γεωργικό υπόβαθρο, θα αρχίσει να συγκεντρώνει πόρους πολλά χρόνια πριν ε, την έναρξη, την επίσημη έναρξη της γεωργικής εκμετάλλευσης. Θέλει να δημιουργήσει ένα ζωικό κεφάλαιο, για παράδειγμα, και γι' αυτό χρειάζεται ε, χρόνο. Μερικές φορές έχουμε ε, εποχιακή βόσκηση. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και η πενταετία είναι προβληματική σε ό,τι αφορά το ανώτατο όριο για το, το επίπεδο των ενισχύσεων που μπορεί να, να ληφθεί από ένα γεωργό είναι προτιμότερο κριτήριο από ότι η πενταετής διάρκεια για το δικαίωμα της λήψης ενισχύσεων. Τώρα θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε και τους νέους ερχόμενους. Ε, τα επιχειρηματικά μοντέλα είναι πολύ σημαντικά και με τη συμμετοχή του στα μέτρα αυτά, οι νέοι ενθαρρύνονται να αναπτύξουν δεξιότητες, επιχειρηματικά μοντέλα και θεωρώ ότι οι δεξιότητες αναπτύσσονται ε, επί τόπου στην Ήπεθρο με κατάλληλη κατάρτιση και με ενημέρωση για τις ε, ενισχύσει. Επίσης θα πρέπει να προβλέψουμε και παροχή συμβουλών και νομίζω ότι μέσω της EIP Agri έχουμε κατάλληλα δίκτυα για να βοηθήσουμε τους νέους ερχόμενους. Ε, θα ξεκινήσει το σχετικό μέτρο από τον Ιανουάριο, θα είναι τετραετές, θα εντοπίσει νέα επιχειρηματικά μοντέλα και την διάδοσή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ενημερωθούν και να καταρτιστούν καλύτερα οι νέοι γεωργοί αυτά και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω στις απορίες σας. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τους δύο καλεσμένους εμπειρογνώμονες. Περνάμε στο γύρω των ερωταπαντήσεων. Η πρώτη που ζήτησε το λόγο είναι η κυρία Σένερα. Ευχαριστώ πολύ για την ε, έκθεση αυτή. Για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξετάσουμε το θέμα ε, της ε, προσέγγισης των νέων ε, και της προσέλκυσης των νέων στον τομέα της γεωρίας διότι η Ήπεθρος ερημώνει και ορισμένε περιοχέ πραγματικά έχουν πληγεί σημαντικά, είναι κάποια σημεία εξαιρετικά σημαντικά για μένα. Πρέπει να υπάρχει μια συνοδεία, μια πλαισίωση για ένα νέο κατά τη διάρκεια τη εγκατάστασή του. Να φέρουμε σε επαφή αυτόν που αποσύρεται με αυτόν που ξεκινάει και αυτό είναι σημαντικό. Επίσης είναι πολύ σημαντικό και αναφέρεται άλλωστε ε, το θέμα της πρόσβασης στη γη για τους νέους όλες αυτές οι πτυχές ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Επιπλέον όμως θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποια άλλα θέματα. Δεν ξέρω εάν η λύση είναι να αυξήσουμε την ηλικία ή να επιτρέψουμε μια σταδιακή διαδικασία ενσωμάτωσης. Ε, αυτό που αναφέρατε προηγουμένως ότι οι νέοι ε, σιγά σιγά ε, μαζεύουν κάποια χρήματα για να μην ε, πάρουν μεγάλο ρίσκο σημαίνει ότι και εμείς πρέπει να έχουμε σταδιακή προσέγγιση. Ε, και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο στη Γαλλική είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ε, προσέλκυση των νέων. Δεν ξέρω αν στη μελέτη τη δική σας έχετε διαπιστώσει κάτι αντίστοιχο, αλλά όταν κάποιος κληρονομεί μια εκμετάλλευση και ο, ο πατέρας ή η μητέρα μεταφέρει ε, στον γιο της, ε, ε, τα δικαιώματα πληρωμής, η, η φορολόγηση είναι στάξη στο 15% για αυτή τη μεταβίβαση. Και φανταστείτε, μια μικρή, μια μεσαία εκμετάλλευση με μικρά εισοδήματα ε, με τις τιμές τις πολύ χαμηλές που έχουν αυτή τη στιγμή αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Επίσης ε, το 1 τρίτον περίπου του πριμ ε, της επιδότησης για τους νέους πάει στους φόρους. Ένας νέος λοιπόν, ο οποίο λαμβάνει αυτό το πρίμιο των 22.000 ευρώ, τελικά πληρώνει 5-6.000 ευρώ σε φόρους. Και το πιο σοβαρό είναι ότι αυτό γίνεται στο, το, το έτος ε, της εκκίνησης έναρξης ε, ε, δραστηριότητα. Δηλαδή βάζουμε εμπόδια στους νέους. Δεν ξέρω τώρα αν η ίδια ενίσχυση ε, έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση τελικά της διοίκησης ε, ή ε, του νέου που θέλει να ξεκινήσει αυτή τη δραστηριότητα. Εν πάση περιπτώσει, επεκτάθηκα κάπως, αλλά πραγματικά οι νέοι στη δική μου περιοχή, στη δική μου πατρίδα, τη Γαλλικία, το ζουν πολύ δύσκολα αυτό. Σας παρακαλώ να μην ε, επισημαίνετε τα ίδια προβλήματα συνεχώς ή να μην επαναλαμβάνετε τις ίδιες ερωτήσεις, γιατί μην ξεχνάτε ότι στις 10 θα αρχίσει και δημόσια ακρόαση με το ίδιο θέμα. Και εκεί έχουμε ένα πλούσιο πάνελ. 15 συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο, οπότε ένα, ενάμιση λεπτό το πολύ ο καθένας, παρακαλώ. Ο κύριος Λουαζό. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω έχουμε μια βαθιά κρίση, αλλά η γεωργία εξακολουθεί να προσελκύει του νέου και αυτό ε, είναι πραγματικά εκπληκτικό. Ενώ υπάρχουν τεράστια ελλείμματα, υπάρχουν πτωχεύσει, ε, αλλά οι νέοι ενδιαφέρονται παρόλα αυτά, αλλά έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά εμπόδια. Ε, το πρόβλημα των νέων που δεν προέρχονται από μια ε, γεωργική οικογένεια είναι να βρουν γη. Και για αυτού που έρχονται από οικογένεια είναι κληρονομιά. Ε, Χρειάζεται λοιπόν μια προπολιτική ενίσχυση ε, στην γη αλλά και στην δανειοδότηση. Ε, θα μπορούσε να γίνεται παραδείγματο χάρη ε, δωρεάν η μεταβίβαση. Αυτό αφορά βέβαια κάποιες χώρες, έτσι. Επίσης θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε την υποστήριξη της κατάρτισης ε, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη γη. Επίση, θα πρέπει να βοηθάμε τους νέους που θέλουν να κατασταθούν ε, και να αγοράσουν εξοπλισμό. Ένας ε, ε, γνωστός συγγραφέας λέει ότι η γη έχει πολλά δώρα για τα παιδιά της εφόσον την δουλέψουν. Ο Άλμπερ Ντές έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και για τις ε, δύο εισηγήσει ε, που ακούσαμε. Θέλω να παρατηρήσω το εξής. Εχθές ε, αποφασίσαμε για θέματα που αφορούν και στους νέους γεωργούς και ορισμένα κράτη-μέλη ξέφυσαν την επιθυμία από το 35% να πάμε στο 50% όσον αφορά τις επιδοτήσεις για τους νέους γεωργούς. Και θέλω να γνωρίζω την άποψή σας. Επίσης, εχθές αποφασίσαμε ότι οι νέοι γεωργοί που έχουν αναλάβει την εκμετάλλευση για κάποιο χρονικό διάστημα, ακόμα και αν είναι μικρό αυτό, μπορούν να λαμβάνουν την επιδότηση για πέντε ολόκληρα χρόνια. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για τους νέους γεωργούς. Πιστεύω ότι οι πληρωμές για τον πρώτο πυλώνα δεν βοηθούν να επιτευχθεί ο στόχος, γιατί έχουμε δύο εκμεταλλεύσεις ο ένας ε, νέος ε, παίρνει από τον πατέρα του, από την οικογένειά του, μια εκμετάλλευση που είναι καταπληκτική και έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις, ο άλλος παίρνει μια εκμετάλλευση που είναι στα χάλια της. Και οι δύο όμως παίρνουν το ίδιο ποσό ενίσχυσης. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να καταβάλλονται ενισχύσεις και επιδοτήσεις με βάση και την κατάσταση της εκμετάλλευσης. Εγώ έρχομαι από τη Βαβαρία με 0,2% επιτόκιο μπορούσε κανείς ε, να πάρει στη Βαβαρία δάνειο για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην Κροατία όμως ε, ε, τα επιτόκια είναι και μέχρι 7 και 8%. Τι πιστεύετε λοιπόν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να μην υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Έχω να σας πω και άλλα, αλλά δεν θα ήθελα να ξεπεράσω το χρόνο μου γιατί νομίζω ότι και αργότερα θα έχουμε χρόνο για να μιλήσουμε. Ευχαριστώ κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση της μελέτης. Θα ήθελα απλώς να πω ότι και η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου έδειξε ότι παρά τις υψηλές επενδύσεις ε, στους νέους γεωργούς δεν έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε ακόμη την ανανέωση των γενεών στη γεωργία. Οπότε χρειάζονται περισσότερα κίνητρα και ανάβσματα για τους νέους γεωργούς για να τους ε, επικουρήσουμε. Στην Κροατία οι νέοι γεωργοί έχουν τα ίδια προβλήματα με τους γεωργούς άλλων χωρών σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη γη, αλλά αντιμετωπίζουν και υψηλά επιτόκια στο δανεισμό τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει με διαβουλεύσεις ε, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να βρει τρόπους για να αντισταθμίσει αυτές τις μεγάλες διαφορές στα επιτόκια. Δεν μπορεί ο Γερμανός νεαρός, ε, γεωργός να έχει επιτόκια 2% και ο κράτης να πρέπει να πληρώνει 7% και 8%. Ε, νομίζω επίσης ότι καλό είναι να ε, καταργήσουμε την πενταετή διάρκεια και επίσης ε, να παρατείνουμε στα 45 το ηλικιακό όριο και να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ νέων νερόγιοργων και νεοεισερχόμενων. Επίσης, ε, ως προς τους μηχανισμούς, θα ήθελα να μου πείτε ποια πρόταση προτείνετε καλύτερη και ποια πιστεύετε θα είναι θετική λύση. Και ευχαριστώ τους κυρίους Ντές και που στα πλαίσια του κανονισμού ε, Omnibus κατάφεραν να διαπραγματευτούν ένα καλύτερο πλαίσιο από αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα. Σα ευχαριστώ λοιπόν και αν είχατε κάποιε προτάσει θα ήθελα να τι ακούσω. Ο κύριο Άγνιο. Ευχαριστώ. Ακούστε, αν εθνικοποιούσαμε όλες, όλη τη γη και όλοι οι γεωργοί ήταν δημόσιοι υπάλληλοι δεν πούμε, ε, θα μπορούσαμε να έχουμε αυτά τα προγράμματα, αλλά δεν είναι έτσι η πραγματικότητα, δεν είναι έτσι η ζωή. Πρέπει να ζήσουμε με αυτά που έχουμε. Καταλαβαίνω ότι η Κομισιόν προσπαθεί να κάνει κάτι με τη μεταρρύθμιση. Ε, έχουν, υπάρχουν κάποια περίπλοκα μέτρα. Ποιο είναι νέο γεωργό, σε τι, τι, δικαιούται, δεν νομίζω πως έχει νόημα όλο αυτό το εγχείρημα, κατά τη γνώμη μου. Ε, είναι πολύ ελκυστικό για έναν ε, ηλικιωμένο γεωργό ε, να αφήσει τη γη του σιγά σιγά να, να κάνει τη δουλειά της και μόνο δύο φορές το χρόνο να, το να χάνει την αξία της και κάθε δύο χρόνια απλώς να την κουρεύει. όμως θα θέλαμε να υπάρχει κτηνοτροφία, παραδείγματο χάρη εκεί, αλλά χρειάζεται επιχειρηματικό πνεύμα. Χαίρομαι που υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα ε, στου νέου γεωργού και του καινούριου γεωργού. Ε, εγώ είπα ε, στο γιο μου ότι εγώ ε, θα αποσυρθώ την τάδε ημερομηνία και ο γιος μου το μετράει. Μετράει πότε θα γίνει. θα ήθελα όμως να είμαστε λίγο εδώ κάπως πιο ενεργοί. Πολλοί γεωργοί αυτή τη στιγμή τους αγοράζουν τη γη μεγάλες εταιρείες ε, είναι ο καλύτερο τρόπος για να χρησιμοποιήσει κάποια τα μηχανήματα. Ε, και εκεί χρειάζεται όμως κάποιος διαχειριστής. Ε, υπάρχουν εκεί λοιπόν δυνατότητες για τους νέους γεωργούς να έχουν ένα εισόδημα και να κάνουν αυτή τη δουλειά της διαχείρισης. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με τον προραλήσαντα. Πράγματι θα πρέπει ίσως ε, το πρόγραμμα της Ολλανδικής Οργάνωσης Νέων Γεωργών να το παρατείνουμε. Δηλαδή σε εμά οι νέοι γεωργοί ε, έρχονται σε επαφή με τους ε, συνταξιοδοτούμενους γεωργούς. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, απλά πρέπει τους ανθρώπους να τους φέρουμε πιο κοντά. Δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε συνεχώ νέους κανόνες. Το μόνο που χρειάζεται να σκεφτόμαστε είναι πώς μπορεί να γίνεται η μετάβαση και οικονομικά. Στην Ολλανδία λοιπόν υπάρχουν ε, κοινωνίες, υπάρχουν ε, μορφές συνεργασίας. Μέσα από αυτά μπορεί κανείς να κερδίσει πάρα πολλά. Υπάρχουν πολλοί που ψάχνουν δουλειά. Ειδικά οι νέοι ενδιαφέρονται αρκετοί από αυτούς πάρα πολύ για την παραγωγή τροφίμων, για να ζουν στη φύση. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το προάγουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαντενκάντα Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την παρουσίαση της μελέτης. Ε, τα θέματα που επισημάνατε ακριβώς τα συζήτησα εγώ και με, την, ε, ε, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Γεωργών και με την ε, Ολλανδική Ένωση Νέων Γεωργών. Ε, χρειάζεται μια αναθεώρηση του συστήματος άμεσων ενισχύσεων για να βελτιωθεί η πρόσβαση στη γη, σίγουρα. Πολύ επίκαιρο το θέμα. Επίση, ω προ την αποτελεσματικότητα των κονδυλίων που καταβάλλονται, πιάνουν τόπο γιατί θα πρέπει να δούμε πόσο αποτελεσματική και ποιοτική είναι η ενίσχυση αυτή. Έχετε κάποια ιδέα αν πραγματικά πιάνουν τόπο και πόσο τόπο πιάνουν τα χρήματα που χρησιμοποιούνται. Είναι αποδοτικά αυτά τα κονδύλια όντω. Και επίση, ε, μία καταποκοπή πληρωμή, μήπω είναι πιο αποτελεσματική, λιγότερο αποτελεσματική από άλλου μηχανισμού, άλλα μέσα. Α το εξετάσουμε και αυτό. Και γιατί να μην εξετάσουμε και το συσχετισμό μεταξύ των δεξιοτήτων και τη σωστή αξιοποίηση των κονδυλίων. Γιατί ένας πιο ειδικευμένο ε, και ικανός ε, γεωργός δεν ε, χρησιμοποιεί και δεν αξιοποιεί καλύτερα τα κονδύλια από έναν ανειδίκευτο. Και μήπως θα πρέπει κάποιο τμήμα των κονδύλων να το δαπανίσουμε στην καλύτερη ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον γεωργό, ο κ. Δεκάστρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονές μας, πολύ ενδιαφέρουσες οι ομιλίες τους. Από αυτά που είπε ο κύριος Ντες, να πω το εξή. Εχθές μόλις ε, ψηφίσαμε για το πακέτο για τη δέσμη μέτρων Omnibus. Ε, πρόκειται για έναν κανονισμό επίσης αυτόνομο που αφαιρέσαμε από το κανονισμό Omnibus. Ε, εκεί λοιπόν θέλω να υπενθυμίσω το εξή. Στου νέου, κυρίω στου νέου γεωργού, δώσαμε τη δυνατότητα να έχουν ένα top-up για πέντε χρόνια ανεξάρτητα από το πότε ξεκινάνε την επιχείρησή τους ή όχι. Βλέπετε λοιπόν αυτό είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση και δώσαμε και τη δυνατότητα ε, στα κράτη-μέλη το top up αυτό να το πάνω από 25% σε 50%. Επίσης δώσαμε τη δυνατότητα στο δεύτερο πυλώνα σε όλους τους νέους να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια με έναν τρόπο ε, συνεργασιών, δηλαδή συνεταιρισμοί νέων μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια κάπως σωρευτικά. Αν θέλετε με όλα αυτά ακολουθούμε μια σωστή κατεύθυνση και ίσως εσείς μπορείτε να μας πείτε, να μας κάνετε κάποιες περισσότερες προτάσεις για το τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να προσθέσουμε στην επόμενη κοινή γεωρική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη μελέτη. Δείξατε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι η πρόσβαση στην ε, γη στις ε, γεωργικές εξετάσεις. Νομίζω ως ε, πολιτική καλούμεθα αυτές οι ενισχύσεις για γεωργικές εκτάσεις ε, επειδή δίδονται πολύ φιδωλά να καλέσουμε, να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδυτές γιατί ε, δεν ε, είναι αποτελεσματικά τα μέτρα στο τέλος καταλήγουμε στην επίμορτη γεωργία και αυτό θεωρώ ότι δεν είναι το, η καλύτερη λύση. Η πρόσβαση για νέους είναι αρκετά περιορισμένη. Αναφερθήκατε στην παροχή συμβουλών. Καλή είναι αυτή, αλλά δεν νομίζω ότι αρκεί. Δεν αρκεί η παροχή συμβουλών. Ε, όταν εμφανίζεται ένας ε, νέος γεωργός, ε, αυτομάτως δημιουργούνται νέα προβλήματα και δεν νομίζω ότι λύνονται με την παροχή συμβουλών αυτή η παροχή συμβουλών προφανώς ε, για αυτήν χρειάζεται και ένα συγκεκριμένο οικονομικό πλαίσιο. Αναφερθήκατε στο, στην ηλικία από 40 να πάμε μέχρι και τα 55. Ε, δεν ξέρω αν αυτό ε, είναι θέμα ηλικιακό ή θέμα προϋπηρεσίας γιατί αναφερθήκατε σε κάποιους που κατά το παρελθόν έχουν κάποια άλλη εργασία και εφόσον μιλάμε για έτη ε, το θέμα είναι πότε ξεκινάει κανείς να ασχολείται με τη γεωργία. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι 40-45 ετών και αρχίζουν να ασχολούνται με τη γεωργία σε αυτή την ηλικία. Να δούμε λοιπόν πότε είναι ε, το έτος κατά το οποίο εισέρχονται στη γεωργία. Δείξατε επίσης ε, στατιστικά διαφορές κάτω από 35 και πάνω από 55 σε εμά όταν παραδίδεται μια γεωργική εκμετάλλευση προκύπτουν και κάποια χρόνια όπου συνεργάζεται η παλαιότερη με την νότερη γενιά. Στα στατιστικά σας δεδομένα αυτό το στοιχείο αποκρισταλώνεται ή όχι. Ευχαριστώ κυρία Μαγκίνες. Σας ευχαριστώ. Λίγα σχόλια έχω μόνο. Καταρχήν ε, χαίρομαι και είναι πολύ αναζωογονητικό που ακούμε ότι μερικές από τις μεταρρυθμίσει τη ΚΑΠ είχαν θετικά αποτελέσματα. Βέβαια εντοπίσατε και κάποιε προκλήσει. Σε ό,τι αφορά το σχόλιο σα για το ότι πρόσκομα δημιουργεί πρόσβαση στη γη και που εν μέρει οφείλεται στη διάρθρωση των βασικών ενισχύσεων. Πώς μπορούμε όμως να τροποποιήσουμε αυτή τη δομή των βασικών ενισχύσεων. Επίσης, ε, τι γίνεται με την πιθανότητα ενό μηχανισμού εξόδου από τη γεωργική δραστηριότητα των πιο ηλικιωμένων. Το σκεφτήκατε. Στην Ιρλανδία έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα που διαχειρίζεται η Μόκρονα Φέρμα, η οργάνωση νέων γεωργών και 27.000 εκτάρια, μάλιστα, μεταφέρονται από μία γενιά στην άλλη με 282 συναλλαγές. Αυτό είναι ένας τρόπος ε, συνεργασίας και επαφής των γενεών. Ε, θα μπορούσε να βελτιωθεί βέβαια, αλλά ως σημείο αφετηρίας δεν είναι κακό. Επίσης, ε, τα φορολογικά συστήματα των κρατών μελών, πώς μπορούν να συμβάλλουν και να βοηθήσουν αυτή την ανανέωση των γενεών που επιδιώκουμε στη Γεωργία. Ευχαριστώ. Καπούτο. Ε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους ε, δύο εμπειρογνώμονες ε, για όλα αυτά που μας είπαν, για τις μελέτες τους. Οι μελέτες αυτές κατ' ουσίαν επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες που έχουμε. Κατ' ουσίαν τα τελευταία χρόνια δεν έχουν αλλάξει και πολλά παρά τις ε, προσπάθειες ε, που έχουμε κάνει σε νομοθετικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά ε, δεν συνέβη τίποτα το σπουδαίο. Τα αποτελέσματα ε, δεν είναι εντυπωσιακά. 6% είναι μόνο εκείνοι που είναι κάτω το ηλικία ε, των 35 ετών. Η βασική πρόκληση είναι η πρόσβαση στη γη αλλά και στην πίστη, στην τραπεζική πίστη. Η τραπεζική πίστη είναι καθοριστικό στοιχείο για να μπορούν οι νέοι να διασφαλίσουν ε, ένα μέλλον στη γεωργία. Είναι λοιπόν απόλυτα σαφές ότι θα πρέπει ίσως να αναζητήσουμε νέα μέτρα έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά σημαντική παρουσία των νέων στη Γεωργία. Θέλω να σας πω ότι κάποιες από τις συστάσεις ε, που προέκυψαν από τη μελέτη, ε, αυτές οι συστάσεις περιλαμβάνονται και στη δική μου την έκθεση. Θέλω όμω να κάνω και κάποιες ερωτήσεις. Παρακαλώ ο πρόεδρος να είναι λιγάκι πιο γενναιόδρος απέναντί μου όσον αφορά στο χρόνο. Θα ήθελα να αναφερθώ κυρίω στο εξή. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει περιθώριο παρέμβασης ε, σε θέματα νομοθεσίας ε, για την παροχή πιστώσεων. Αλλά θα ήθελα να εκφράσω κάποιες ιδέες, να σας τις ε, παρουσιάσω για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε κατά πόσον υπάρχουν ε, κάποιες δυνατότητες. Να δώσουμε κίνητρα έτσι ώστε να υπάρχουν νέες δράσεις και να υπάρχει δυνατότητα κινητικότητα σε τραπεζικό επίπεδο. να υπάρξουν νέα μοντέλα, νέα επιχειρηματικά μοντέλα στον γεωργικό τομέα καινοτόμε μορφέ συνεργασία ανάμεσα στου γεωργού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και να υπάρχουν πιο ε, ενεργέ εθνικέ πολιτικέ, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει και καλύτερη πρόσβαση στην πίστη και σε θέματα γης. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτά που μόλις τώρα σας είπα, εσείς συμφωνείτε, γιατί είναι κάτι το ιδιαίτερο κατά την άποψή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ανδριέ. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους ομιλητές για την πολυπιωτική αυτή παρουσίαση. Τέσσερα γρήγορα σημεία. Για το θέμα της συλλογική οργάνωσης των γεωργών υπάρχουν διαφορετικέ προσεγγίσεις από χώρα σε χώρα. Θα ήθελα λοιπόν να εμβαθύνετε κάπω, διότι σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση αλλά και την κληρονομιά, ε, με βάση τι νέες απαιτήσει απασχόληση ε, σε ό,τι αφορά την οικονομική και κοινωνική οργάνωση, ε, υπάρχουν δυνατότητε εδώ να ενθαρρυνθούν, να ενθαρρυνθεί η εγκατάσταση. Δεν ξέρω αν το ψάξατε αυτό επαρκώς. Νομίζω πω είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι αμεληταίο. Για το θέμα της κατάρτισης τώρα. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχουν κάποια σημαντικά ε, διλήμματα. Ε, υπάρχει το θέμα της αγρονομικής κατάρτισης. Ε, συχνά βλέπουμε ότι το παραμελούμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον της και βεβαίως ό,τι έχει να κάνει με τις νέες τεχνολογίες, ε, ε, την επιστημονική πρόοδο, θα ήταν σημαντικό και αυτά τα σημεία να τα εμβαθύνουμε στα πλαίσια της συζήτησης για τη μελλοντική ε, μεταρρύθμιση. Τώρα, βεβαίως, το θέμα ε, του δικαιώματος στη γη δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους να το εμβαθύνουμε και αυτό και για τους νέους, τους καινούριους γεωργούς μάλλον, ε, πρέπει να γίνει ένα σαφής διαχωρισμός μεταξύ των νέων γεωργών και των καινούριων γεωργών. Ε, ε, αλλάζει και η σχέση που έχουμε με τη δουλειά και υπάρχουν όλο και περισσότεροι καινούργοι γεωργοί, όχι απαραίτητα νέοι, και δεν μπορούμε να μην του θεωρήσουμε, να μην τους ε, ε, λάβουμε υπόψη μα αυτού με συγκεκριμένε ενισχύσει. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε, να εξετάσουμε περαιτέρω προτάσει που παρουσιάσατε πριν. Ο κ. Φλάνναγκαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση. Ορισμένα θετικά σημεία, η αύξηση της ηλικία στα 45, ε, καθώς και η ιδέα ότι μπορεί κάποιος να λαμβάνει ένα ποσοστό ενίσχυσης ε, για πάνω από πέντε χρόνια και αυτές είναι καλές ιδέες. Υπήρχε μια έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου ε, στην Επιτροπή Ελέγχου των Συνόρων και προέκυψε τον προπολογισμό συγγνώμη ε, θα πρέπει να κάτσουμε να ακούσουμε διότι είναι απειλείται αυτή τη στιγμή ο προπολογισμό της Γεωργίας και αν το λένε τέτοια πράγματα οι ελεγκτές του Ελληνικού Συνέδριου σημαίνει ότι ε, ε έχουν πιο πολλά επιχειρήματα αυτοί που, είναι, που δεν είναι γεωργοί για να πάρουν τα χρήματα που περισσεύουν. Επίσης ε, πρέπει να υπάρχει μια σωστή τιμή για το προϊόν. Όταν κάποιο θέλει να γίνεται ξυλουργό είτε τεκομωτή, γιατί να ξεκινήσει να το κάνει αυτό όταν δεν μπορεί να βγάλει χρήματα. Επίσης πρέπει να έχει κάποιο πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Ε, δεν μπορεί να υπάρξει κέρδος χωρίς χρηματοδότηση αρχική. Επίσης ο Άλμπερτ Ντες και ο κύριος Ντεκάστρο αναφέρθηκαν στην ε, οδηγία Omnibus ε, και τα πέντε χρόνια του προγράμματος. Πολύ καλό αυτό. Αλλά υπήρξε ένα αίτημα του Συμβουλίου να αλλάξει το κείμενο και αντί για σάλ να λέμε may, να είναι δυνητικό δηλαδή. Μια χώρα δηλαδή να μην δεσμεύεται. Εγώ πραγματικά ε, ντρέπομαι, που αυτό το ζήτησε η χώρα μου μάλιστα και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το ζήτησαν αν είναι, βλέπουν σοβαρά το θέμα της ανανέωσης ε, ε, των, της γεωργίας από ό,τι φαίνεται από τη, τα δικά μας υπουργεία που έχουν τα προβλήματα και όχι από την Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε την υπερβολική διόγκωση των εκμεταλλεύσεων λόγω της συγκέντρωσης. Συνήθως ε, οι συγχωνεύσεις γίνονται σε γειτονικά αγροκτήματα, κάτι που συστηματικά αυξάνει την ε, επιφάνεια των ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Μέσα σε 10 χρόνια έχουν διπλασιαστεί τα μεγέθη, οι διαστάσεις των αγροκτημάτων. Επίσης, ε, επειδή επικεντρωνόμαστε όλο και περισσότερο στην ε, οικονομική πλευρά, θα πρέπει να δημιουργήσουμε άλλα κίνητρα και ενάβσματα για τους νέους για να αναλαμβάνουν γεωργική δραστηριότητα. Δεν μπορούμε να διαφορούμε για το θέμα αυτό. Θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υποβάλουμε το ταχύτερο δυνατό κάποιες προτάσεις, ώστε να κρατήσουμε μια οικογενειακή γεωργία εγκύτητος και ποιότητος, γιατί αν... Ε, μεταβούμε σε γιγαντιές ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα απομακρυνθούμε πολύ από την ουσία μιας αγροτικής εκμετάλλευσης. Ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στους εμπειρογνώμονές μας, τους οποίους ε, παρακαλώ να είναι σύντομοι στις απαντήσεις. Αν καταφέρετε μέσα ένα πεντάλεπτο να απαντήσετε θα ήταν ε, ευχής έργο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Έχουμε καταγράψει τα κύρια σημεία των ερωτήσεών σας και θα προσπαθήσουμε να τα απαντήσουμε εντάχει. Το πρώτο ζήτημα που αναφέρθηκε είναι το φορολογικό. Ε, ιδιαίτερο φόρος κληρονομίας για τη μεταβίβαση, ε, την κληρονομική διαδοχή στα αγροκτήματα. Γνωρίζω από την πατρίδα μου την Τσεχία ότι ε, το θέμα της φορολογίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην Δημοκρατία της Τσεχίας ε, ο φόρος κληρονομιάς ε, ήταν ίδιος με το φόρο στην πώληση σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση ενός αγροκτήματος και κάτι τέτοιο επηρέασε πολύ τον τρόπο διαδοχής ε, στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Πολύ σημαντικό λοιπόν το θέμα ότι η φορολογία επηρεάζει ιδιαίτερως η συνάδελφο, όντω, τα σχόλια ήταν πολύ θετικά για την εκμάθηση, την κατάρτιση και την συγκέντρωση δεξιοτήτων. Θα πρέπει να γίνει επένδυση πριν την έναρξη τη γεωργικής δραστηριότητα με την ε, συσσόρευση εφοδίων και δεξιοτήτων. Και ε, αν ένα επιχειρηματικό μοντέλο παρόλα αυτά δεν είναι προσοδοφόρο, ε, αξίζει να συγκεντρωθούν ε, δεξιότητες και εφόδια και προσόντα. Επίσης, η παροχή συμβουλών είναι πολύ σημαντική ε, και, και όντως πολλές ε, συμβουλές ε, παρέχονται προκειμένου να ενημερωθούν όχι μόνο στην Ιλλανδία αλλά και αλλού στην Αγγλία για τη δυνατότητα μεταβίβασης ή κινητικότητας των γεών και σίγουρα η παροχή συμβουλών βοηθά και η κατάρτιση επίσης εξυπηρετεί για να έχουμε ένα είδος επιχειρηματικής κατάρτισης και στις ε, αγροτικές περιοχές. Η τροποποίηση των άμεσων ενισχύσεων, ε, άλλο βασικό σημείο που προέκυψε από τη συζήτηση. Φάνηκε και από τη μελέτη ότι οι άμεσες ενισχύσεις είναι σημαντικό μέσο για την ε, ε, βοήθεια, την ε, υποστήριξη των γεωργών και έχει γίνει αποδεκτό και από τους ε, διαφερομένους, τους άμεσους δικαιούχους. Είναι όμως σαφές ταυτόχρονα ότι το σύστημα άμεσων ενισχύσεων έχει και αρνητικά αποτελέσματα. Αυξάνει τη τιμή της γης και επίσης δίνει έμφαση στο πρόβλημα της εξόδου γιατί οι άμεσες ενισχύσεις ε, που είναι στρεματικές ε, δίνουν κίνητρα για μη μεταβίβαση στους ηλικιωμένους γιατί οι άμεσες ενισχύσεις αποτελούν σημαντικό ε, τμήμα του εισοδήματός τους. Γι' αυτό είναι απρόθυμη στη μεταβίβαση. Σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση του συστήματος άμεσων ενισχύσεων με τρόπο που να τις καθιστά πιο ευνοϊκές για τους νέους, όντως το ανώτατο είναι προβληματικό ειδικά για τους ε, νέους γεωργούς, ε, καλό θα ήταν τα ανώτατα όρια να μην αποθαρρύνουν ε, τους επενδυτές από την συγκέντρωση γεών. Επίσης, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε εναλλακτικές λύσεις, όπως είναι η βιολογική γεωργία ή οι βραχίες αλυσίδες διανομής. Επενδύοντας λοιπόν και σε αυτά τα είδη γεωργίας με τις συγκεκριμένες προσεγγίσεις, οι νεαροί και οι καινούργοι γεωργοί δυστυχώς ε, δεν επωφελούνται ισότιμα από τους μηχανισμούς. Ε, είναι, ήταν σαφές από την έκθεση και του ελεκτικού συνεδρίου ότι το μείζον πρόβλημα ε, με τις ενισχύσεις για τους νεαρούς γεωργούς είναι το πώς προσδιορίζονται και ποιο θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα αυτής της ενίσχυσης. Εμείς στη μελέτη μας διαπιστώσαμε ότι έχουμε τέσσερι, υπάρχουν τέσσερις γενικοί στόχοι ε, για το μηχανισμό των νέων γεωργών. Και δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν ταυτόχρονα και οι τέσσερις στόχοι. Εξαρτάται από το είδος εφαρμογής που χρησιμοποιούν οι διάφορες χώρες. Πάντως, όντως ε, υπάρχει μια αρνητική εντύπωση για το θέμα αυτό, γιατί δεν είναι σαφές Ποιο είναι ακριβώς ο στόχος των ενισχύσεων για του νεαρού γεωργούς πέραν της αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Γιατί δεν φαίνεται οι ενισχύσει να βοηθούν την υλοποίηση του στόχου της ανανέωσης των γενναιών στη γεωργία. Σε ό,τι αφορά την παρέμβαση στι αγορές, ε, τι κτηματικέ, ε, φυσικά υπάρχουν εθνικά αλλά και ευρωπαϊκές αρχές που προβλέπουν την ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων γιατί και η γη είναι ένα αγαθό όπως και άλλα αγαθά. Πάντως ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα έπρεπε πιο άμεσα να επεμβαίνουν στις κλιματικές αγορές με κάποιες απαιτήσει διαμονής ή άλλους περιορισμούς για τον τρόπο μεταβίβασης των γεών. Έτσι υπάρχουν δυνατά, υπάρχει δυνατότητα για κάποιες επεμβάσεις, αλλά να και τις εθνικές κυβερνήσεις να επιλέξουν τον τρόπο επέμβασης και φυσικά υπάρχουν περιορισμοί. Και το τελευταίο σχόλιο που αφορά τη διαδοχή στα αγροκτήματα. Στην μελέτη μας έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τους διαφορετικούς τρόπους διαδοχής και μεταβίβασης και φαίνεται πόσο περίπλοκο είναι το θέμα λόγω των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, των διαφορετικών παραδόσεων, ε, την οικονομική κατάσταση της γεωργίας και λόγω πολλών άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την διαδοχή και μεταβίβαση. Ίσως ε, θα πρέπει να επανεξεταστεί ε, η ενίσχυση για την πρόορη δεξιοδότηση των γεωργών. Δεν προτείνουμε κάποιες συγκεκριμένες λύσεις στην έκθεση, αλλά ζητούμε απλώς επανεξέταση. Γιατί δεν είναι θέμα μόνο έναρξη γεωργικής δραστηριότητας από τους νέους ή ανάληψη ε, της, ή συνέχιση μιας γεωργικής δραστηριότητας. Το θέμα είναι και οι ηλικιωμένοι να είναι πρόθυμοι να μεταβιβάσουν τις εκμεταλλεύσεις τους στη νέα γενιά. Ναι, να πω ότι βεβαίως είναι μια ανησυχία εξαιρετικά θεμητή διότι επενδύονται κάποια χρήματα και θέλουμε να έχουν επιπτώσει. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όταν εξετάζουμε την παρούσα κατάσταση δεν είμαστε σε θέση να συγκρίνουμε με μια κατάσταση όπου τα χρήματα αυτά δεν είχαν επενδυθεί. Δηλαδή ένα συμπέρασμα είναι ότι τα χρήματα δεν έχουν επίπτωση. Η άλλη επίπτωση, η άλλη, το άλλο συμπέρασμα είναι ότι ο αντίκτυπο είναι ότι παραμένει στο status quo και ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα χωρί αυτή την επένδυση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα και να το εξετάσουμε πιο λεπτομερώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Πραγματικά εξαιρετική. Νομίζω ότι σήμερα έχουμε μια σειρά από ακροάσεις. Ε, έχουμε άλλωστε πρόσβαση και στις, στην παρουσίασή σας, η οποία θα μοιραστεί στα μέλη. Απαντήθηκαν και τα ερωτήματά μας και τώρα θα περάσουμε στην ακρόαση για την εφαρμογή της ε, στρατηγικής πολιτικής για τους νέους γεωργούς και την ε, ανανέωση των γενεών. Και βεβαίως ε, θα έχουμε παρουσιάσει από τον κύριο Γιάννους Βοτσιχόφσκι από το Ελληνικό Συνέδριο που έχει ετοιμάσει μία μελέτη κατόπιν ενός, έρευνας τον είδαμε και προχθές στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και είναι ε, επίσης εδώ μαζί μας να, να παρέμβει ο κύριος Ρόμπλε από το Υπουργείο Γεωργίας της Σλοβενίας. Έχετε 8 με 10 λεπτά για να παρέμβετε. να τι παρεμβάσετε και μετά θα έχουμε ερωτήσεις. 10 λεπτά παρακαλώ. Ο κύριος Βοτσιχόφσκι θα ξεκινήσει και στη συνέχεια ο κύριος Ρόμπλεκ από τη Σλοβενία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Από το 2015 έως το 2017 είχαμε ε, μια μείωση των γεωργών στα 10,7 εκατομμύρια από τα 15 περίπου. Χάσαμε περίπου 4 εκατομμύρια γεωργούς μέσα σε 10 χρόνια το 2005 από το 2015. 400.000 γεωργοί το χρόνο, 30.000 γεωργοί το μήνα, 1.000 γεωργοί τη μέρα, έτσι, μέσα σε μία συζήτηση που κάνουμε εμείς εδώ, σε αυτό το χρονικό διάστημα, 60 γεωργοί εγκαταλείπουν τη γη τους. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Ε, το εξετάσαμε, το είδαμε και στην έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου ε, του Ιουνίου ο υπενθύμησε ο κ. Φλάναγκαν ε, είχε παρουσιαστεί στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου ε, αλλά και στην Επιτροπή Γεωργίας τον Ιούλιο. Θα δείξω μόνο μερικές διαφάνειες με τα βασικά στοιχεία από αυτή την έκθεση. Εδώ διαπιστώνεται το πρόβλημα η μείωση του πληθυσμού των γεωργών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες βλέπετε το μπλε κάτω οι νέοι γεωργοί δηλαδή νεότεροι των 45 έχουν μόλις 21% των γεωργών κάτω των 45. Σχεδόν 80% των Ευρωπαίων γεωργών είναι πάνω από 45 χρονών. Και αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό, το θέμα της ε, γύρανσης ε, του γεωργικού πληθυσμού. Βλέπετε τώρα εδώ σε αυτό το γράφημα για την οικονομική, δημοσιονομική περίοδο 2007-2013 ο πληθυσμός των νέων γεωργών ο αριθμός των νέων γεωργών μειώθηκε από 3,3 εκατομμύρια στα 2,3 εκατομμύρια. Είναι η μπλε γραμμή στο γράφημα. Η κόκκινη γραμμή τώρα δείχνει την αύξηση ε, της μέσης έκτασης από τα 19 εκτάρια στα 44 εκτάρια περίπου. 24 είναι ο μιλητής μάλλον. Είχαμε όμως ε, μια μείωση της συνολικής γης εκμετάλλευσης από τα 57 εκατομμύρια εκτάρια στα 51 εκατομμύρια εκτάρια για την περίοδο 7, αυτή την πταετή. Σε αυτό το γράφημα τώρα βλέπετε το πρόβλημα της γύρανσης ε, των Ευρωπαίων γεωργών. Στη μέση αυτή η κόκκινη γραμμή είναι η κατανομή η ε, ηλικιακή στον πληθυσμό. είναι λίγο κάτω του 40% σήμερα ημέρα οι, οι, οι άνθρωποι νεότεροι του 45. Εδώ βλέπετε τι γίνεται με τους μισθωτούς γενικότερα των ε, εργαζομένων. Το 50% των ε, εργαζομένων είναι κάτω 45. Στον τομέα της γεωργίας όμως, ε, βλέπετε εδώ την πράσινη γραμμή, Μόλις 21%. Είναι εξαιρετικά σοβαρό το πρόβλημα λοιπόν το θέμα της γύρανσης των ε, γεωργών του γεωργικού πληθυσμού. Εδώ ε, βλέπετε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, ενδεχομένως βέβαια να μην μπορείτε να τα δείτε τώρα γιατί είναι μικρά, ε, μικρά τα στοιχεία. Βλέπετε τι σημαίνει σε κάθε χώρα και η κατάσταση διαφέρει, ποικίλει, πάση περιπτώσει, από χώρα σε χώρα. Μόνο δύο κράτη-μέλη έχουν ποσοστό νέων γεωργών κάτω των 35, των 35 είναι πάνω από 10% η Αυστρία και η Πολωνία. Πάνω από 10% γεωργών ε, κάτω από το 35%. Δεξιά βλέπετε τώρα τους γεωργούς ε, άνω των 65 οι πιο ηλικιωμένοι. μόνο σε τρία κράτη-μέλη αυτό το ποσοστό είναι κάτω από 10%. Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία. Σε κάποιες χώρες αυτό το ποσοστό είναι κοντά στο 40%. Στην Πορτογαλία πάνω από 50% των γεωργών είναι άνω των 65%. Επίσης ε, εδώ βλέπετε τα κράτη-μέλη όπου διαπιστώνουμε μία βελτίωση. Είναι σημειωμένη με χρώμα, σημειωμένα με χρώμα αυτά τα κράτη-μέλη, αλλά μιλάμε για μία μειοψηφία. Στην πλειοψηφία των κρατών μελών η κατάσταση το 2013 ήταν χειρότερη από το 2007. Στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, ο πληθυσμός των γεωργών κάτω από το 45 μειώθηκε από το 36% στο 26%. Στη Γαλλία από το 32% στο 28%. Υπάρχει μια μικρή πρόοδος στη Βουλγαρία, στην Πολωνία, στη Σλοβακία, στη Σλοβενία την Ιταλία λίγο, αλλά σε γενικές γραμμές δεν βλέπουμε τον θετικό αντίκτυπο της κοινή γεωργικής πολιτικής σε ό,τι αφορά την ηλικιακή διαστρωμάτωση ε, των γεωργών. Μια σημαντική πληροφορία τώρα. Στον έλεγχό μας, στη μελέτη μας, ε, δεν βρήκαμε καταχρήσεις ή παρατυπίες μεταξύ των γεωργών. Αυτό είναι το πρόβλημα της λογικής της παρέμβασης. Δείξαμε στην έκθεσή μας, δώσαμε παραδείγματα. Ένας νέος Γιώργος με πάνω από 500 εκτάρια λαμβάνει 100.000 ευρώ άμεσες πληρωμές και άλλες 3.000 ως νέος Γιώργος. Εντάξει, ενδεχομένω να τον βοηθάνε και αυτά τα 3.000, αλλά δεν μπορεί να πει κανεί ότι αυτό υποστηρίζει την ανανέωση. Και στην έκθεσή μα υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Νομίζω ότι το συμπέρασμα, το πολιτικό συμπέρασμα, δεν λέω ποια είναι η σύστασή μας, αλλά η μελλοντική κοινή γεωργία θα πρέπει να εξεταστεί όχι μόνο με μια προοπτική 7 ετών, αλλά μια προοπτική 27 ετών. Τι γεωργία θέλουμε, μακροπρόθεσμα. Αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Βοητσοχόφσκι. Θα μελετήσουμε ενδελεχώς ε, το υλικό και τα έγγραφα που μας δώσετε. Και τώρα το λόγο κύριος Ρόμπλεκ ε, από την ε, Σλοβενία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Όπως είπατε, ονομάζομαι Ρόμπλεκ. Έρχομαι από τη Σλοβενία και ε, συμμετείχα σε μια μη κυβερνητική οργάνωση νέων γεωργών και τώρα ε, εφαρμόζω το πρόγραμμα ανάπτυξης ε, της γεωργίας στη Σλοβενία. Παρακολουθώ τα αποτελέσματα της κοινή γεωργικής πολιτικής εδώ και πολλά χρόνια και θα σας παρουσιάσω τις σκέψεις μου για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων της ΚΑΠ από το 2013 και μετά και πώς επηρέασαν τους νέους γεωργούς. Το μείζο ζήτημα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα και το κύριο ερώτημα είναι το κατά πόσο τα νέα μέτρα της ΚΑΠ υλοποιούν το στόχο της ανανέωσης των γενναιών και αν ανταποκρίνονται στο πρόβλημα της γύρασης του γεωργικού πληθυσμού. Για να αναλύσουμε κάποια μέτρα για να δούμε τι συμβαίνει στη Σλοβενία. Η επιλέξιμη γεωργή για το πρόγραμμα νέων είναι 18 με 40 ετών με την κατάλληλη εκπαίδευση και κάποια εμπειρία και δεξιότητες. Στον κύκλο εφαρμογής των μέτρων αυτών αντιμετωπίσαμε τρία μέτρα. Τι χρειάζεται για την δημιουργία μιας γεωργικής εκμετάλλευσης ή για την έναρξη γεωργικής δραστηριότητας, ποιος είναι ο ενεργός γεωργός, ποιος χαρακτηρίζεται ενεργός γεωργός και πώς μπορούμε να προσελκύσουμε τους νέους για να ξεκινήσουν ορικές δραστηριότητες και να παραμείνουν σε αυτές. Πώς θα καταστήσουμε θελκτική λοιπόν την ενασχόληση με τη γεωργία για τους νέους. Έχουμε καταρχήν ε, κατόφλια, ανώτερα και κατώτερα, ε, για τη γεωργία και την κτηνοτροφία και φυσικά θα πρέπει να αποδεικνύονται ε, και οι δεξιότητε και εκπαίδευση. Και μάλιστα η οικονομική ενίσχυση δίνεται σε δύο φάσει: 45.000 ευρώ αν είναι απασχολούμενο ο νερό στο αγρόκτημα και 18.600 ευρώ σε περίπτωση που δεν απασχολείται στη γεωργική εκμετάλλευση. Η δημοσιονομική περίοδος, περίοδος ε, χρηματοδότησης είναι τριετή, 70% καταβάλλεται με την υποβολή τη αίτηση και το 30% με την ε, ολοκλήρωση. Έχουμε κάποια υποχρεωτικά ε, συστήματα συμπληρωματικής ε, ενίσχυσης για τους νέους και περίπου 70.000 νέους γεωργούς, 7% των, ε, του συνόλου των δικαιούχων άμεσων ενισχύσεων και χρησιμοποιούμε το 25% του, της μέσου όρου για τη Σλοβενία και το χρησιμοποιούμε ε, για να φτάσουμε στο μέσο όρο του συνολικού κονδυλίου που δεν πρέπει να ξεπερά το 2% για το συγκεκριμένο μέτρο. Κατά το σχεδιασμό των μέτρων για τους νέους γεωργούς, σύντομα, γρήγορα μάλλον συνειδητοποίησαμε ότι τα μέτρα της ΚΑΠ δεν είναι τα μόνα που υπάρχουν. Ε, χρειαζόμαστε μια πιο σφαιρική συνολική προσέγγιση για την υλοποίηση των μέτρων. Και στο μέτρο για την δημιουργία γεωργικής εκμετάλλευσης θα πρέπει ε, να λαμβάνουν επιπλέον κονδύλια αν εφαρμόζουν κάποια περιβαλλοντικά μέτρα, συμπληρωματική ενίσχυση για κάποια επενδυτικά μέτρα και ούτω καθεξής. Και το 2014 θα σπίσαμε ένα σχέδιο δράσης για τους νέους γεωργούς που περιλαμβάνουν κάποια φορολογικά και άλλα μέτρα προκειμένου να προσελκύσουμε τις νέες γενιές στην γεωργία με μια πιο σφαιρική προσέγγιση. Και περνάω σε κάποιες σκέψεις για τα ωφέλη αυτών των μέτρων. Ε, σε ό,τι αφορά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα είναι ε, ουσιαστική ενίσχυση για τους νέους, ουσιαστική στήριξη, γιατί είναι αρκετά υψηλά τα κονδύλια. Είναι εύκολος ο σχεδιασμός ε, και η διαχείριση των μέτρων και για το δημόσιο και για τους δικαιούχους. Επίσης έχουμε ανώτερα και κατώτερα όρια που μας επιτρέπουν να επικεντρωθούμε σε πραγματικά ενεργούς γεωργούς που παράγουν για την αγορά και είναι το μόνο μέτρο που προτείνει ε, και προώθηση του επιχειρηματικού μοντέλου, του επιχειρηματικού σχεδίου. Γίνεται, δίνεται ενίσχυση με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο. Η εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι το επίκεντρο. Αυτά ως προς τα πλονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, οι αδυναμίες. Συμφωνώ με κάποιον προλαλήσαντα που είπε ότι στο σχεδιασμό θα πρέπει να έχουμε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δεκαετίες και όχι λίγα χρόνια, γιατί ε, δεν μπορούμε να αλλάζουμε πολιτικές κάθε τρεις και λίγο. Αυτό επιβαρύνει και νέους και πιο πεπειραμένους Γιώργους, γιατί δεν μπορούν να, ε, η διαχείριση των πολιτικών δεν γίνεται σε καθημερινή μόνο βάση. Επίσης, τα μέτρα προβλέπουν κάποια βοήθεια για την εκκίνηση, αλλά πολύ ε, λίγοι είναι οι καινούργοι νέοι Γεωργοί. Οι περισσότεροι νέοι Γεωργοί κληρονομούν την οικογενειακή εκμετάλλευση και τη συνεχίζουν. Ελάχιστοι είναι οι καινούργοι που πρώτοι ασχολούνται με την γεωργία. Επίσης, θέλουν μια σταθερότητα οι νέοι για να μπορούν να διατηρήσουν και μετά την τριετία τη δραστηριότητά τους. Επίσης, χρειάζονται κονδύλια για τις επενδύσεις, για την ανταγωνιστικότητά τους και για την κερδοφορία της επιχείρησής τους. Έχουμε εντοπίσει κάποια προβλήματα λόγω των εθνικών νομοθεσιών. Για παράδειγμα, η φορολογία στη Σλοβενία είναι ένα πρόβλημα και οι διαφορέ μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα. Γιατί είναι διαφορετικό ορισμό για τον ε, νεαρό αγρότη στου δύο πυλώνε. Οπότε, ε, μια τέτοια αντίφαση ή έλλειψη συνοχή ε, δεν είναι θετική. Τώρα, ποιε είναι οι προκλήσει πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις λειτουργίες και να προσελκύσουμε περισσότερους νέους στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Θα πρέπει καταρχήν να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή μακροπρόθεσμα του επιχειρηματικού σχεδίου και να είναι εύρωστο, στιβαρό το επιχειρηματικό σχέδιο ε, με κάποια ευελιξία φυσικά που είναι απαραίτητη. Πιστεύω ότι το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο, γιατί είναι ένα ζωντανό οργανισμός και οι τιμέ των γεωργικών προϊόντων είναι αρκετά ασταθεί. Και επίσης πώς θα το συνδέσουμε με τη δημογραφική και διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Σε μερικές περιφέρειες και στη Σλοβενία, η αύξηση του μεγέθου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθιστά τα αγροκτήματα πιο παραγωγικά και αποδοτικά. Το θέμα είναι πώς στις τάσεις αυτές να συμπεριλάβουμε και νέους για να επενδύσουν και αυτοί και να ενισχύσουν τη γεωργία. Επίσης, πώς θα προσελκύσουμε και καινούριους γεωργούς και πώς θα ελέγξουμε τη νομιμότητα και την συμμόρφωση με τις διατάξεις. Ε, άλλος προβληματισμός είναι κατά πόσο χρειαζόμαστε ένα καθεστώς πρόορης ε, συνταξιοδότησης, πώς θα απλουστεύσουμε το διοικητικό άχθος, πώς ε, θα σταθεροποιήσουμε το εισόδημα, πώς θα δώσουμε κίνητρα για την οργάνωση των γεωργών, θα βελτιώσουμε την πρόσβαση στη γη και στην πρόσβαση στον δανεισμό και πώς θα προσδιορίσουμε τον ενεργό αγρότη. Σημαντική είναι η συνεργασία με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή τους νεαρούς γεωργούς. Και να σας δείξω και δύο γραφήματα. Το πρώτο δείχνει τον αριθμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και πώς ε, ε, αναπτύσσονται. Έχουμε τις, ε, ε φάρμες, τα αγροκτήματα που περιβαίνουν το κατόφλι των τεσσάρων εκταρίων. Αν, αν δείτε όμως τους νεαρούς γεωργούς, το χαμηλότερο ποσοστό είναι 80% και φτάνουμε στο 100% το 2017. Αυτός ο δείκτης δείχνει τον αριθμό των νέων γεωργών και σε σχέση με τον αριθμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που είναι σταθερές. Βλέπουμε όμως τι αλλαγές γίνονται στα μεγέθη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στις αλλαγές στον πληθυσμό διαπιστώνουμε ότι ο αριθμός των νέων γεωργών αυξάνεται. Επίση, οι γεωργικές πολιτικές και οι πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης βελτιώνουν ε, την ανανέωση των γεωργών και την αντιμετώπιση του φαινομένου της γύρασης του γεωργικού πληθυσμού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που μας κάνατε, γιατί πραγματικά ε, επισημάνατε τα ουσιαστικά προβλήματα για τους νέους γεωργούς. Ο κύριος Φλάνναγκαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε ε, στην τελευταία διαφάνεια. Βλέπουμε πλήρης αντίφαση με αυτά που είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ε, κατ' ουσίαν έχουμε ε, με συγχωρείτε, το ελεγκτικό συνέδριο. Ε, το θέμα είναι πώς μπορέσαμε να καταλήξουμε σε τόσο διαφορετικές απόψεις. Ε, εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι απόλυτα απογοητευμένος με αυτά που έχει κάνει η κυβέρνησή μου ε, με τους νέους γεωργούς ε, στις διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό Omnibus. Ίσως κάποιος από την Ιρλανδία μπορεί να μου εξηγήσει γιατί θελήσαμε να αλλάξουμε το κείμενο, να πάμε από το σαλ στο ΜΕΙ και με τον τρόπο αυτό να περιορίσουμε τα χρήματα που δίδονται στους νέους γεωργούς. Το ΣΑΛ, έχω μιλήσει με πολλούς κατά την άποψή μου, σημαίνει κατ' ουσίαν ποτέ. Έτσι ερμηνεύεται. Ο κύριος Ντεκάστρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ε, και θα ήθελα πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω για την ομιλία, να ε, χαιρετήσω και τον πρώην συνάδελφό μας ε, για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε. Εγώ θέλω να διευκρινίσω κάτι, περισσότερο οικονομικά, όχι τόσο από το πρίσμα του Ευρωβουλευτή. Εδώ και δεκαετία δεκαετίες έχει αναφερθεί ότι το θέμα της μείωσης των γεωργών είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο της αναπτυσσόμενης οικονομίας και δεν είναι παθογένεια. Δηλαδή, ε, με την ανάπτυξη της ε, οικονομίας, την ε, εκβιομηχάνηση και τη χρησιμοποίηση όλο και περισσότερων μηχανών, προφανώς και περιορίζεται το εργατικό δυναμικό ένα πέμπτο του σύτου, του παργόμενου σύτου. Παλαιότερα απαιτούσε χ αριθμορών, τώρα παράγεται σε λιγότερο από μισό λεπτό. Είναι λοιπόν σαφές ότι η ανάπτυξη της οικονομίας οδηγεί σε μείωση της απασχόλησης. Υπάρχει βέβαια και το θέμα της γύρανσης, γιατί είναι προφανές ότι οι πρώτοι που εγκαταλείπουν τη γεωργία είναι οι νέοι, αυτοί που έχουν περισσότερες δυνατότητες απασχόλησης. Είναι λοιπόν σημαντικό ε, να λαμβάνονται υπόψη αυτά τα οικονομικά στοιχεία και οι πολιτικές για τους νέους να μπαίνουν σε ένα πλαίσιο, να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική ανάπτυξη γιατί είναι δυστυχώς αναπόφευκτο να υπάρχει αυτή η διαρροή. Αντίθετα, αν δεν υπάρχει ανάπτυξη στην οικονομία, αν ε, δεν αυξάνονται τα εισοδήματα, έχουμε το αντίθετο. Δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο το οποίο κατά την άποψή σα εντάσσεται σε μια δυναμική ε, οικονομία που είναι χαρακτηριστική για μια αναπτυσσόμενη οικονομία. Ναι, δύσκολους καιρούς έχουμε μία ε, επιστροφή το, του πληθυσμού προς, τις, προς την Ήπεθρο, γιατί εκεί βρίσκουν πολύ πιο εύκολα τα προστοζήν και επιβιώνουν καλύτερα. Κύριε Μαγκίνες. Ευχαριστώ. Εγώ δεν βλέπω ποια είναι η αντίφαση. Αφενός έχουμε την πρακτική, ε, την πραγματικότητα ε, που ζει ένα Υπουργείο και από την άλλη έχουμε τον, το ελεγκτικό συνέδριο αυτό που με ανησυχεί είναι ότι ο ελεγκτής, ο κύριος Βοητσαχόφσκι, έδωσε κάποιες ε, αναφορές ε, σε ό,τι αφορά τα top-ups για τους νέους γεωργούς. Ελπίζω ότι δεν θα επηρεαστούν οι ελεγκτές από μία υπόθεση για να πούν ότι δεν λειτουργούν οι πληρωμές προς τους νέους γεωργούς. Διότι, όπως είπα και προηγουμένως, στο προηγούμενο πάνελ, δεν μπορούμε να φτάσουμε στο συμπέρασμα αυτά, διότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε με το τι θα γινόταν εάν δεν είχαμε δώσει τα κίνητρα αυτά. Το συμπέρασμά μου από την Ιρλανδική εμπειρία είναι ότι είχαμε πολύ σημαντική αύξηση νέων ε, που εκπαιδεύονται στις ε, ακαδημίες ε, τις αγροτικές πραγματικά δημιουργήθηκε ένα ενδιαφέρον για τους νέους και αυτό είναι θετικό. Τώρα δεν ξέρω εάν έχουν προτάσεις βελτίωσης ε, οι παρεμβαίνοντες. Ευχαριστώ κύριο Μπόγκοβιτς. Ε, Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους δύο καλεσμένους μας και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον συνάδελφο, τον συμπατριώτη μου από τη Σλοβενία και ευχαριστώ και τους συντονιστές ε, που δέχτηκαν την πρόταση ε, να καλέσουμε Σλοβαίνο για να μας παρουσιάσει το σύστημα για τους νέους γεωργούς στη Σλοβενία. Ήμουν για αρκετά χρόνια υπουργό Γεωργία στη Σλοβενία και μπορώ να σα πω ότι τα μέτρα για του νέου γεωργού λειτουργούν πολύ καλά στην πατρίδα μου. Χωρί τα μέτρα αυτά, αποκλειόταν να προσελκύσουμε 4-5 χιλιάδες νέους για να αναλάβουν ή να συνεχίσουν γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Σίγουρα τα χρήματα αποτελούν ένα κίνητρο για να έρθουν στη Γεωργία οι νέοι και να παραμείνουν ζωντανές οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Συμφωνώ επίσης με τον κύριο Δεκάστρο ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιο τμήμα της τάσης είναι μια φυσιολογική εξέλιξη και ποιο τμήμα της τάσης οφείλεται στη δυσκολία πρόσβασης στη γη γιατί η δύσκολη πρόσβαση στη γη περιορίζει τον αριθμό των γεωρικών εκμεταλλεύσεων και ενισχύει τη συγκέντρωσή τους. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πόσο αποτελεσματική είναι η κάψη ό,τι αφορά το μέγεθος των γεωρικών εκμεταλλεύσεων, αλλά δεν είναι το μόνο κριτήριο αυτό για να κρίνουμε την αποτελεσματικότητα της ΚΑΠ. Ε, οι νέοι γεωργοί έχουν την ευκαιρία με τη μείωση του αριθμού των ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κυρίως την απάλληψη των αναποτελεσματικών εκμεταλλεύσεων να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην ανάληψη μιας πιο κερδοφόρας εκμετάλλευσης. Χρειάζεται φυσικά ε, μια αποδοτική εκμετάλλευση που θα συντηρεί το γεωργό και σίγουρα είναι διαφορετική η κατάσταση αν ε, η γεωργική εκμετάλλευση είναι 30 ή 3.000 εκταρίων. Αλλά θα πρέπει ακόμη και οι οικογενειακέ εκμεταλλεύσει να μπορούν να συντηρούνται και να εξασφαλίσουμε μεταβίβαση στου νέου. Σήμερα οι νέοι δεν ασχολούνται μόνο με τη γεωργική παραγωγή. Ε, περιλαμβάνουν και τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας ε, στις εκμεταλλεύσεις τους είναι πιο δεκτική στη διαφοροποίηση. Και μια και θέλουμε ευφυή χωριά όπως έχουμε τις ευφυείς πόλεις, γιατί να μην εμπλέξουμε και άλλους τομείς και άλλες πολιτικές, κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, υγεία. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την παροχή αυτών των υπηρεσιών στην Ήπεθρο, ώστε οι βιωτικές συνθήκες εκεί να βελτιωθούν και να έχει νόημα η παραμονή Στι αγροτικέ ζώνες. Χωρίς σφαιρική προσέγγιση δεν πρόκειται να ευδοκιμήσουν τα μεμονωμένα μέτρα για τους νεαρούς Γιώργου. Ευχαριστώ. Στην επόμενη παρουσίαση θα επεκταθούμε σε τέτοια σημεία. Στο δεύτερο πάνελ των εμπειρογνωμόνων. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόγκοβιτς είπε μέρος των που ήθελα να πω, διότι για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα σε ό,τι αφορά τι επενδύσεις στον τομέα τη γεωργία Δεν αρκεί ε, να φέρουμε του νέου στη γεωργία για να καταπολεμήσουμε τη γύρανση. Πρέπει μετά αυτέ οι εκμεταλλευσει να είναι βιώσιμε για πολλά χρόνια. Ε, να καταπολεμήσουμε τη γύρανση αφενό, αλλά οι νέοι γεωργοί στη συνέχεια να μπορέσουν να ε, ασκήσουν τη δραστηριότητα αυτή για πολλά χρόνια. Αυτός είναι ο σκοπός μας στην Επιτροπή αυτή ε, και στην Επιτροπή Ρέτζη πρέπει να υπάρξουν συνέργειες ε, σε ό,τι αφορά χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους νέους. Μιλάμε για την ε, υγεία, μιλάμε για το διαδίκτυο. το έχετε εξετάσει αυτό τη βιωσιμότητα της επένδυσης διότι ομολογώ ότι είμαι αρκετά ανήσυχος διότι συζητάμε για εμπορικές συμφωνίες με τη Νέα Ζηλανδία, με τις χώρες του Μερκοσούρ Και όλα αυτά θα δημιουργήσουν ενδεχομένω νέα προβλήματα με αθέμητο ανταγωνισμό από τα προϊόντα που έρχονται από τις χώρες αυτές. Διότι αφενός δίνουμε κάποια χρήματα, και επενδύουμε ε, προς τους νέους γεωργούς για να έρθουν στη γεωργία, ε, τους βοηθούμε να πάρουν δάνεια ε, για να επιβιώσουν, αλλά από την άλλη πλευρά η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνάπτει εμπορικέ συμφωνίε και φτάνουν προϊόντα εδώ τα οποία δημιουργούν του ανταγωνισμό. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ισορροπημένοι στην προσέγγιση μα. Από τη θέση σε ισχύ της μεταρρύθμισης ε, του 2013 μόνο τρία χρόνια έχουν περάσει ουσιαστικά γιατί άρχισε να εφαρμόζεται το 2014 η μεταρρύθμιση του 2013 οπότε ε, μόλις μια τριετία πέρασε. Τα αποτελέσματα δεν είναι όλα ορατά. Και έγινε σωστή η κατανομή των κονδυλίων. Αυτό το διαπίστωσε και ο έλεγχος του ελεκτικού συνεδρίου. Αλλά θα πρέπει ε, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τα, μειονεκτήματα της μη υλοποίησης της ανανέωσης των ε, ε, γενεών. Γιατί θα πρέπει να δούμε τι απέδωσε καρπούς και τι όχι. Ο κύριος Άγνιο, αλλά παρακαλώ, χρόνο φίδου. Ναι, ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα προς τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνεδρίου. Ε, ας πούμε ότι έχουμε μια οικογένεια γνωρίζει ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα για τους νέους γεωργούς. Ένα από τα νέα μέλη της οικογένειας λοιπόν ε, λέμε ότι αυτό είναι ο Γιώργος. Ε, συμπλήρωσε το, την αίτηση εσύ, ε, να λάβουμε αυτά τα έξτρα χρήματα, αλλά δεν αλλάζει τίποτα στην εκμεταλλευσή μας. Συμβαίνουν αυτό. Μπορείτε να μας πείτε αν συμβαίνουν τέτοιες περιπτώσεις. Σας ευχαριστώ. Τρία λεπτά καθένας παρακαλώ για τις απαντήσεις. I Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, τα πολωνικά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ε, καταρχήν, ε, δεν υπάρχει ε, διαφορά μεταξύ των στοιχείων του Ελεκτικού Συνεδρίου και των στοιχείων της Σλοβενίας, γιατί ε, στη Σλοβενία όντως έχουμε ανανέωση των γενεών, όντως έχουμε πρόοδο και συγχαρητήρια στη Σλοβενία που τα κατάφερε. Δεν είναι αντιφατικό αυτό με τα αποτελέσματα του ελεκτικού συνεδρίου. Ο κύριο Καλινόφσκι, ε, που ήταν υπουργό Γεωργία στην Πολωνία, ξέρει ότι και στην Πολωνία είχαμε θετικά αποτελέσματα και στην Ιταλία, ε, κύριε Ντεκάστρο, έχουμε βελτίωση τη ανανέωση των γενναιών. Αλλά στην πλειοψηφία των χωρών μελών η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και δεν έχει βελτιωθεί. Ναι, όντω, είναι μια φυσιολογική εξέλιξη, κύριε Ντεκάστρο. έχετε δίκιο, αλλά ε, ο ελέκτης του ελεκτικού συνεδρίου ε, δεν έχει πολιτικό όραμα. Οι πολιτικοί θα πρέπει να δώσουν το πολιτικό όραμα και την κατεύθυνση της γεωργίας ε, από το 2040-2050. Αν, αν έχουμε ήδη χάσει τόσα εκατομμύρια εκμεταλλεύσει, τι θα γίνει σε 20 χρόνια θα έχουμε μισό εκατομμύριο ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις ε, τεράστιες ή θέλουμε να διαφυλάξουμε και την επιβίωση των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων. Γιατί όσο περισσότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις έχουμε, τόσο δύσκολο θα, θα συμβιβάσουμε τα συμφέροντα της γεωργίας ε, με τα συμφέροντα του περιβάλλοντος. Όσο περισσότερες οικογενειακές εκμεταλλεύσεις έχουμε, τόσο μικρότερες θα είναι οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Επίσης, τι θα γινόταν αν δεν είχαμε καθόλου βασικές ενισχύσεις. Θα ήταν πολύ χειρότερη η κατάσταση, γιατί οι γεωργοί εκμεταλλεύτηκαν τις άμεσες ενισχύσεις και χωρίς ενισχύσει αυτές η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη. Απλώς διαπιστώνουμε ότι ήταν ανεπαρκείς αυτές οι ενισχύσεις, γιατί ο στόχος ήταν η ανανέωση των γενναιών, η βελτίωση της ηλικιακή κατάστασης του γεωργικού πληθυσμού και τέτοια βελτίωση δεν διαπιστώσαμε συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το συμπέρασμα του Ελεκτικού Συνεδρίου. Κύριε Μπούντα, κύριε Μπογκόβιτ, χρειάζεται καλύτερο συντονισμό. και αυτό λένε και τα συμπεράσματα του Ελεκτικού Συνεδρίου και καλύτερο συντονισμό τη γεωργική πολιτική με τι υπόλοιπε πολιτικέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί μόνο οι ενισχύσει δεν αρκούν για να παραμείνουν οι οικογένειε στην Ήπεθρο. Να βελτιωθούν οι υποδομέ χρειάζεται, να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο. Αυτό είναι το ουσιαστικό έναυσμα για να παραμείνουν οι νέοι στην Ήπεθρο. Σα ευχαριστώ γιατί και οι δικέ σα παρατηρήσει συνάδουν με τα δικά μα συμπεράσματα. Κύριε Έγγινιο, Άγγινιο, πραγματικά έχουμε τέτοια παραδείγματα και στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Είχαμε ένα ε, συνεταιρισμό με μέλη και μόνο ο ένας είχε 16% ε, του, ε, της εταιρείας και χωρίς να είναι καν ενεργός γεωργός ελάμβανε ενισχύσεις. Αυτό όντω είναι μια κατάχρηση του συστήματος. Όντω θα πρέπει ο ενεργός Γιώργο είναι αυτός που απολαμβάνει τις βασικές ενισχύσει και όχι με τεχνάσματα να καρπώνονται τις ενισχύσει και άλλοι. Ο κύριος Ρόμπλεκ. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ ε, πράγματι ε, δεν υπάρχει καμία διαφορά στα στατιστικά νούμερα. Αν δούμε τους απόλυτους αριθμούς, η κατάσταση στη Σλοβενία ε, καταδεικνύει μια σχετική βελτίωση. Νομίζω ότι το ποσοστό των γεωργών κάτω από 35 ετών έχει αυξηθεί κατά τη με βάση τα τελευταία στοιχεία. Αλλά αν δούμε λιγάκι το δίκτυ που δείχνει τη μείωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την απόλυτη αύξηση του αριθμού των νέων γεωργών, τότε πράγματι διαπιστώνουμε αύξηση γενικότερη, αλλά είναι και θέμα αρμηνίας. Και θέλω να πω, συμφωνώ, στη Σλοβενία όλοι πιστεύουν ότι τα μέτρα για τους νέους γεωργούς είναι από τα καλύτερα. Αυτή είναι μια άποψη που τη συμμερίζονται και οι νέοι και οι πιο ηλικιωμένοι γεωργοί. Οι πιο ηλικιωμένοι γεωργοί ε, ξέρουν πια ότι πρέπει να παραδώσουν στους νέους και οι νέοι είναι εκείνοι που πρέπει να επιφέρουν διαρθρωτικές αλλαγές, ε, να απασχολήσουν περισσότερα άτομα. Είναι αλήθεια ότι τα επιδόματα δεν ε, αλλάζουν τη ζωή σε μια γεωργική εκμετάλλευση. Όμως σε συνδυασμό με άλλα μέτρα πρέπει να εστιάσουμε ε, στο να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, να μπορούν οι νέοι να εμπλακούν στη γεωργία και επίσης να μπορούν να επιφέρουν και διαρθρωτικές ε, εκμεταλλεύσεις, να απτύξουν και άλλες δραστηριότητες, να αγοράσουν νέα γη για διαφοροποίηση. Ε, στην Σλοβενία υπάρχει το εξής θέμα ότι περίπου το 80% των εκτάσεων βρίσκεται σε περιοχές που δεν ενδείκνυνται για γεωργική δραστηριότητα. Αν θέλουμε λοιπόν να προσφέρουμε κίνητρα στους νέους να παραμείνουν στην περιοχή ε, και να συνεργάζονται με άλλους και να πτύξουν άλλες δραστηριότητες, ποιος θα κάνει όμως τελικά την καλλιέργεια. κάνει για θα καλλιεργεί πια τη γη. Και αν υπάρξουν αλλαγές στην Ήπετρο, αυτό θα επηρεάσει και τον τουρισμό και, άλλες, και άλλα θέματα. Εμείς καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ΚΑΠ μπορεί να μην είναι και η καλύτερη, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, συμπληρώνει αποτελεσματικά και σε εθνικό επίπεδο πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και άλλα στοιχεία υγείας ε, και άλλα. Θερμότητα, ευχαριστώ. Νομίζω ότι μας δώσετε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες ε, και ο κύριος Βοητσεχόφσκι από το Ελεκτικό Συνέδριο και εκπρόσωπος ε, του Σλοβενικού Υπουργείου Γεωργίας. Και σας ευχαριστώ θερμά όλους που τηρήσατε και τους χρόνους αγόρευσης. Περνάμε στο δεύτερο πάνελ. Έχουν ήδη καθίσει στη θέση τους ε, οι Θα δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Iris Bowers, που είναι αντιπρόεδρος ε, της, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νέο, Νεαρών Γεωργών και από την ε, Ολλανδική Ένωση Νεαρών Γεωργών. Θα λάβει πρώτα το λόγο, μετά η κυρία Ταλιαλιώνη ε, από την Τζόλη, συγγνώμη, από το Ιταλικό Συμβούλιο ε, Αγροτικής Έρευνα και Ανάλυσης ε, ε, Γεωργικών Οικονομικών και μετά ο κύριο Γκυγιόμ Κρό από την Επιτροπή των Περιφερειών, την Επιτροπή Φυσικών Πόρων. Πρώτα η κυρία Ήρις Μπάουερς για 8 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Ε, συνάδελφοι νεαροί Γεωργοί, κύριε και κύριοι. Ονομάζομαι Iris Bowers και είμαι νεαρή αγρότης από, την, τις κάτω χώρες. Ε, δουλεύω με τους γονείς μου σε μια μεικτή γεωργική εκμετάλλευση με αρρώσιμες καλλιέργειες και, πάχηση και ε, χείρων. Επίσης είμαι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νεαρών ε, Γεωργών και μέλος του Συμβουλίου της Ένωσης Νέων Γεωργών στην Ολλανδία. Η ανακοίνωση για το μέλλον της ΚΑΠ έχει μεγάλη σημασία για τους νεαρούς γεωργούς στην Ευρώπη και για τη γεωργία γενικώ. Ε, γιατί χωρίς νεαρούς γεωργούς ε, δεν θα μπορούμε να παράγουμε τρόφιμα, να κρατήσουμε ζωντανή την υπεθρό και να προωθήσουμε την βιωσιμότητα και την καινοτομία. Και η υπεθρός μας θα ε, βρισκόταν σε κακή κατάσταση. Μόνο 5,6% των γεωργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 135 και μία μελέτη της Δελαβάλ και της Έτζα έδειξε άλλο ανισχυτικό αποτέλεσμα. Μόνο ένας στους πέντε ερωτηθέντες ε, έκρινε ότι έχουν κάποιο μέλλον στη γεωργία. Ε, αυτό δείχνει μια κρίση στην Ευρωπαϊκή Γεωργία και θα πρέπει να διαρωτηθούμε γιατί αυτή η κρίση είναι κανόνα σε τόσε πολλέ ευρωπαϊκέ γεωργικέ περιοχέ και είναι καθήκον μα ω εκπροσώπων πολιτικών, ε, γεωργών αλλά κυρίω ω Ευρωπαίων πολιτών να βρούμε λύσει και να βοηθήσουμε του νέου να επιστρέψουν στα χωράφια. Και εδώ είναι που έρχεται και κολλάει η ΚΑΠ. Ως ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, Νεαρών Γεωργών έχουμε πολλούς μηχανισμούς ε, για να ενισχύσουμε την ανανέωση των γενεών στην ΚΑΠ. Επίσης θέλουμε ένα πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό της ΚΑΠ. 20% να αφιερώνεται στην ανανέωση των γενεών και ξεκάθαρο ορισμό του ενεργού γεωργού, που είναι η βάση για τις ενισχύσεις. Το Συμβούλιο μας θεωρεί ότι είναι ενεργός γεωργός αυτός που αναλαμβάνει την οικονομική ευθύνη της διαχείριση μιας επιχείρηση και παραγωγής, παράγει μεμονωμένο ή μέσω ε, συνεταιρισμών, αναγνωρίζεται από το δημόσιο και προσφέρει δημόσια αγαθά από την ε, γεωργική του δραστηριότητα. Σε ό,τι αφορά τις ενισχύσει και τη διαδοχή θα πρέπει να επαναπροσανατολίσουμε τι άμεσε ενισχύσει για να εξασφαλίσουμε βιωσιμότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων και να βελτιώσουμε την ανανέωση των γενεών με βάση συνδυασμό στρεματική ενίσχυση και ενίσχυση που δράζεται στη γεωργική δραστηριότητα και να βοηθήσουμε τη συνδεδεμένη και με συνδεδεμένη υποστήριξη στου ευάλωτου τομεί. Να εξυγχρονίσουμε το σύστημα των αποσυνδεδεμένων πληρωμών και να μην έχουμε μόνο στρεματική ενίσχυση και να, λάβουμε και νομοθετικέ δράσει για να, για να θεσπίσουμε εθνικά προγράμματα, για να βελτιώσουμε την κινητικότητα των υγεών και την σωστή σωστό προγραμματισμό της διαδοχής. Επίσης, ε, θέλουμε καλύτερη μεταφορά τεχνογνωσίας ε, και παροχή συμβουλών και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των γενεών μέσω επίμορτης οργοληψίας, ε, μακροπρόθεσμης αγρομίστωσης και υπηρεσιών κινητικότητας της γης. Και εγώ αξιοποίησε τη μεταφορά τεχνογνωσία από την οικογένειά μου. Το 61 ο παππού μου ανέλαβε από το δικό του πατέρα. Είχε 5 γελάδε, 2 χείρου και 7 εκτάρια γης. Κατάφερε να καλλιεργήσει και να συντηρηθεί χάρη στις τράπεζες, στην ΚΑΠ και τη δική του επιχειρηματικότητα. Το 1997 ο πατέρας μου ανέλαβε από τον παππού μου την γεωργική εκμετάλλευση. Είχε τότε 25 γελάδες, 360 χείρους και 60 εκτάρια γης. Κατάφερε λοιπόν και αυτό να συνεχίσει τη γεωργική εκμετάλλευση και να επιβιώσει χάρη στην τράπεζα, την ΚΑΠ και την επιχειρηματικότητά του. Τώρα, το 2017, εγώ δουλεύω στη γεωργική εκμετάλλευση των γονιών μου. Έχουμε 1250 χείρους προσπάχηση και 120 εκτάρια γης. Και ελπίζω να αναλάβω εγώ την εκμετάλλευση αυτή στο μέλλον. Για να συντηρηθώ όμως θα χρειαστώ την τράπεζα, μια κατάλληλη κοινή γεωργική πολιτική και φυσικά τη δική μου επιχειρηματικότητα. Είναι προφανές ότι δεν θα μπορούσα να ασχολούμαι με τη γεωργία τώρα αν δεν είχαμε την οικογενειακή μας ε, εκμετάλλευση. Η πρόσβαση στη γη μάλιστα είναι από τα σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι γεωργοί όταν θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Γεωργών θεωρεί ότι είναι σημαντικό τα μελλοντικά μέτρα τη ε, ΚΑΠ θα πρέπει να περιέχουν και μέτρα για ε, υποχρεωτικό σύνδεσμο μεταξύ της πρόσβασης στη γη και του ορισμού του ενεργού ε, γεωργού, να έχουμε μέσα για την πλήρη μετάβαση της διαχείρισης ε, της εκμετάλλευσης ώστε να πραγματοποιεί τέτοιες αποφάσεις ο νεαρός γεωργός και επίσης να προσέξουμε ιδιαίτερα όσους δεν έχουν γεωργικό υπόβαθρο εφαρμόζοντας υποχρεωτικά προγράμματα για να βελτιώνουμε τις δυνατότητες πρόσβασης νέων, καινούριων, εισερχόμενων γεωργών. Θεωρούμε ότι η εξαίρεση από τις κρατικέ ενισχύσει για την απόκτηση γη είναι σημαντικό για την αύξηση των νέων γεωργών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, θα πρέπει να βελτιώσουμε την πρόσβασή τους στον τραπεζικό δανεισμό ε, και να προβλέψουμε και κάποιες ενισχύσει για την εκκίνηση ή συνεχίσει επενδυτικέ ε, βοήθειε καθ' όλη την δημοσιονομική περίοδο. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Περιφερειακής Αγροτικής Ανάπτυξης ε, θα πρέπει να μην είναι το μόνο μέσο στήριξη ε, της ανάπτυξης υπαίθρου. Θα πρέπει να έχουμε και εθνικά αποθεματικά που να συμβάλλουν. Ένα ε, σημαντικό θέμα της ανακοίνωσης για την ΚΑΠ, παρόλο που παρέλειψε πολλά σημεία, είναι ότι οι νέοι στην Ήπεθρο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες αντίστοιχη με αυτές που έχουν οι νέοι στις πόλεις γιατί η γεωργία δεν είναι αμυγός ε, οικονομικός κλάδος, έχει και μια κοινωνική διάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να παραμείνουν νέοι στην υπεθρό ε, και να μπορούν να συντηρούν τις οικογένειές τους. Θα πρέπει να έχουμε σωστές διασυνδέσεις με κατάλληλες συγκοινωνίες, μεταφορές, με ευρυζωνικό διαδίκτυο. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για την υπεθρό, όπως και οι παράγοντες που προανέφερα τη σήμερα ημέρα. Το να είναι κανεί νέο και γεωργό είναι σαν να ανεβαίνει ένα κακοτράχαλο ανήφορο. Μερικέ φορέ φαίνεται το πάθο είναι το μόνο που μα κρατά στην πορεία αυτή. Γι' αυτό και η ανανέωση των γενναιών θα πρέπει να αποτελέσει αγκονάρι τη μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική. Και έχουμε υψηλέ προσδοκίε και φιλοδοξίε από την ανακοίνωση. Η γεωργία έχει θεμελιώδη σημασία για την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών και για να καταφέρουν να τα βγάλουν πέρα οι νέοι και να μην εγκαταλείψουν τον κλάδο, όπως δείχνουν οι στατιστικές μέχρι τώρα, θα πρέπει να αναλάβουμε κάποιες προσπάθειες. Γιατί τώρα ήρθε η ώρα ώστε να κάνουμε πραγματικότητα το όνειρο της ανανέωσης των γενεών στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που τηρήσατε σχετικά το χρόνο σας. Θα είχα μία πρόταση τώρα. Η πολύ ενδιαφέρουσα και ωραία εμπειρία που είχατε από την οικογενειακή σας εκμετάλλευση που πολύ γλαφυρά μας την ε, περιγράψατε ε, είναι πολύ σημαντική και δείχνει πόσο ε, χρήσιμη ήταν η κοινή γεωρική πολιτική όλα αυτά τα χρόνια για την οικογένειά και για αντίστοιχα παραδείγματα μεταβίβασης. Ευχαριστώ και άλλους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νεαρών Γεωργών που είναι παρόντες ε, στην αίθουσα και σας ευχαριστώ θερμά γιατί έχουμε τακτική ε, συνεργασία και πολύ αγαστή με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νεαρών Γεωργών. Θα περάσουμε τώρα στη δεύτερη ομιλητριά μας, την κυρία Σερένα Ταραντζόλη από το Τελικό Συμβούλιο Έρευνα στην Γεωργία και Ανάλυσης Γεωργικής Οικονομίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ κυρίως ε, που με προσκαλέσατε. Ε, θέλω να πω ότι δεν θα μακρηγορήσω αλλά θα ασχοληθώ λιγάκι με το θέμα των πολιτικών που ισχύουν σήμερα για τους νέους γεωργούς στην Ευρώπη. Και θα προσπαθήσω κυρίως να φερθώ στην αποτελεσματικότητα γιατί ε, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές ε, που ελέγχονται και παρουσιάζονται και από το ελεγκτικό συνέδριο. Πολιτικές έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα και να προχωρήσει και η ανανέωση των ε, γεωργών. Είναι επίσης αλήθεια ότι η νέοι γεωργοί, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ε, από την εκπρόσωπη της ε, ΣΕΖΑ ε, και όπως αναφέρεται επίσης και σε κάποιες μελέτες που έχουν γίνει στην Ιταλία, έχει καταδειχθεί ότι οι νέοι δεν είναι ικανοποιημένοι από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, γιατί οι πολιτικές αυτές κατ' ουσίαν στιάζουν στις νέες επιχειρήσεις, ε, χωρίς όμως να ασχολούνται ποιοι είναι οι νέοι εκείνοι οι οποίοι ξεκινούν μια νέα δραστηριότητα και δεν ενδιαφέρονται και το τι θα γίνει ακριβώς στο μέλλον. Δεν παρακολουθούν τους νέους στη μελλοντική τους δραστηριότητα. Ε, ως εκ τούτου ε, δεν ασχολούνται οι πολιτικές αυτές κατά πόσον υπάρχει κεφάλαιο, κατά πόσον οι νέοι έχουν ε, γες και όλα τα απαραίτητα αγαθά για να μπορέσουν να πτύξουν μια επιτυχημένη γεωργική δραστηριότητα. Αυτό λοιπόν, όπως σας είπα και προηγουμένως, ε, ε, τίνει στο να πιστεύουμε όλοι ότι βεβαίω και υπάρχουν πολιτικές, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο οι πολιτικές αυτές είναι επιτυχημένες. Διερωτηθήκαμε λοιπόν, διερωτήθηκε κυρίως ε, το Υπουργείο Γεωργίας στην Ιταλία, αλλά και όλοι οι βασικοί οικονομικοί παράγοντες, πώς είναι οι νέοι εκείνοι οι οποίοι παραμένουν στη γεωργία, ακόμα και αν ξεκινήσουν μια γεωργική δραστηριότητα. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένοι πίνακες, ε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ε, θέλω να πω το εξής, ότι κάναμε συγκρίσεις και διαπιστώσαμε ότι εκτός γενικά από τους νέους στην Γεωργία διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία μείωση κυρίως στους ανθρώπους του νέου που ασχολούνται για 10 χρόνια με τη Γεωργία και μετά την εγκαταλείπουν. Άρα δηλαδή αν δεν υπάρχει η σωστή υποστήριξη, διαπιστώνουμε ότι είναι δύσκολο να παραμείνει κανεί στη Γεωργία. Και αυτό ισχύει κυρίω για άτομα ηλικία μέχρι 40 ετών. Η Ιταλία δημογραφικά παρουσιάζει γύρανση και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να επισημάνουμε ότι η εγκατάλειψη της ε, γεωργικής ενασχόλησης, αν δεν υπάρχει ικανοποιητικό εισόδημα, δεν βοηθάει την οικογένεια να επιβιώσει. Αυτό ισχύει κυρίως για τις αγροτικές περιοχές και για περιοχές όπου υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι. Ε, υπάρχει όμως και κάτι το θετικό που πρέπει να επισημάνουμε. Συγκρίναμε αυτά τα στοιχεία από απογραφές ε, και διαπιστώσαμε ότι ότι υπάρχει διαφοροποίηση. Διαφοροποίηση ως εκ τούτου υπάρχουν και κάποια μέτρα που βοηθούν τους γεωργούς να προσπορίζονται μεγαλύτερο εισόδημα. Βλέπουμε εδώ ότι κυρίως ε, οι επιχειρήσεις, οι εκμεταλλεύσεις μάλλον, οι οποίες ε, δραστηριοποιούνται σε πιο καινοτόμες τεχνικές, ε, με νέες μορφές τεχνολογίας, με τον τουρισμό, αυτές οι εκμεταλλεύσεις τελικά διατηρούν τους νέους τι κάναμε λοιπόν. Σε αυτή τη μελέτη την οποία σας προνέφερα και είναι μια μελέτη που δεν την κάναμε μόνο εμείς αλλά είναι μελέτη που έχουν κάνει και άλλοι. Προσπαθήσαμε να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες των νέων γεωργών και είναι απόλυτα σαφές ότι ε, πλέον ε, είναι, έχει ξεκαθαριστεί, χρειάζονται πρόσβαση σε τραπεζική πίστη ε, κυρίως και διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν και άλλες ανάγκες Από αυτή τη διαφάνεια βλέπετε ότι πολλές φορές ε, δεν είναι μόνο η αρχική ενίσχυση που δίδεται στους νέους αλλά ε, χρειάζονται οι νέοι και άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες. Ε, ε, κάναμε μία μελέτη στην οποία ανταποκρίθηκαν πάρα πολλοί νέοι και ένα από τα πράγματα που πέρα από την τραπεζική πίστη και τις εκτάσεις είπαν οι νέοι ότι χρειάζονται βοήθεια για να βρουν πρόσβαση στις αγορές. Εύκολο να πει κανείς ότι αναπτύσσει γεωργική δραστηριότητα αλλά αν δεν έρχεται από μία παραδοσική οικογένεια, καταξιωμένη οικογένεια στον κλάδο, είναι δύσκολο να βρει κανείς νέες αγορές. Κάτι άλλο που χρειάζονται είναι να ε, μπορούν να αναπτύσσουν έναν ευρύτερο διάλογο στην περιοχή τους ε, γιατί όσοι ασχολούνται με τη γεωργία δεν ασχολούνται μόνο με την παραγωγή θέλουν λοιπόν οι νέοι να έχουν μια επαφή με την τοπική κοινωνία με τις τοπικές αρχές και ενδεχομένως από κοινού ε, να μπορούν να προβάλλουν τις γεωργικές τους δραστηριότητες υπάρχουν και άλλα που χρειάζονται που ε, τουλάχιστον στην Ιταλία δυστυχώς πάρα πολλές φορές οι νέοι δεν έχουν όλες αυτές τις ευκολίες και υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο έχει σχέση με την πρόσβαση στις χαρασόμενες πολιτικές. Πάρα πολλοί γεωργοί διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δημόσιες πολιτικές. Δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Γίνεται λόγος για την απλούστευση των πολιτικών, αλλά ξέρετε αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά το έδειξαν όλοι οι γεωργοί. Όσον αφορά λοιπόν τις ε, ανάγκες τους... Ε, εδώ βλέπουμε πώς ε, η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, ε, η οποία πολιτική είναι η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε στους νέους στην Ευρώπη, πώς η πολιτική αυτή ε, προσανατολίζεται, πώς χαράσεται στρατηγικά. Υπάρχουν δύο θέματα που αφορούν κυρίως τους νέους γεωργούς είναι το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης και μετά το θέμα της απασχόλησης. Όλες οι άλλες ε, ανάγκες κατά κάποιον τρόπο καλύπτονται από τις χαρασόμενες ε, πολιτικές. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ε, να ασχοληθούμε κυρίως με την αρχική, με την έναρξη του επαγγέλματος, να υπάρχει μια ευρύτερη στρατηγική που να αφορά στις ανάγκες των νέων γεωργών. Κατά τη δική μας λοιπόν άποψη, τουλάχιστον κατά τη δική μου, αλλά ξέρετε αυτή είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται στην Ιταλία ε, πλέον και με άλλους ε, κοινωνικούς παράγοντες, διερωτώμεθα πώς πρέπει να εξελιχθεί η πολιτική που αφορά τους νέους γεωργούς. Σίγουρα να προσελκύσουμε νέους και πώς μπορεί να γίνει αυτό ε, για να προσελκύσουμε νέους στη γεωργία μπορούμε να δημιουργήσουμε μία δεξαμενή νέων γεωργών ε, οι οποίοι θα ασχολούνται με τη γεωργία οποτεδήποτε παρουσιάζεται ανάγκη. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία για να προσελκύσουμε τους νέους, είναι τα κουπόνια, είναι ε, ε, εργασιακά επιδόματα και πάρα πολλά άλλα. Ένα άλλο εργαλείο είναι το να τους υποστηρίζει κανείς και μετά την έναρξη του επαγγέλματος. Ο πρώτος πυλώνας της ΠΑΚ ε, σίγουρα αφορά όλο αυτό το θέμα και αφορά αυτή την κατεύθυνση, αλλά εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να στοχεύσουμε περισσότερο ε, να δώσουμε κίνητρα για την ε, ένταξη των νέων ε, μέσα σε ήδη υπάρχοντες συνεταιρισμούς γιατί ξέρετε θεωρώ ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον η βοήθεια που δίδεται στους γεωργούς βοηθάει στο να πιάσει καλύτερα τόπο, το πούμε με απλά λόγια. Η διαφοροποίηση σίγουρα και αυτή είναι ένα θέμα το οποίο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Σας ευχαριστώ πολύ διαφοροποίηση και καινοτομία. Ευχαριστώ παρακαλώ να περιορίσετε το χρόνο ομιλίας. Ε, είναι κρίμα να το κάνουμε αυτό βέβαια όταν έχουμε τα συμπεράσματα. Ίσως θα ήταν καλύτερα να ξεκινάμε από τα συμπεράσματα. Ε, εν πάση περιπτώσει, να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο, τον Κρός από την Επιτροπή Φυσικών Πόρων της Επιτροπής των Περιφερειών που είναι και αντιπρόεδρος του ε, Συμβουλίου, του Περιφερειακού Συμβουλίου της Οξυτανίας και είναι και εισηγητής για, το, για την έκθεση Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά ε, το 2020. Έχουμε μάλιστα συνεργαστεί. Για μένα η Επιτροπή των Περιφερειών έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει ε, στην ανάπτυξη της υπαίθρου, στη γεωργική ανάπτυξη και γενικότερα για την ορθή λειτουργία της κοινή γεωργικής πολιτικής μιας και σε αυτές τις περιφέρειες ζει η Γεωργία. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Συμμερίζομαι και εγώ την άποψη ότι όντως θα πρέπει οι εργασίες της πλήρωσης περιφερειών και αυτά που λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να ε, συντονίζονται. Η πρόσκλησή μου εδώ είναι μια ευκαιρία και ελπίζω να έχουμε και άλλες στο μέλλον ε, και για τη σύνταξη άλλωστε της γνωμοδότησης συναντήσαμε μια σειρά από ε, συναδέλφους σας ε, δεν θα μιλήσω βέβαια για την έκθεση, για το σύνολο της έκθεσης, σε περιπτώσει, διότι αυτή αφορούσε την κοινή πολιτική μετά το 2020, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα στην ε, ανανέωση των εκμεταλλεύσεων. Μιλώντας ε, γι' αυτό, βεβαίως θα μιλήσω για το σύνολο της έκθεση μιας και θα μιλήσουμε για το σύνολο της κοινωνική πολιτική διότι ε, συνδέονται. Όπως και εσείς ε, γνωρίζουμε, ελέγχθηκε σήμερα το πρωί, ότι υπάρχει ε, μια έλλειψη ελκυστικότητα ό,τι φορά το επάγγελμα αυτό της, του Γιώργου. Ε, αυτό σημαίνει σε πολλούς, πολλούς τομείς παραγωγής και αυτή τη στιγμή η ηλικιακή, ο ηλικιακός καταμερισμός είναι συντριπτικός χίλιοι γεωργοί τη μέρα ε, χάνονται στην Ευρώπη ε, είναι αρκετά τραγικό. Η Επιτροπή των Περιφερειών θεωρεί ότι αυτή η έλλειψη νέων στον τομέα της γεωργίας αποτελεί μια απειλή ε, για την διαφύλαξη της, γεω... της ε, γεωργικής δραστηριότητας στο σύνολό της, αλλά ιδιαίτερα για την οικογενειακή ευρωπαϊκή γεωργία ε, και τη ζωτικότητα των, των, ε, της υπαίθρου. Και θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να παρθούν μέτρα υποστήριξης για την είσοδο των νέων γεωργών στον κλάδο, την, την προσέλκυσή τους. Αυτό αναφέρεται και στην έκθεση. Πρέπει αυτό το θέμα να το εξετάσουμε στη ρίζα του. Βεβαίως και πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό το επάγγελμα του Γεωργού. Διαπιστώνουμε όμως ότι συχνά οι γεωργοί υποχρεώνονται να πολλούν τα προϊόντα τους ε, σε τιμές ακόμα και χαμηλότερες από το κόστος παραγωγής. Αυτό οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο μείωσης του κόστους, μείωσης της τιμής. Δεν μπορούμε να βασίσουμε ε, μια ε, γεωργική οικονομία υγιή σε, στο, πουλώντας κατά το κόστος ούτε να προσελκύσουμε, προσελκύσουμε νέους βέβαια. Όσο θα εξαρτάται το εισόδημα το γεωργικό από τις επιδοτήσεις, που μάλιστα ε, διακυβεύονται σε κάθε μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να αδειάζει την Ήπεθρο από τις ζωτικές της δυνάμεις. Το Υπηρεσία των Περιφερειών ε, λοιπόν συστήνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ρυθμίσει αυτές τις γεωργικές αγορές, να σταθεροποιήσει τις τιμές σε ικανοποιητικά επίπεδα. Είμαστε πεπισμένοι ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από την ε, θεραπεία και βεβαίως ε, κοστίζει και λιγότερο στον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Οι ΗΠΑ μας δείχνουν ότι τα ε, εργαλεία αυτά ε, ασφάλισης που σκεφτόμαστε για την Ευρώπη και κοστίζουν και θα θα είναι υποφελή κυρίω για τι ασφαλιστικέ εταιρείε και όχι για του Γιώργου. Αν δείτε τι έγινε στι ΗΠΑ, πραγματικά τελικά πλούτησαν οι Αμερικανοί ασφαλιστέ και το όφελο για του Γεωργού είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Η κοινή γεωργική πολιτική λοιπόν δεν είναι το μόνο ζήτημα εδώ. Εάν θέλουμε ε, δίκαιες και σταθερές τιμές ε, για, εκμετα... για πολλές εκμεταλλεύσεις ε, ανθρώπινες διαστάσεις θα πρέπει ε, να παρέμβουμε εκεί που καθορίζονται οι τιμές. Ε, ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ό,τι μπορεί ως πρώτος εισαγωγέας και εξαγωγέας ε, τροφίμων για να αλλάξουν οι κανόνες του διεθνούς εμπορίου στον βιολογικό τομέα για να έχουμε εμπορικές σχέσεις πιο δίκαιες και πιο αλληλέγγυες. το ζήτημα βεβαίως της γης. Εξαιρετικά σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό εμπόδιο για την εγκατάσταση. Οι άμεσε πληρωμέ ένα εκτάριο χωρί οροφή από το 1992 έχουν συνεισφέρει σημαντικά στη συγκέντρωση τη γη σε γεωργικέ εκμεταλλεύσει όλο και πιο μεγάλε, που είναι όλο και πιο δύσκολο βεβαίω από εκεί πέρα να μεταβιβαστούν. Μήπω θα ήταν απαραίτητο ε, για να ενθαρρύνουμε την εγκατάσταση νέου Γεωργού και την εκμετάλλευση να περάσουμε ε, από την υποστήριξη ένα εκτάριο στην υποστήριξη αναδραστηριότητα η γνώμη ε, τη γνωμοδότηση τη κοινή του τη των περιφερειών που στην κατεύθυνση αυτή. Επίση, οι άμεσε πληρωμέ και αυτέ έχουν αυξήσει την τιμή τη γη. Έχει γίνει πλέον αντικείμενο κερδοσκοπία ορισμένε φορέ. Πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα, ε, κινέζικα funds ε, αγόρασαν 900 εκτάρια στην περιοχή του Αλίε στη Γαλλία. Όχι βεβαίω για να κατασταθούν Κινέοι γεωργοί όπω αντιλαμβάνεστε Μήπως λοιπόν θα ήταν χρήσιμο για να διευκολύνουμε την εγκατάσταση νέων γεωργών να ρυθμίσουμε και τη γεωργική υγιή ε, στο επίπεδο κρατομελών, να, το, να μην αφήσουμε περιθώριο για κρατοσκοπία. Επίσης η Επιτροπή μας θεωρεί ότι τα κράτη-μέλη αλλά και οι περιφέρειες πρέπει να έχουν περισσότερες εξουσίες, περισσότερες αρμοδιότητες να νομοθετήσουν για γεωργικές, γεωργικές μεταλλεύσεις και να προβλέψουν κάποιους περιορισμούς, ιδιαίτερα σε αφορά ε, την... Ε, ε, καταπολέμηση της αρπαγής γης στην Ευρώπη και το φαινόμενο της συγκέντρωσης, κάτι που περιορίζει τις δυνατότητες που έχουν οι νέοι γεωργοί να δημιουργήσουν μια γεωργική εκμετάλλευση. Ζητούμε επίσης μια αξιολόγηση των άμεσων και έμεσων επιπτώσεων της γεωργικής πολιτικής ό,τι αφορά τη συγκέντρωση γης και της αρπαγής γης στην Ευρώπη. Σε κάποια κράτη-μέλη, σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση, κάθε, κάθε γενιά μάλλον ξαναγοράζει τη γεωργική εκμετάλλευση και μάλιστα με υποστήριξη δημοσίων χρημάτων. Αυτό είναι σπατάλι. Θα πρέπει να το εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να εξετάσει τι συνθήκε μεταβίβαση, διαδοχή ό,τι αφορά τι γεωργικέ εκμεταλλεύσει. Χαίρομαι που υπάρχει μια αύξηση ό,τι αφορά του οικονομικού κανόνε που αφορούν τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό με τον κανονισμό Omnibus, σε ό,τι αφορά την οροφή για την. Ε, αύξηση της, των ενισχύσεων κοινής πολιτικής πολιτικής του γεωργούς. Αυτό πάει προς την ίδια κατεύθυνση με αυτή που πιστεύουμε εμείς ότι πρέπει να ακολουθηθεί, όμως πολύ συχνά, όπως είπε και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Συνεδρίου, η υποστήριξη της της κοινής πολιτικής για τους γεωργούς δεν είναι αρκετά σαφώς ορισμένο. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η υποστήριξη να συνεισφέρει σε μια βιώσιμη αλληλέγγυα γεωργία και όχι στη συγκέντρωση των εκμεταλλεύσεων. Αυτή η η επιδότηση ή η υπερεπιδότηση δεν πρέπει να οδηγεί σε ανάπτυξη παραγωγικών μοντέλων που δεν αντιστοιχούν στις προσδοκίες των καταναλωτών και των οποίων οι αρνητικές επιπτώσεις θα επιβαρύνουν τους φορολογούμενους και τις μελλοντικέ γενιές. Πέρα από την κοινή πολιτική, όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει να συνεισφέρουν στην ανανέωση των γενναίων στον γεωργικό τομέα η μικρή ελκυστικότητα της υπαίθρου που δεν, όπου δεν υπάρχουν επαρκείς υπηρεσίες, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και υγείας είναι άλλο ένα φρένο για την εγκατάσταση των νέων Γιώργων, άλλο ένα εμπόδιο. Εμείς ζητούμε να ληφθούν υπόψη περισσότερο οι ζώνες της υπαίθρου σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές και να ενισχυθεί συνολικά η οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην γεωργική ανάπτυξη. Η Επιτροπή των Περιφερειών εμένει στην έκθεσή της ό,τι αφορά τα διακευευόμενα για την ανάπτυξη των ε, ε, εδαφών της υπαίθρου, των ζωτικών αυτών εδαφών και αυτό μπορεί να γίνει ε, μόνο αν δεν σταματήσουμε την αιμορραγία των αγιορικών εκμεταλλεύσεων. Ελπίζουμε ότι αυτά θα βοηθήσουν για τις συζητήσεις σας και τις αποφάσεις που θα πάρετε κυρίως. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εμείς σας ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και για τη συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών. Περνάμε στη συζήτηση. Ο κύριος Ανδρία, ο πρώτος που ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα ε, επισταμένος ε, τους καλεσμένους μας και συμμερίζομαι την ανάλυση του εισηγητού της Επιτροπής των Περιφερειών για τη ρύθμιση των αγορών, την πρόσβαση στη γη, τους μηχανισμούς δικαιοσύνης, ισοτιμίας και το σύστημα των άμεσων ενισχύσεων. Πολύ εχέφρονα τα επιχειρηματά σας και πιστεύω ότι θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και στη δική μας έκθεση. Η κυρία Ταραντζόλη ε, είπε ότι είναι απαραίτητε οι ενισχύσεις για την εγκατάσταση, αλλά δεν είναι επαρκής. Και αυτό μας προβληματίζει και εμάς. Εδώ και πολύ καιρό δουλεύουμε σε στεγανά, ε, συστήνοντας τα διαδοχικά γεωργικά ταμεία, αγροτικής ανάπτυξης, μεταπεριφερειακής ανάπτυξης, αλλά το θέμα είναι ε, να μην ε, ε, μένουμε σε τέτοια στεγανά, γιατί λέμε ότι το κοινωνικό ταμείο είναι για την κοινωνική πολιτική, τα δύο γεωρικά ταμεία για τη γεωρική πολιτική. Καλό είναι να ξεπεράσουμε αυτά τα στεγανά, γιατί ο κόσμος είναι συστημικός και περίπλοκος ε, και υπάρχουν αλληλεπιδράσεις. Ε, εδώ δεν είμαστε σε ένα, ένα γεωργικό συνδικάτο. Είμαστε πολίτες ερετοί που εκπροσωπούμε 500 εκατομμύρια συμπολίτε μας. Μέχρι στιγμής ε, παρόλο που διαπιστώνουμε τη σκληρή πραγματικότητα, δεν έχουμε καταφέρει να αναχαιτήσουμε τις απειλές για τους γεωργούς. Και η κυρία Μπόερς από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νεαρών Γεωργών επίσης είπε πολλά σημαντικά θέματα. Το θέμα της ανανέωσης των γενεών είναι μια προφανής ανάγκη και τόνισε και το λεκτικό συνεδρίο ότι οι σημερινές πολιτικές είναι αναποτελεσματικές ως προς το στόχο της ανανέωσης των γενεών στη Γεωργία. Επίσης, σε σχέση με το, την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, κύριε Βοητσεχόφσκι, εκεί, ε, εσείς προσπαθήσατε να κάνετε μια πιο ε, συνθετική προσπάθεια και να μας δώσετε μια, μας κάνετε μια ανακεφαλαίωση ε, με πολύ σύνεση και λογική. Εμείς όμως ως πολιτικοί θύνοντες θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο είναι αναπόδραστη η εξαφάνιση της Γεωργίας. Θα πρέπει να μας προβληματίσει αυτό και να δούμε ε, σε τι γεωργικό μοντέλο προσβλέπουμε και τι ε, ευρωπαϊκή κοινωνία επιδιώκουμε. Αυτή θα πρέπει να είναι η κεντρική συζήτηση. Δεν θέλουμε ε, τη μεγάλη γεωργία ένα ξέφραγο αμπέλι με γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και ούτω καθεξής ή ένα πιο ρομαντικό μοντέλο. Θέλουμε μια γεωργία που θα εξασφαλίζει πιστιστική ασφάλεια, ανθρώπινη υγεία, προστασία του περιβάλλοντος, ε, θα τονώνει την οικονομία των τοπικών κοινοτήτων, των ορεινών κοινοτήτων, ε, θα δημιουργεί θέσει απασχόλησης και στη συζήτηση για τη μελλοντική μεταρρυθμίση όλα αυτά τα στοιχεία του πολιτικού προβληματισμού θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Δεν είμαστε γεωργικό συνδικάτο, είμαστε πολιτικοί θυνόντες. Θα πρέπει να προβλέψουμε την κατάσταση. Τι θα γίνει σε μια πεντηκονταετία. Ε, θα πρέπει να διαφυλάξουμε το γεωργικό μας μοντέλο και να μην μιμηθούμε την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Κίνα και αλλού. Δεν πρόκειται εμείς να θρέψουμε ολόκληρο τον πλανήτη. Αλλά καλό θα ήταν να εστιαστούμε στη διαφύλαξη του δικού μας γεωργικού μοντέλου. Σας ευχαριστούμε θερμά για τα διαφωτιστικά σα σας σχόλια που θα συμπεριληφθούν υπόψη και στις εκθέσεις μας. Επειδή δεν είχατε λάβει, το... δεν λάβει μέρος στην προηγούμενη συζήτηση, σας επέτρεψα να παραβείτε λίγο το χρόνο αγόρευση. Κυρία Σλάιερ τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους καλεσμένους εμπειρογνώμονες και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Iris Bowers που μας παρουσίασε την Ολλανδική εμπειρία από τη σκοπιά μιας νεαρής αγρότησας. Προς τα πού οδεύουμε, προς μια βιομηχανική γεωργία με συγκέντρωση γεών, με επενδυτικό χαρακτήρα και με κερδοσκοπία. Αυτό έχουμε στη Γερμανία. 4-5 χιλιάδες ε, εκτάρια είναι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις ε, και μια τέτοια τάση διαπιστώνουμε και αλλού, στη Γαλλία, στην Ολλανδία. πού θα ε, ρίξουμε τα κονδύλια μας ε, σε τέτοιες υπερμεγέθεις ιωρικές εκμεταλλεύσεις ή θα στηρίξουμε τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Αν κρατήσουμε τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις στην Ήπεθρο, διαφυλάσσοντας την κοινωνική συνοχή, στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον αγροτουρισμό, την κυκλική οικονομία ή το θέμα της δέσμευσης διοξιδίου του άνθρακα. Και αυτό είναι σημαντικό. Ε, δεν θα πρέπει να απασχολεί μόνο την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Επίσης, μιλήσαμε για το Ταμείο Ζου, Γιουνκέρ ε, και την αξιοποίησή του και για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί θα μας εξασφαλίσουν μια πιο βιώσιμη γεωργία. Θα πρέπει όμως να λάβουμε σχετικές αποφάσεις. Βλέποντας την κατάσταση, διαπιστώνουμε ότι οι πολυεθνικές ε, θα συγκεντρώσουν τα χέρια τους τη γη τελικά, αν δεν ε, αντιταχθούμε σε αυτή την τάση. Συμφωνώ μαζί σας και συμφωνώ με τους συναδέλφους. Θα πρέπει να κάνουμε μια πολιτική επιλογή ε, για το πώς θα λειτουργήσουμε, ποιο τμήμα των κονδυλίων θα χρηματοδοτήσει τι πολυεθνικές και πόσα κονδύλια της ΚΑΠ θέλουμε να βάζει στα χέρια των πραγματικών γεωργών. Ευχαριστώ. πλησιάζει 12 το μεσημέρι. Παρακαλώ χρόνο φίδους στις παρεμβάσεις σας. Ο κύριος Μπούντα. Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος θέλω να σας πω ότι ανησυχώ πάρα πολύ όσον αφορά τη συγκέντρωση γης και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που το θίξατε το θέμα. Θέλω λοιπόν να μας πείτε αυτό το φαινόμενο πόσο έχει επεκταθεί στη Ρουμανία πάνω από 40% των αγροτικών εκτάσεων βρίσκεται στα χέρια άλλων ιδιοκτητών ε, που δεν είναι Ρουμάνοι δεν είναι καν από χώρε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή εμείς δίνουμε χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Σύριους, σε Λίβιους. Νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε πολύ. Χρειαζόμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθυντήριες γραμμές ε, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτή την συγκέντρωση γης. Και επίσης να γνωρίζουμε και πού κατευθυνόμεθα. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μεγάλες ε, γεωρικές εκμεταλλεύσεις αλλά και μικρές οικογενειακές. Ε, να υπάρχει όμως κάποια ισορροπία ανάμεσα στα δύο γιατί υπάρχουν περιοχές όπου δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλες εκμεταλλεύσεις και άλλες δεν μπορούμε να έχουμε μικρές. Ε, αυτή η συγκέντρωση γης είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα να το προσέξουμε γιατί αλλιώς θα είναι πάρα πολύ αργά. Με μεγάλη, μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα την εμπειρία της πρώτης ομιλήτριας από την Ολλανδία. Ε, κοιτάξτε, αυτά γίνονται αν δεν υπάρχουν ε, αδέλφια. Μπορείτε να μας απαντήσετε αν εσείς έχετε αδέλφια που να θέλουν ίσως και αυτά να συμμετέχουν. Γιατί αυτό κάνει τη διαφορά. Και αν πρόκειται για ένα μοναχό ε, τα πράγματα πάνε μια χαρά αυτά που είπατε για τους χείρους ε, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι της εκμετάλλευσής σας. Η ΚΑΠ δεν έχει σχέση με επιδοτήσεις για χείρους. Εσείς ε, από ό,τι άκουσα θέλετε να επεκτείνετε την επιχείρησή σας ανεξάρτητα από την ΚΑΠ. Μπράβο σας και κάτι άλλο. Εάν περιοριστούν οι ενισχύσεις και είσαστε λίγο πιο κάτω από ό,τι προβλέπετε, ε, αυτό θα αποτελέσει αντικίνητρο για σας, για να επεκταθείτε. Και αν αυτό γίνεται για νέους, ε, για να αρχίσουν να ασχολούνται με την γεωργία, αυτό πιστεύετε ότι επηρεάζει. Επίσης, ε, κάποιος είπε προηγουμένως ότι η γεωργία είναι επάγγελμα. Δεν είναι επάγγελμα, είναι ένας κλάδος. Και μένα αυτό που με ανησυχεί είναι το να μιλάμε εδώ για τους γεργούς ε, σαν να είναι υπάλληλοι που δουλεύουν για την κυβέρνηση. Ο ΠΟΕ ε, δεν θα το δεχτεί αυτό ο πρόεδρος περιμένει να χτυπήσει το ε, σφυρί του και έτσι όπως είναι και εύσομος δεν θέλω να τον προκαλέσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε πάρα πολλά για τη γύρανση στη γεωργία. Ακούσαμε για το ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στη γη, στη χρηματοδότηση, ε, σε καλές αγορές, ε, ότι υπάρχουν ε, περιοχές που αποδυναμώνονται, που οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τη γη. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής ή αναπτυσσόμετα ή καταραίουμε. Τώρα λοιπόν έχουμε τους νέους ε, που θέλουν να αρχίσουν να ασχολούνται με τη γεωργία και καλούνται να πληρώσουν το τίμημα. Ο κύριος Αντρουέ έκανε ακριβώς το σωστό ερώτημα. Για το μέλλον ποιο γεωργικό μοντέλο επιθυμούμε, αυτό πρέπει να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε. Και όταν θα αποφασίσουμε να κατευθύνουμε εκεί τα κονδύλια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ε, οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και τελικά να υποφελούνται οι μεγάλοι όμιλοι επιχειρήσεων. Αυτό αυτό όμω συνέβη ε, στο παρελθόν και αυτή είναι η κατάσταση. Οι νέοι έχουν δικέ του ιδέε, γνωρίζουν πολύ καλά ποιε είναι οι προκλήσει, είτε είναι το περιβάλλον, ε, οι όλε δημόσιε συζητήσει. Υπάρχουν και οι στόχοι τη αηφορία ε, που θέλουμε να επιτύχουμε. Για να τα κάνουμε όμω όλα αυτά είναι απαραίτητο να υπάρχει διαφοροποίηση στι γεωργικέ εκμεταλλεύσει, στη φύση, στην παραγωγή και προς τα εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε τις απαιτήσεις μας. Η αηφορία είναι η λέξη κλειδί του μέλλοντος και όχι η εντατικοποίηση. Χαίρομαι που πολλοί νέοι θέλουν να ασχοληθούν με την γεωργία. Εμείς τώρα καλούμεθα να δημιουργήσουμε ένα σωστό και δίκαιο πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ καλή η παρουσία της κυρίας Μπάουερ. Η κυρία Μπάουερ ζήτησε έναν σαφή ορισμό για τον ενεργό γεωργό και είστε από τους λίγους που το λέτε αυτό. Ε, το, η Κομισιόν και το Συμβούλιο θέλουν να καταργήσουν αυτόν τον ορισμό. Λένε ότι αυτό απλοποιεί τα πράγματα από δική πλευρά διότι κοστίζει πολύ να αναπαληθεύσει κανείς ε, ε, ποιος είναι ο ενεργός γεωργός. Πώς λοιπόν θα μπορούσαμε να έχουμε έναν ορισμό ε, σαφή και ταυτόχρονα όμως ε, να υπάρξει απλοποίηση σε διοικητικό επίπεδο. Δεν μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή σένος ή θα τι αντιμετωπίσουμε αυτόν τον νόρο; Κυριακόταουλα τρένος Ένωση για να διαφυλάξουμε, διαφυλάξουμε αυτόν τον όρο. Ευχαριστώ. Η βάση για το μέλλον της ε, ε γεωργίας ε, είναι οι νέοι. Θα πρέπει να αποφασίσουμε λοιπόν πόσο μεγάλο θα είναι το μέγεθος μιας εκμετάλλευσης. Δεν είναι το ίδιο για όλες τις χώρες. Αυτό είναι το καθήκον μας. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο πρόσωπο τη Επιτροπή των Περιφερειών. Να συμφωνήσουμε πόσοι εργάζονται σε μια εκμεταλλευσή. Επίση θα πρέπει να συνδυάσουμε διάφορες πολιτικές. Εντό τη Ένωσης έχουμε περιφερειακή πολιτική, ψηφιακή πολιτική, γεωργική πολιτική, πρέπει να συνδυάσουμε αυτά. Και σε εθνικό επίπεδο έχουμε την πολιτική υγεία, κοινωνικέ πολιτικέ, ψηφιοποίηση, ε, απασχόληση, τα κράτη-μέλη είναι πάντα υποπίεση να μειώσουν τις δαπάνες ε, τις κρατικές. Θα πρέπει λοιπόν να συντονίσουμε τις πολιτικές μας σε διάφορους τομείς και να ενθαρρύνουμε την ε, γεωργική ανάπτυξη. Θα είναι η γεωργία πάντα μια σημαντική δραστηριότητα αλλά πρέπει να αξιολογήσουμε τις πολιτικές μας και σε οριζόντιο και σε κάθε το επίπεδο να τις βελτιώσουμε και τις συναρμονίσουμε. Σύμφωνοι. Αλλά η αγορά και ο εξωτερικός ε, ανταγωνισμός ε, επηρεάζουν την κατάστασή μας, πώς θα κρατήσουμε αυτόν τον ε, εγχώριο χαρακτήρα της γεωργίας επηρεαζόμαστε από εξωτερικούς παράγοντες. Καλά, την επόμενη φορά, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Μαγκίνες, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Προ την Αρία Γρότησα, θα ήθελα να πω, είναι ενδιαφέρον ότι ο παππούς σας ε, μπορούσε να συντηρηθεί με 7 ε, εκτάρια και εσείς έχετε 120 σήμερα. Δεν ξέρω τι είναι πιο βιώσιμο, αν πρέπει να επεκταθείτε περαιτέρω για να επιβιώσετε. Υπάρχει πάντως μια φυσική εξέλιξη προς μια συγκέντρωση των, της γης λόγω της πίεσης του γεωργικού εισοδήματος. Επίσης, θα πρέπει να γίνει συζήτηση για τον ενεργό γεωργό. Όταν συζητούσαμε τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, ήμασταν όλοι της γνώμης ότι τα κονδύλια θα πρέπει να δοθούν στον ενεργό γεωργό, αλλά λιώθηκε αυτή η πρόταση στην στον κανονισμό Omnibus. Επίσης, ε, για τα σχόλια για το τι ε, γεωργία επιθυμούμε ε, θέλουμε ανώτατο όριο σε χαμηλότερο επίπεδο. Αυτό θα συζητηθεί στην επόμενη μεταρρύθμιση, ώστε να μην πηγαίνουν τα χρήματα στις μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις βιομηχανικής κλίμακας, όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι. Επίσης υπάρχουν κάποιοι τομείς που δεν καλύπτονται από την ΚΑΠ και είναι μεγάλης κλίμακας στην ακτινοτροφία, όπως τα πουλερικά και οι χείροι. Οπότε θα πρέπει να κρατήσουμε ένα ευρύ φάσμα γεωρικών εκμεταλλεύσεων, αλλά δεν ξέρω αν το μοντέλο αυτό είναι βιώσιμο για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλάναγκαν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσες οι ομιλίες. Έχω επανειλημμένως παρατηρήσει στην Επιτροπή μας ότι ακούμε τη φράση ότι είμαστε υπέρ της οικογενειακής εκμετάλλευσης και κάποιος είπε ότι όλοι είμαστε υπέρ των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, είπε ο κ. Μπόκοβιτς ή ο κ. Βανκαντελάρε. Ε, ναι, εδώ όμως ζούμε σε, κάπως απομονωμένοι στο χρυσό μας πύργο ε, και η πραγματικότητα δεν μας δικαιώνει, είναι αντιφατική. Και στην πατρίδα μου ε, οι μεγαλοκτηματίες είναι αυτοί που καρπώνονται τα κονδύλια και δεν πηγαίνουν στους ε, μικρούς καλλιεργητές. Μπορεί να είμαστε όλοι αναφαδόν υπέρ των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Παρακαλώ οι καλεσμένοι μας. Έχουν δύο λεπτά καθένας για να απαντήσουν. Η κυρία Μπάουερ, σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τι ερωτήσει και τα σχόλιά σα. Έχω έτσι την ευκαιρία να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μου για την ευκαιρία που μου δίνεται να συνομιλήσω με τόσου ευρωβουλευτέ και με εκπροσώπου τη Γενική Διεύθυνση Γεωργία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήταν πολύ δεκτική και διαλλακτική στη συζήτηση. Με ρωτήσατε αν είμαι μοναχοπέδη, αν έχω και άλλα αδέρφια. Όχι. Ούτε εγώ είμαι μοναχοπέδη, ούτε ο πατέρας μου ήταν. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό της οικογενειακής εκμετάλλευσης ε, που πραγματικά όταν δουλεύει κανείς ε, σκληρά επιβραβεύεται και έχει συζητήσεις ε, με το, τα αδέρφια. Δεν είναι εύκολο να είναι κανείς μοναχοπέδι και θα ήταν δύσκολο να αναλάβω μόνο μου την επιχείρηση. Και φυσικά και το οικονομικό εδώ κριτήριο συνυπολογίζεται. Αναφέρθηκε χειροτροφία. το επισήμαναν πολλοί ευρωβουλευτές. Εγώ είμαι περήφανη που εργάζομαι σε μια μεικτή εκμετάλλευση, γιατί έτσι είναι πιο βιώσιμη η εκμετάλλευση, ε, γιατί έχει πιο κυκλικό χαρακτήρα η δραστηριότητα. Έχουμε αφενός αρρώσιμες καλλιέργειες, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ενισχύσεις της ΚΑΠ, ενώ με τη χειροτροφία δεν έχουμε τέτοιες ενισχύσεις. Για μένα το σύστημα είναι βιώσιμο. Δεν θεωρώ βέβαια ότι ο κάθε νέος γεωργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να ε, έχει μεικτή εκμετάλλευση, αλλά για μένα είναι βιώσιμη αυτή η εκμετάλλευση και θα τη συνεχίσω. Τώρα, όταν θα αναλάβω την επιχείρηση, θα είμαι μία από τους νέους αγρότες που θα χρειαστούν και επενδυτική υποστήριξη όταν περάσει σε μένα η οικογενειακή εκμετάλλευση. Θα χρειαστώ και βοήθεια στην διαχείριση κινδύνου και κάποιες πληροφορίες ενημέρωση για την αγορά. Γιατί είναι δύσκολο να είναι κανεί επιχειρηματία σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι κλιματικέ αλλαγέ, τι εκκλήσει για ηφορία. Και εμεί θα βγούμε και στου αγρού. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη ό,τι αφορά τα ανώτατα όρια του προπολογισμού τις οροφές του προϋπολογισμού. Θεωρώ ότι αν γίνει μια πιο αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων μπορεί να έχουμε οροφές και φαντάζομαι θα συμφωνείτε μαζί μου. Επίσης, ο ορισμός του ενεργού ε, αγρότη έχει κύρια σημασία. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε καλύτερη στοχοθέτηση των άμεσων ενισχύσεων. Για να πάντα κονδύλια στους χρήζοντες βοήθειας, στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, γιατί αυτό θέλουμε. Μια διαφοροποιημένη ποικιλόμορφη γεωργία, μια αποτελεσματική κοινή γεωργική πολιτική και θεωρώ ότι όταν έχουμε στόχο την απλούστευση της ΚΑΠ και με την ψηφιοποίηση μπορούμε να το επιτύχουμε μεταξύ άλλων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά δημιουργήσετε πολλές συμπάθειες στην αίθουσα. Κυρία Ταραντζόλη. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ ενδιαφέροντα σχόλια. Είναι ότι μιλάμε για συστημική παρέμβαση και μερικές φορές ε, δεν καλούμεθα να επανακαλύψουμε τον τροχό. Υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία και σε νοσιακό και σε εθνικό επίπεδο. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι τα εργαλεία αυτά να τα χρησιμοποιούμε με πιο αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο τρόπο. Ε, Πράγματι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες ε, στο να καταρτήσει κανείς ε, μια ολοκληρωμένη γεωργική πολιτική. Υπάρχουν ε, κανονιστικές δυσκολίες αυτή τη στιγμή στα κρατημέλη. Άρα δηλαδή εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να απλουστευτούν τα εργαλεία και σιγά σιγά να υιοθετηθούν στα διάφορα κράτη-μέλη. Γιατί εκείνο που υπάρχει είναι πράγματι, υπάρχει ένα πρόβλημα συγκέντρωσης γεών. Από την άλλη, ε, στο νότο της Ευρώπης ε, διαπιστώνουμε το, ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, συνεχιζόμενη κατάτμιση και κατακαιρματισμός των γιών. Άρα δηλαδή και εκεί, στο Νότο, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις που να είναι πιο ανταγωνιστικές στην αγορά. Με λίγα λόγια, εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να χαράσονται οι σωστές πολιτικές και μετά τα μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, επίπεδο κράτους μέλους ή ακόμα και επίπεδο περιφέρειας. Και κάτι άλλο που θέλω να υπογραμμίσω έχει σχέση με το ε, ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο. Ε, είναι ρεαλιστικό πράγματι το ότι σήμερα δεν μπορούμε να παρετηθούμε από το ισχύον ε, μοντέλο γιατί η μόνη προστιθέμενη αξία που βλέπουμε στις αγορές είναι ακριβώς από τη Γεωργία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα το λόγο έχει εκπρόσωπος της Επιτροπής Περιφερειών. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτήν την ε, ε, συναρπαστική συζήτηση. Άκουσα πολλά και διάφορα, θα επιμείνω σε δύο-τρία σημεία. Ε, πρώτα απ' όλα ελέγχθη βέβαια, αλλά για την εγκατάσταση. Η εγκατάσταση δεν είναι μόνο, δεν έχει να κάνει με την ελκυστικότητα του, του επαγγέλματος του Γιώργου, Έχει να κάνει και με πολλά άλλα πράγματα και με τη δυναμική ε, της ζωής στην Ήπεθρο. Θα πρέπει να υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες, ε, δημόσιε δημόσιες υπηρεσίες ε, εγκαταλείπουν όλο και περισσότερο την Ήπεθρο, και αυτό βεβαίως ε, οδηγεί και σε μια αίσθηση εγκατάλειψης ε, και αυτό βέβαια μετά δημιουργεί και άλλα συναισθήματα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πραγματικό ζήτημα. Όταν μιλάμε για την κοινή γεωργική πολιτική δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για το επάγγελμα του γεωργού. Ε, κάτι που ενδεχομένω να μην ανέφερα σαφώ είναι ότι στην Επιτροπή περιφερειών ζητούμε να υπάρξει μια ατζέντα για την Ήπεθρο. Όπως υπάρχει η ατζέντα για τις πόλεις, να υπάρχει μια ατζέντα για την Ήπεθρο. Νομίζω το ζητάει και η Επιτροπή Γεωργίας αυτό. Είναι ίσως η πιο ευρωπαϊκή πολιτική στην οποία φερειώνουμε ένα σημαντικό μέρος του προπολογισμού. Να πάμε λοιπόν προς μια ατζέντα για την Ήπεθρο στην ανακοίνωση της Κομισιόν βέβαια δεν αναφέρεται αυτό, στην ανακοίνωση της 29ης. Ε, θα πρέπει όμως εμείς να επιμείνουμε, ελπίζω να το κάνει και το Κοινοβούλιο για να υπάρξει μία ατζέντα για την Ήπεθρο. Τώρα για την ε, συγκέντρωση, βεβαίως ε, είναι θέμα ε, επιλογής, το είπαν σχεδόν όλοι αυτό. Τι γεωργικό μοντέλο θέλουμε, ποιο θέλουμε να διαφυλάξουμε το μοντέλο του διατροφικό. Ε, εγώ θα ήθελα να λέγεται κοινή γεωργική διατροφική πολιτική. Στην ανακοίνωση της Κομισιόν γίνεται βεβαίως αναφορά σε αυτό, στην διατροφή και αυτό είναι ενδιαφέρον και υπάρχει και το μεγάλο ζήτημα ε, του διεθνού εμπορίου και τη ρύθμιση και τη απορρίθμιση. Εάν δεν μπορούμε και να τροποποιήσουμε κάποια πράγματα, ό,τι και να κάνουμε, θα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου εκμεταλλεύσει θα γίνονται όλο και πιο μεγάλε, όπου θα πρέπει να πέσουν οι τιμές κτλ. Και τελειώνοντας, ε, ε το τι θα συμβεί με την κοινωνική πολιτική θα δείξει και τι, πόσο φιλόδοξοι είμαστε για την Ευρώπη γενικότερα. Θα πρέπει, πιστεύω, να πάμε προς μια κοινωνική πολιτική που να είναι αλληλέγγυα, που να επιτρέπει στους γεωργούς ε, να μπορέσουν να επιβιώσουν και τα προσελκύσει και τους νέους. Και χαίρομαι που αυτό μας το επισημαίνει εκπρόσωπος ε, της ε, Επιτροπής Περιφερειών για τις ε, τοπικούς παράγοντες. Τώρα εκπρόσωπος ε, της ε, Σλοβενίας. Για ένα λεπτό όμως μόνο. Ευχαριστώ. Και εγώ μίλησα για τον ορισμό του ενεργού αγρότη στη δική μου ομιλία. Και πιστεύω προσωπικά ότι αν ορίσουμε τι εστί ενεργός γεωργός, ε, θα έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Ο τελικός δικαιούχος των ενισχύσεων είναι ο πραγματικός γεωργός, αυτός δηλαδή που παράγει τα τρόφιμα και τα διαθέτει στην αγορά. Είναι σημαντικό να έχουμε σωστούς ορισμούς. Ευχαριστώ. Τώρα, το λόγο έχει ο Διευθυντής, ο κύριος Χανιώτης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Χανιώτη. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε. Θα ήθελα εν συντομία να παρουσιάσω την ε, άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να επαναλάβω κάτι που έχει δηλώσει πολλά και ο Επιτροπός μας. Είναι σημαντικό και δίνουμε μεγάλη σημασία η ανανέωση των γενεών στη Γεωργία. Και ανανέωση των γενεών δεν σημαίνει περισσότεροι νεαροί αγρότες στη Γεωργία, αλλά σημαίνει ανανέωση του φυσικού κεφαλαίου, των δεξιοτήτων και της γνώσης στον κλάδο της Γεωργίας και υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ τι μπορεί να κάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο και οι γεωργοί στο δικό του επίπεδο τη αγροτική εκμετάλλευση. Και αυτό θα βρεθεί στον πυρήνα τη συζήτηση για το μέλλον τη ΚΑΠ. Μια ναι, και έχω λίγο χρόνο, δεν πρόκειται να καλύψω όλα τα ζητήματα, αλλά θα επικεντρωθώ σε ορισμένα από αυτά. Ξεκινώ από την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που μα έκανε η νεαρή αγρότησα. Γιατί Υπάρχει κάτι που εμέσως προέκυψε από την ομιλία της, αλλά δεν το δια, διασαφηνίσαμε. Από όλες τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της Γεωργίας, ε, ο αριθμός των ε, γεωργών μειώθηκε, ο το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αυξήθηκε, αλλά μειώθηκε και ο αριθμός των γεωργικών εκτάσεων. Ελαφρώς μεν, αλλά υπάρχει μια τέτοια μείωση και των γεωργικών επιφανειών. Οπότε έχουμε όλες αυτές τις στάσεις και τις πιέσεις ταυτόχρονα. Προσπαθούμε να μπούμε στο μυαλό των ε, νεαρών γεωργών, αλλά βλέποντα από έξω, θεωρώ ότι η επιλογή της παραμονής ή όχι στη γεωργική εκμετάλλευση ξεκινά από, την, ε, από το υπόβαθρο του καθενό. το γεωργικό του υπόβαθρο, την ιδιοκτησία τη γης, τι δεξιότητε, την παιδεία που έχει ο κάθε γεωργό και ειδού το λαμπρό παράδειγμα που έχουμε με την ε, νεαρή αγρότησα από την Ολλανδία. Αλλά θα πρέπει να ξεχνάμε και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές, όχι του κλάδου ολόκληρου, αλλά κυρίως της οικονομίας, της γενικότερης οικονομίας, μετά του κλάδου και, με, και της περιφέρειας. Και έχουμε και κάποιες βραχυπρόθεσμες ε, ε, παρατηρήσεις. Ε, ποιο είναι το κόστος της γης και το κόστος του εργατικού δυναμικού, της εργασίας. Ε, υπάρχουν κάποια ζητήματα που εξαρτώνται από τις πολιτικές και άλλα που είναι ανεξάρτητα. Έχουμε τις άμεσες ενισχύσει που είναι ένα δίκτυο ασφαλείας για το γεωργικό εισόδημα και όσο περισσότερο συνδέονται με κάποια αντικειμενικά κριτήρια, είναι, είτε αναφορά το κόστο τη γη είτε το εργατικό δυναμικό αυτό, δημιουργεί τεράστιε διαφορέ ε, και μεταξύ των χωρών μάλλον και εντό της ε, κάθε χώρα μεταξύ των περιφερειών. Και αυτό αντικατοπτρίζει το τι επιδιώκουμε να στηρίξουμε. Και το καθεστώς για τους νέους γεωργούς είναι ένα μικρό τμήμα του όλου συστήματος και δεν θα πρέπει να ε, ε, κριθεί μόνο με βάση το πιθανό θαυμάτο που θα μπορέσει να προκαλέσει. Είναι μόνο ένα συμπλήρωμα και μιλούμε για έναν πάγιο και περιορισμένο προπολογισμό. Και να δούμε τι δεν εμπίπτει στην ΚΑΠ ε, ή σε μια ευρωπαϊκή πολιτική. Καταρχήν η φορολογία. Η φορολογία δεν είναι κοινοτική αρμοδιότητα. Σε μεγάλο βαθμό όμω η φορολογία ξε... Ε, καθορίζει τις ευκαιρίες ε, για την είσοδο ή την έξοδο από το ε, ε, επάγγελμα. Επίσης, κληρονομική διαδοχή. Και γι' αυτό ισχύουν διαφορετικοί κανόνες στα κράτη-μέλη για τη διαδοχή και τη μεταβίβαση. Επίσης, ε, το 50% των γεωργικών εκτάσεων ε, δίνονται με αγρομίσθωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό είναι ο μέσος όρος. Ε, η ψελίδα είναι από 15% μέχρι 80% και ανάλογα με το ποσοστό αγρομίσθωσης η κατάσταση είναι διαφορετική. Και το θέμα των ευρύτερων υποδομών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Οπότε πολλά επηρεάζουν την κατάσταση. Επίσης θα πρέπει να τραβήξουμε μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ ενός προβλήματος που καλούμαστε να λύσουμε και κάποιων καταστάσεων που παρατηρούμε παντού στον κόσμο, άσχετα από το αν εφαρμόζουν μια κοινή αγροτική πολιτική ή όχι. Αυτό κάναμε πριν από μία διετία, στα πλαίσια της Expo του Μιλάνου. Είχαμε ένα σεμινάριο για νεαρούς γεωργούς. Καλέσαμε περίπου 100 και μάλιστα οι δικές τους οργανώσεις τους επέλεξαν και τους φέραμε σε 10 διαφορετικές τρογγυλές τράπεζες ε, και μετά από συζητήσεις μεταξύ τους τους ζητήσαμε να καταλήξουν στις ε, τρεις κατά τη γνώμη του πρωταρχικέ προτεραιότητες για τα προβλήματα που χρήζουν επίλυση Σε μία από τι 10 στρογγυλέ τράπεζε. και μόνο τρίτη προτεραιότητα ήταν η αστάθεια των τιμών. Και τα δύο πρώτα θέματα ήταν η πρόσβαση στη γη και η πρόσβαση στο δανεισμό. Αυτά ήταν τα πρωτεύοντα ζητήματα που προέκυψαν από τι δέκα στρογγυλέ τράπεζε. Και με εξέπληξε η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου που έκανε κάποιες διαπιστώσεις ε, για τις πολιτικές. Όπου και αν βλέπουμε στον κόσμο, βλέπουμε, παρατηρούμε ε, μείωση του αριθμού των γεωργών. Το είπε και ο κύριος Δεκάστρο. Μείωση του αριθμού των γεωργών ε, υπάρχει παντού στον κόσμο. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το θέμα είναι η πολιτική επιβραδύνει ή επιταχύνει αυτή τη διαδικασία. Και μάλιστα θα δείτε σε δύο εβδομάδες ότι η ΚΑΠ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιβράδυση αυτής της ε, τάσης και στη μείωση της φτώχειας στην Ήπεθρο. Επίσης, οι ε, θέσεις που χάνουμε στον πρωτογενή τομέα αντικαθίστανται από καλύτερε θέσεις απασχόλησης, περισσότερες δεξιότητες και υψηλότερους μισθούς στην Ήπεθρο σε άλλους τομείς της οικονομίας. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα της ανάπτυξης. Πράγματι έχουμε το πρόβλημα της γέρανσης του πληθυσμού σε ολόκληρο τον αναπτυσσόμενο κόσμο, το πρόβλημα της πυραμίδας κυρίως ε, στις ηλικίε, άρα δηλαδή είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και υπάρχουν και μακροχρόνιες τάσεις που και αυτές επηρεάζουν, όμως δεν έχουμε δει ή δεν εξετάσαμε την άμεση σχέση που υπάρχει με την οικονομία και το περιβάλλον. Και μάλιστα συγκεκριμένα στο πλαίσιο της, εξ, της έκθεσης του Μιλάνου είχαμε ένα εργαστήριο που έδειξε ότι μπορούμε να έχουμε μικρές εκμεταλλεύσεις που να είναι εξίσου αποτελεσματικές και αποδοτικές όπως και μεγάλες. Στις βιολογικές καλλιέργειες οι πιο αποτελεσματικές είναι αυτές που είναι μεγάλης έκτασης και όχι μικρές. Και τα λέω όλα αυτά γιατί έγινε λόγος για τα εργαλεία, ε, το, τι μπορεί και να πετύχει με τα εργαλεία. Δεν ζούμε πια στη δεκαετία του 50 όπου είχαμε την ιδέα ότι για κάθε στόχο υπάρχει ένα συγκεκριμένο εργαλείο. Τώρα πια ζούμε σε ένα πολυεπίπεδο, πολύπλοκο κόσμο Τώρα πια λοιπόν πρέπει να εντοπίσουμε πρώτα απ' όλα ποιος είναι ο πρωταρχικός στόχος και κατά δεύτερον να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια βεντάλια εργαλείων ε, τα οποία θα χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο που θα είναι συμπληρωματικά για την επίτευξη του στόχου. Θέλουμε περισσότερους νέους γεωργούς ε, που να ασχοληθούν με τη γεωργία και αν το θέλουμε πραγματικά αυτό ε, πρέπει να γνωρίζουμε απολύτως ε, πώς μπορεί να γίνει χωρίς να απασχολούνται περισσότερο, περισσότεροι γεωργοί στον ενεργό πρωτογενή τομέα. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό στο μέλλον, πώς μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός, ε, να είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχουμε σήμερα. Ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε, να πούμε ότι σε όλες τις περιφέρειες ε, πρέπει να έχουμε γεωργικές ε, περιοχές οι οποίες θα προσφέρουν απασχόληση, θα έχουν σχέση με την αλυσίδα διατροφής και εκεί θα απαιτούνται ε, περισσότερες δεξιότητες. Οφείλουμε να εστιάσουμε και στο θέμα της αηφορίας. Είτε έχει σχέση με το κλίμα, είτε με το περιβάλλον, είτε και με την κοινωνική αηφορία των γεωργικών, των αγροτικών περιοχών. Για να τα πετύχουμε όλα αυτά πρέπει να ε, συνδυάσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη, στα χέρια μας. Τέλος, για τις τιμές των γεωργικών προϊόντων. Υπάρχει μια ανακοίνωση ως προς ότι μπορεί και τι δεν πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη. Να είμαστε σαφείς περί τίνος πρόκειται. Ε, στο πλαίσιο ε, της διεύνησης, ε, όταν είχαμε αυτά τα νέα κρατημέλη, γνωρίσαμε πολύ καλά ότι τα περισσότερα εξ αυτών έρχονται χωρίς κανένα επίπεδο ενισχύσεων. Ε, ή άμεσες εγχύσεις ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο υποστήριξης, γνωρίζαμε ότι αυτό θα επηρέαζε τις τιμές των γεωργικών προϊόντων. Το περιμέναμε. Όμως, ε, σε επίπεδο γεγονότων, δεν βλέπουμε αυτή την άμεση διασύνδεση που κάνουν πολλοί, δηλαδή ανάμεσα στην ύπαρξη εισοδηματικής υποστήριξης ε, ε, σε, όλα τα κρατημέλη και στην κεφαλαιοποίηση της γης. Και δεν το βλέπουμε για τον εξής λόγο. Πρώτον, υπάρχει μια περίπτωση ενός ε, κράτους μέλους το οποίο ε, ισοπαίδωσε όλες ε, τις ενισχύσεις και εκεί υπήρξαν ε, περιφερειακές αλλαγές. Σε όλες τις άλλες χώρες, Ολλανδία παραδείγματος χάνει, η πίεση στις γεωργικές τιμές δεν προέρχεται από το επίπεδο επιδομάτων, αλλά από τις πιέσεις που υπάρχουν γενικότερα. Τι εννοώ? Εννοώ ότι δεν πρέπει να υιοθετούμε το αποτέλεσμα της ανάλυσης, αλλά θα πρέπει να εστιάζουμε στα πραγματικά πραγματικά γεγονότα, τα οποία μάλιστα είναι ακόμα πιο περίπλοκα από τον τρόπο που σας τα παρουσίασα. Σας ευχαριστώ πολύ που με αφήσατε να μιλήσω. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο κύριος Χανιώτης μας έκανε μια πολύ εύστοχη ανακεφαλαίωση της όλης συζήτησης και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ε, τρία σημεία. Οι σημερινές ε, ομιλίες ε, δίνουν πολύτιμες πληροφορίες ε, στον ε, κύριο Καπούτο, τον εισηγητή μας. Ε, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας παρουσίασε και κάποιες σκέψεις και σας καλώ και εσείς να διαβάσετε στον Επίτροπο Χόγκαν τα, τις γραμμέ γραμμές της σημερινής συζήτησης, γιατί ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται, περί του μέλλοντος της κοινή γεωρικής πολιτικής. Και έτσι τροφοδοτείται η όλη συζήτηση. Ε, όπως μας είπε ο πρώην Ευρωβουλευτής ε, και με, νυν μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου, ο κ. Βοητσεχόφσκι, ε, θέλουμε οι διατάξεις να φέρουν τους νέους γεωργούς ε, σε μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. Όχι για 5-10 χρόνια, όχι για το 2030, αλλά εν ώψη του χρονικού ορίζοντα 2040-2050. Και θα πρέπει ταυτόχρονα να διορθώσουμε την κατάσταση με μια σφαιρική προσέγγιση και ε, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και τη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου. Σας ευχαριστώ θερμά, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ θερμά τους εμπειρογνώμονες από το πάνελ μας και πιστεύω ότι και οι νέοι Γεωργοί έμειναν ικανοποιημένοι από τη σημερινή δημόσια κρόση και από την ε, έμφαση που δώσαμε στο θέμα αυτό των νέων γεωργών. Και ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής των Περιφερειών. Ο Πέραμε τώρα στο επόμενο σημείο. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριο Σταγιάννη, είναι πεπισμένο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίξει πιο σημαντικό ρόλο στην ε, μελλοντική διάσκεψη κορυφή Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής που θα γίνει στην ε, Αμπιτζάν 29 και 30 Νοεμβρίου και γι' αυτό ε, στην εβδομάδα της Αφρικής που ξεκίνησε στις 20 Νοεμβρίου ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσε τις επιτροπές να περιλάβουν στις ε, συνεδριάσεις τους και ένα θέμα για την Αφρική. Εμείς ε, έχουμε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας έχουμε συνήθως εκπροσώπους από τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη στην Επιτροπή μας και έχουμε ε, τον κύριο Κλάρκε λοιπόν από την DG Άγκρη και από την ε, Γενική Διεύθυνση ε, Αναπτυξιακής Συνεργασίας έχουμε τον κύριο Λέοναρντ Μίτσι. Σε αυτούς τους δύο εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δώσω το λόγο για να μας ενημερώσουν για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ε, νέους γεωργούς στην Αφρική. Καλώς ορίσατε κύριε Κλάρκ και κύριε Μίτσι από την Άγκρη και την Δεύκο. Ε, αποφασίστε μεταξύ σας ποιος θα μιλήσει πρώτος. Παρακαλώ. Well, thank Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μου φαίνεται πως μιλάω σε μια άδεια αλλά φαντάζομαι θα έρθουν και άλλοι συνάδελφοι. Είναι εξαιρετικά επίκαιρη αυτή η συζήτηση. Έχουμε τη Συνόδο Κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Αφρική ε, την ερχόμενη εβδομάδα στην Ακτή το βασική θεματική είναι η επένδυση στου νέου. Ξέρετε ότι οι οικονομικέ και κοινωνικέ αλλαγέ που λαμβάνουν χώρα στην Αφρική είναι δραματικέ. Η δημογραφική ε, εξέλιξη ε, είναι απίστευτη. Θα έχουμε διπλασιασμό. Ε, του, του, του πληθυσμού από 2,2 δις 4,4 δις ε, ένα δις μεσαία τάξη ε, και ένα μεγάλο ποσοστό επίσης θα είναι γεωργοί. Η γεωργία ε, εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή 33% του ΑΕΠ, παράγει 33% του ΑΕΠ της Αφρικής. Θα πρέπει λοιπόν κάθε χρόνο να προκύπτουν νέες θέσεις, 18 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας για να καλύπτεται μόνο και μόνο αυτή η αγορά εργασίας και ο τομέας διατροφής και γεωργία είναι ο μόνος τομέας που μπορεί να δημιουργήσει αυτές τις θέσεις απασχόλησης. Η γεωργική ανάπτυξη λοιπόν είναι κεντρική σημασίας για να μπορέσει η Αφρική ε, να ε, αλλάξει οικονομικά με επιτυχία. Εφόσον το πολιτικό πλαίσιο είναι το κατάλληλο, εφόσον αναπτυχθεί αυτός ο γεωργικός διατροφικός τομέας με κατάλληλο τρόπο, ε, γη υπάρχει, η παραγωγικότητα είναι πολύ μικρή όμως ε, και αυτή τη στιγμή έχουμε κυρίως εξαγωγή πρώτων υλών ε, και προϊόντων ε, πώς μπορεί να συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε ιδιαίτερα οι νέοι γεωργοί να βοηθηθούν. Καταρχήν πρέπει η επιπτώση της δικής μας εμπορικής και γεωργικής πολιτικής να υποστηρίζει την ανάπτυξη τη γεωργίας στην Αφρική. Τα τελευταία 25 χρόνια και η γεωργική πολιτική έχει περάσει από πολλέ σημαντικέ μεταρρυθμίσεις που έχουν ελαχιστοποιήσει τι παρεμβάσει, έχουν καταστήσει ε, την πολιτική προσανατολισμένη προ την αγορά και έχουν, έχουν απαλληφθεί και κάποιε στρεβλώσει στην αγορά, κάποιε επιδοτήσει, οι περισσότερε ε, ενισχύσει, δεν είναι πλέον συνδεδεμένες, έχουμε ένα πολύ ανοιχτό καθεστώς ε, εμπορικό σε ό,τι αφορά ε, τα προϊόντα, ε, τα γεωργικά και διατροφικά που προέρχονται από την Αφρική μέσω του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων, ε, των εταιρικών σχέσεων στο γεωργικό τομέα. Όλες οι χώρες ΑΚΕ αυτή τη στιγμή χαίρουν πλήρους μηδενικού δασμού μάλλον για όλα τα προϊόντα τους και τα EPA, αυτές οι συμφωνίες εταιρικής σχέση επίσης δίνουν μεγάλο περιθώριο στην γεωργία από την Αφρική ε, είναι εκτός ε, των, ε, της απελευθέρωσης η, όλη αυτή η λεπτή τομή, η ευαίσθητη, η λεπτή, η η ευαίσθητη, η οι πιο νέοι γεωργοί τώρα, οι πιο δραστήριοι είναι σε καλύτερη θέση για να ξεκινήσουν εμπόριο και εξαγωγή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως πληρώνονται καλύτερα αυτές οι δουλειές από ότι άλλες το αποτέλεσμα της εμπορικής μας πολιτικής ε, στον τομέα της χειοργίας είμαστε ξέρετε το μεγαλύτερος εξαγωγίας αλλά και εισαγωγέας ε, διατροφικών προϊόντων αλλά είμαστε σίγουρα ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ε, αγροτικών προϊόντων από την Αφρική και από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ε, εισάγουμε ε, περισσότερο από, την, από τις νομισμένες Πολιτείες, την Κίνα, τη Ρωσία, την Ιαπωνία και τον Καναδά μαζί ε, αντιλαμβάνεστε ότι είναι αρκετά εντυπωσιακό αυτό το στοιχείο. Επίσης ενθαρρύνουμε τους νέους γεωργούς στην Αφρική ε, μέσω της διαμόρφωσης πολιτικής ε, έως πριν από μερικά χρόνια ο τομέας ο γεωργικός διατροφικός ήταν παραμελημένος ε, από την εξουσία αυτή τη στιγμή πολλές χώρες της Αφρικής αντιλαμβάνονται ότι ο τομέας της γεωργίας και της διατροφής όλη η αλυσίδα αυτή δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, δημιουργεί ανάπτυξη ε, και εμείς λοιπόν και αυτοί επικεντρωνόμαστε ε, στο να επιλέξουμε τις κατάλληλες πολιτικές στον ΦΑΟ, στην G20, στο G7 συνεχίζουμε τις προσπάθειες, ενισχύουμε τις προσπάθειες για να ε, καθοριστεί μια πολιτική γεωργική στην Αφρική. Και η γεωργική πολιτική όλο και πιο συχνά θεωρείται ένα καλό μοντέλο διότι ε, παραμένει, κρατά ζωντανή την Ήπεθρο και ε, χρησιμοποιεί τι βέλτιστες πρακτικέ από την κάθε περιοχή της Ευρώπης. Ε, είναι το, το κατάλληλο σημείο αφετηρίας ε, το να υπάρξουν δηλαδή κατάλληλε πρακτικέ πρακτικές όταν ε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια νέα γεωργία. επίση είμαστε σε επαφή και με την Αφρικανική Ένωση, την οποία θα συναντήσουμε και την επόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε οι περιφερειακές δυνατότητες του τη γεωργίας να αναπτυχθούν. Θα πρέπει να βρεθούν τα κατάλληλα μέσα έτσι ώστε η Γεωργία να γίνει ελκυστική για του νέου ανθρώπου. Η συζήτηση μόλι είχατε το έδειξε αυτό. Να χρησιμοποιήσουμε τι νέε τεχνολογίε, τα big data, ε, την ε, βιομηχάνηση, την εκβιομηχάνηση. Ε, θα πρέπει να υπάρχει προσταμένη αξία των γεωργών να συμμετέχουν στην διατροφική αλυσίδα. Οι νέοι γεωργοί βεβαίω είναι πιο πιθανό να αγκαλιάσουν τι νέε τεχνολογίε. Είναι θέμα επαγγελματικοποίηση του γεωργού, εν να, να πρέπει ο, η γεωργία να μην είναι απλώς ένα μέσο επιβίωσης, να, επιβίωσης, να γίνει μια μικρομεσαία επιχείρηση, ε, ε, να γίνει ένας επιχειρηματίας ή μία επιχειρηματίας πιο συχνά. Ε, πρέπει επίσης να υπάρχει μεγαλύτερη προσθέμενη αξία για τον Γεωργό στην διατροφική αλυσίδα. Να υπάρχει το κατάλληλη, κατάλληλη πολιτική έτσι ώστε να είναι καλύτερα οργανωμένοι οι Γεωργοί και να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή ε, στην διατροφική αλυσίδα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη και πολύ μεγαλύτερο στην Αφρική θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι γεωργοί και οι διατροφικές εταιρείες ε, είναι αντίπαλοι. Αυτή είναι η εντύπωση, αυτή είναι η προσέγγιση αυτή τη στιγμή και πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η γεωργία θα γίνει πιο ελκυστική, πιο ελκυστικό επάγγελμα για του νέου ανθρώπου στην Αφρική. Αυτά είναι ε, κάποια από τα ζητήματα σε ό,τι αφορά συνεργασία μα με την Αφρικανική Ένωση. Εμεί αναγνωρίζουμε ε, το κρίσιμο ρόλο του τομέα της γεωργίας και της διατροφής για τη μείωση της φτώχειας, για την ανάπτυξη, για την διατροφική ασφάλεια. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε να αντικοποιήσουμε ε, και να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας με την Αφρικανική Ένωση και να διαθέσουμε κάποιους πόρους γι' αυτό. Η συνεργασία λοιπόν για να υπάρξουν οι κατάλληλες πολιτικές και να υπάρξει και η κατάλληλη όμως ενίσχυση από εκεί και πέρα νομίζω θα αναφερθεί στη συνέχεια ο συνάδελφος από την ΤΕΦΚΟ θα δώσω τώρα κάποια παραδείγματα πρωτοβουλειών που έχουμε αναλάβει με την ε, Αφρικανική Ένωση μέτρα για να μπορέσει να καταπολεμηθεί ο κοινωνικό αποκλεισμό στην Ήπεθρο υποστήριξη για την βιο ε, για αγροβιομηχανικά πάρκα και τη χρήση νέων τεχνολογιών, συμμετοχή στην ΟΖΟΤΑ 2020 στα προγράμματα έρευνας και Αφρικανών και, Αφρικανών και δημιουργία SPS ε, για την ασφάλεια των τροφίμων, για το περιβάλλον και την έξυπνη γεωργία. Εξετάζουμε πιλωτικά προγράμματα έτσι ώστε να καταρτήσουμε, να καταρτήσουμε πιο επαγγελματίε του ε, γεωργού τη Αφρική με τη βοήθεια ευρωπαϊκών οργανώσεων γεωργών και καθώς και συστήματα ανταλλαγής, προγράμματα ανταλλαγής μάλλον. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να δημιουργήσουμε προσθέμενη αξία στην αφρικανική γεωργία και στην στα αφρικανικά τρόφιμα. Ένα από τα παραδείγματα τα οποία θα ε, εγκριθούν την ερχόμενη εβδομάδα στον Σύνοδο Κορφή είναι μια στρατηγική για τα ποιοτικά προϊόντα, για γεωγραφικές ενδείξεις στην Αφρική. Διότι στην Αφρική υπάρχει πλούσια κληρονομιά σε επίπεδο διατροφή και πολλέ ενδεχόμενε γεωγραφικέ ενδείξει που πρέπει να αναπτυχθούν και να δώσουν περισσότερο περισσότερη ποιότητα στο προϊόν που συνεργαζόμαστε λοιπόν με την Αφρικανική Ένωση έτσι ώστε ε, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη συμφόρηση που υπάρχει στις επενδύσεις στα σημεία δηλαδή ε, όπου σκοντάφτουν ε, υπάρχει διακυβερνητική διάσταση Προσπαθούμε όμως να, να συνεργαστούμε και από τον ιδιωτικό τομέα της Αφρικής. Εμείς ε, θα δίνουμε νέες συμπράξεις, νέες ε, επενδυτικές ε, προσπάθειες. Ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα να, να επενδύσουν στην Αφρική, σε ό,τι αφορά τη γεωργία. Είναι πολλές οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Οι εταιρείε μας θέλουν να επενδύσουν στην Αφρική θα πάμε την ερχόμενη εβδομάδα στο Αμπιτζάν για την Σύνοδο Κορυφή μαζί με τη Food Drink Europe για να έχουμε μια πιο δομημένη σχέση μεταξύ Ελλήνων και Αφρικανικών, ε, ευρωπαϊκών και αφρικανικών επιχειρήσεων στον τομέα της γεωργίας. Βέβαια, πρέπει να είναι υπεύθυνη ε, αυτή η σχέση, δεν πρέπει να αποφύγουμε την αρπαγή γης. Ε, ο συνάδελφος θα εξηγήσει φαντάζομαι και το νέο σχέδιο εξωτερικών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα χρησιμοποιήσουν οι επενδυτές ε, για να μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτές τις άμεσες επενδύσεις. Να πω ότι αυτή η έμφαση που δίνουμε στο να, συμμετάσχει ο ιδιωτικό τομέα με τις ε, επενδύσεις του και να επιλεγεί η κατάλληλη πολιτική είναι τα σημεία κλειδιά τα τελευταία πέντε χρόνια, πέντε χρόνια αποτυπώνεται εδώ το γεγονός ότι η ιδιωτική ε, ε, επένδυση είναι πολύ πιο σημαντική από την ενίσχυση ε, να έχουμε μια σχέση που να μην είναι νεοαπικιακή ε, να είναι μια σχέση συνεργασίας ε, χρειάζονται κατάλληλες πολιτικές έτσι ώστε να ενισχύσουμε τις επενδύσεις στον τομέα της γεωργίας και της διατροφής και ελπίζω ο Συνός Κορυφής να είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή και αν το πετύχουμε αυτό τότε οι Αφρικανοί θα αντιληφθούν και αυτοί τις δυνατότητες που έχουν σε επίπεδο ανάπτυξης, σε επίπεδο απασχόληση και αυτή η δημογραφική έκρηξη να ε, ε, γίνει μια, ένας θετικός παράγοντας ε, έτσι ώστε και βεβαίως οι νέοι Γεωργοί να μπορούν να στο έπακρο αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Χαίρομαι που μας κάνατε τη σύνδεση με το προηγούμενο θέμα των νέων γεωργών. Ο κύριος Λέναρτ Μίτσι από τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ και καλησπέρα σας. Πόσο χαίρομαι που ξανάρχομαι στην Γενική Διεύθυνση, στην Επιτροπή Γεωργίας ένα χρόνο αφού άφησε την, τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πάντως ε, δείχνει πόσο ε, συνεργατική είναι η συνεργασία μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν ώψη της ε, διάσκεψης κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής και κατά τη διάρκεια της και μάλιστα θα είναι πολύ στελεχωμένη καλά η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αμπιτζάν και έχουμε και το Business Forum λίγο πριν και είναι σημαντικό ότι η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα έχει κέρια σημασία στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την οικονομική ανάπτυξη και μάλιστα πολλό δε μάλλον που θέμα της ε, διάσκεψης κορυφής είναι το βιώσιμο μέλλον της Αφρικής. Ένα βιώσιμο μέλος για την Αφρική δεν νοείται χωρίς ε, αηφόρο ανάπτυξη και βιώσιμες θέσεις απασχόλησης. Ε, που φυσικά θα συνεκτιμά και τη διάσταση του φύλου. Αυτό είναι σημαντικό ε, αποτέλεσμα που προσβλέπουμε να προκύψει στην Αμπιτζάν και διαπιστώνουμε ότι τέσσερις είναι βασικές κλάδες της ε, διάσκεψης. Ε, ε, επαιδείουμε στους ανθρώπους στην τεχνολογία, στην ανάπτυξη δεξιότητες, επίσης ε, ανάπτυξη ανθεκτικότητες, διαχείριση της κινητικότητας και της μετανάστευσης και το τέταρτο κινητοποίηση των επενδύσεων για, την ε, για το βιώσιμο μετασχηματισμό της ε, αφρικανικής οικονομίας. Όπως είπε και ο Τζον πριν από λίγο, ε, θέλουμε μια πιο σφαιρική προσέγγιση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη νεολαία στην Αφρικανική Ήπειρο. Μάλιστα, τους τελευταίους μήνες επισκεφτήκαμε πολλές χώρες και έχουμε ευρύ χαρτοφυλάκιο στην ΤΕΦΚΟ ε, για το 2014-2020 και περίπου 9 δισεκατομμύρια προπολογισμό. Ε, το μεγαλύτερο τμήμα το αφορά χώρε τη υποσαχάριου Αφρική. Το θέμα όμω δεν είναι μόνο οικονομικό, μόνο χρηματικό. Χρειαζόμαστε ένα κατάλληλο σχέδιο πολιτική, ε, διακυβέρνηση και τα σωστά μηνύματα της πολιτικής, γιατί μόνο έτσι θα προσελκύσουμε νέους ε, στη γεωργία και στον αγροτροφικό κλάδο. Θα πρέπει λοιπόν να διαφυλάξουμε τις επενδύσεις εκεί. Και αν δούμε ε, τι έγινε μέχρι τώρα, θα, κάτι που θα επικαιρώσουμε την επόμενη εβδομάδα, σίγουρα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις δεξιότητες, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και ένα θέμα που επανέρχεται στις, ε, στους Υπουργούς Γεωργίας είναι ε, μια γεωργική πολιτική και γεωργία που θα στηρίζεται όμως από εκτεταμένες υπηρεσίες ε, και αλλού. Και μάλιστα η γεωργική έρευνα για την ανάπτυξη είναι σημαντική και καινοτόμα συστήματα που θα αντικατοπτρίζουν τις προκλήσεις και, τις, και των κλιματικών αλλαγών. Λίγο πριν ε, ολοκληρώσαμε την ΚΟΠ στη Βόνη, όπου και θα έχουμε και το Δεκέμβριο στο Παρίσι συνέχιση, θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις κλιματικές αλλαγές και να αξιοποιήσουμε τα μέσα που μας δίνουν συστήματα γεωργικής και ανατομίας, ώστε να προσελκύσουμε νέους σε γεωργικά και γεωργοτροφικά συστήματα που θα προσαρμόζονται όμως στις κλιματικές αλλαγές. Δύο μείζονες προκλήσεις και δύο ε, βασικά αιτήματα χρηματοδότησης που λαμβάνουμε πρόσφατα και που αφορούν τους επιβλαβείς οργανισμούς και τις αρρώστιες. Ε, ε, Καταρχήν έχουμε ένα σκόλικα, ε, έναν επιβλαβή οργανισμό που θερίζει πολλές καλλιέργειες στην Αφρική και κυρίως την πανόλη των μικρών μερικαστικών που πλήττει κυρίως τα εγωπρόβατα. Πάντως συνεργαζόμαστε στενά με τη ΦΑΟ και την ΟΑΗ προκειμένου να καταπολεμήσουμε επιβλαβείς οργανισμούς και επιζωνο, Η ανθεκτικότητα φυσικά είναι κλειδί, γιατί χωρίς ανθεκτικότητα δεν θα έχουμε μέλλον για τους νέους. Έχουμε πολλούς ε, ε, εταίρους, τη ΦΑΟ, WFP, ε, τις Ηνωμένε Πολιτείες και μάλιστα θα έχουμε μια παγκόσμια έκθεση για την επισητιστική κρίση ε, κάτι που δείχνει πόσο σημαντικό είναι να έχουμε και ανθρωπιστική προσέγγιση και πιο ε, καλή πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια, ώστε να έχουμε και έγκαιρη προειδοποίηση και ε, έγκαιρη δράση. Μάλιστα χρησιμοποιούμε όλα τα συστήματα για δορυφορικού σχεδιασμού και τεχνολογίες των πληροφοριών, ώστε να προλάβουμε κινδύνους που αφορούν τις κλιματικές αλλαγές το φαινόμενο Ελνίνιο ή Λανίνιο, γιατί κάποιες ε, μετεωρολογικές προγνώσεις ε, δεν είναι και πολύ αισιόδοξε για τους επόμενους μήνες. Ε, είχαμε πρόσφατα δημοσιεύματα στον παγκόσμιο τύπο, γι' αυτό και θα πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα μέσα πολιτικής και τους κατάλληλους μηχανισμούς και φυσικά και μέσα διαχείρισης των κινδύνων για τους νέου γεωργού και στην Αφρική για να προλάβουμε τέτοιου κινδύνου. Κινητοποίηση επενδύσεων. Αναφέρθηκε από τον Τζόνο ότι χρειαζόμαστε ένα περιβάλλον ολιστικής ε, πολιτικής. Ε, χρησιμοποιούμε τα υπάρχοντα εργαλεία και τις ε, πλατφόρμες, όχι μόνο την Κάντεπ. Κάντεπ για μας είναι το κλειδί. Πρόκειται για εργαλεία που έχουν άμεση σχέση με συγκεκριμένες χώρες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ε, να υπάρχει μια πολυεπίπεδη συμμετοχή που θα περιλαμβάνει και νέους αλλά και γυναίκες και γυναίκες ηγέτες. Μόλις ε, δημοσιεύσαμε ένα έγγραφο για το πώς να λαμβάνεται η διάσταση του φύλου στα προγράμματα της γεωργίας, ε, στα προγράμματα διατροφής, αλλά και πώς να προσελκύονται οι νέοι στις γεωργικές ε, επενδύσεις. Έτσι λοιπόν φτάνω στο θέμα του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Προγράμματος. Όπως ξέρετε αυτό είναι η ναυαρχίδα μας η ναυαρχίδα στο να ε, ενισχύσουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις, ε, στο ε, προσελκύσουμε επενδύσει, προσφέροντα όχι μόνο νέε εγγύσει μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο αλλά και για να βρούμε ε, πρόθυμους να αναλαμβάνουν κινδύνους στον τομέα της γεωργίας που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και είναι πολύ δύσκολο οι εμπορικές τράπεζες ε, να εμπλακούν στη γεωργία. Αυτό όμως είναι εκ των όνων αν θέλουμε να προσφέρουμε ευκαιρίες για νέους επιχειρηματίες, κυρίως στους νέους ανθρώπους. Όλα αυτά θα συμπληρωθούν και με επιπρόσθετες χρηματοδοτήσεις που έχουν και τον πυλώνα 1 και τον πυλώνα 2 του προγράμματος εξωτερικών επενδύσεων. Ο στόχος λοιπόν είναι απόλυτα να βελτιωθεί το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον όπως ε, και τα τραπεζικά επιλέξιμα προγράμματα για να υπάρξει ε, δυναμισμός ε, και εκβιομηχάνηση κάτι το οποίο δεν υπάρχει ιδιαίτερα στις περισσότερες αφρικανικές χώρες. Ο Τζον είπε ότι υπάρχει και αυτή η ιδέα του να ε, εμπλακούν στην όλη υπόθεση και εταιρείε εταιρείες ε, παραγωγής ε, τροφίμων. Εμείς το θέλουμε αυτό για να ενισχύσουμε το διάλογο ανάμεσα στον αφρικανικό και τον ευρωπαϊκό ιδιωτικό τομέα. Γιατί αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε φραγμούς και ευκαιρίες επενδύσεις. Η ιδέα λοιπόν είναι να χρησιμοποιήσουμε περίπου 4,1 δις κοινοτικό χρήμα για μόχλη για κινητοποίηση, ε, να φτάσουμε περίπου τελικά στα 44 δις ε, ευρώ επιπρόσθετες επενδύσεις. Ε, θεωρούμε ότι αυτό είναι σημαντικό γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν ευημερούσες ε, γεωργικές περιοχές αν δεν έχει κανείς ολιστική προσέγγιση γενικότερα ως προς τις απαραίτητες επενδύσεις. Θα υπάρξουν λοιπόν πολλά παράθυρα και πέρα από τη γεωργία που θα είναι ανοιχτά. Στο Αμπιτζάν θα έχουμε το εναρκτήριο λάκτισμα μιας νέας διαδικασίας και νέων επενδύσεων. Θα ξεκινήσουμε με περιοχές ε, ε, που να έχουν ζωντανή γεωργία. Ε, να μην είναι απαραίτητα περιοχές όπου είναι κανείς αναγκασμένος ε, να μεταναστεύσει, να εγκαταλείψει τις γεωργικές περιοχές και να πάει σε αυτά τα σλάμ των μεγαλοπόλεων στην Αφρική. Αυτό που χρειάζεται είναι συστήματα αλλαγών, μια πιο περιφερειακή διάσταση και προσέγγιση από αυτή την παραδοσιακή προσέγγιση τις γεωργίες που χρησιμοποιήθηκε κατά τα προηγούμενα στις προηγούμενες δεκαετίες. Μετά, το ψηφιακό θεματολόγιο. Οι νέοι και αυτοί πρέπει να προσελκυστούν ε, στο, στην ψηφιακή θεματολογία, να χρησιμοποιούνται περισσότερα κινητά. Υπάρχουν τώρα αυτά στις ε, περισσότερες ε, αφρικανικές χώρες, να χρησιμοποιούνται περισσότερα δορυφορικά συστήματα, καθαρή ενέργεια, να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο Τζον αναφέρθηκε στην αλυσίδα αξίας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι περίπλοκο στις ε, αφρικανικές ε, κοινότητες. Σιγά σιγά πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την προσέγγιση που βασίζεται σε προϊόντα και να περάσουμε σε μια άλλη προσέγγιση. Ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να εξετάζουμε συγκεκριμένα προϊόντα στο Business Forum θα έχουμε και εκεί την ευκαιρία να δούμε το πώς μπορούμε να αυξήσουμε την αξία μέσα από ε, αηφόρα προγράμματα. Υπάρχει ε, μία σειρά ε, παραγόντων που θα προσθέσουν στην αλίδα, αλυσίδα αξίας. Εδώ θα παίξουν ρόλο και ο καφές και το βαμβάκι στο πλαίσιο αυτής της αλυσίδας αξιών. Αναφέραμε ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν με μία προσέγγιση που είναι χωρίς ε, αποκλεισμούς είτε πρόκειται και για ε, ε, υπεύθυνε επενδύσεις. Εμείς ε, νομίζω είμαστε απόλυτα σαφείς. Και τέλος αναφέρθηκε το D72 70 το 2070 αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ε, ακολουθήσουμε το χάρτη των Βρυξελών. Τώρα πλέον θα τον ε, υιοθετήσουμε, θα υιοθετηθεί και από την Προεδρία της Αργεντινής. Ισχυρή συνεργασία, ανάμεσα ε, στον ΦΑΟ, την ΙΦΑΤ και πολλούς άλλους διεθνείς οργανισμούς. Και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη αξιολόγηση των παρεμβάσεών μας. Είναι σημαντικό να δείχνουμε ε, ποιες είναι οι επιπτώσεις που προκύπτουν έτσι ώστε ό,τι και αν γίνει μετά το 2020 να είναι απόλυτα σαφές ότι υπάρχουν ουσιαστικές ε, επιπτώσεις στις επενδύσεις μας, στις ε, παρεμβάσεις μας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα ήθελα να πάρουν το λόγο τώρα ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ πολύ μιλάμε για την Αφρική και υπάρχει ένας ελέφοντα, ελέφαντας στο δωμάτιο, ο οποίος δεν αναφέρθηκε. Είναι η επιπτώση του γεγονός ότι οι Κινέζοι ε, επικίζουν την ε, Αφρική. Τρακτέρ, ε, ορυχεία, είναι η πραγματικότητα αυτή, συμβαίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον ρόλο να παίξει στην Αφρική. Μπορούμε βεβαίως να μιλάμε με ντροπή για την συμπεριφορά μας από 100 χρόνια, ενώ η Κίνα αυτή τη στιγμή το πάει ακόμα παραπέρα. Θεωρούν ότι η Αφρική είναι το κήπος τους, το μποστάνι τους. Λοιπόν, έχετε συναντήσει την Κίνα ε, σε αυτά τα, τα ταξίδια στην Αφρική. Αν δεν το έχετε κάνει, θα, κάποια στιγμή θα τη βρείτε μπροστά σας. Και ποιος θα κερδίσει τότε. οι Αφρικανοί δεν φαίνεται να μπορούν οι ίδιοι ε, να, να βγάλουν μια άκρη και να πάρουν μπροστά παρά τους πόρους που έχουν. Γιατί δεν έγινε αναφορά στην Κίνα, μας περιπτώσει. Ε, και εφόσον την αναφέρουμε, τι θα κάνουμε για αυτήν, πέρα από την αναφέρουμε. Μάλιστα, ευχαριστώ και ο αν έχει το λόγο. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το ζήτημα αυτό. Είναι ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Πρώτον, συχνά μιλάμε για την κρίση των προσφύγων και το τι θα κάνουμε και γενικότερα είναι μια αντίδραση αυτή σε αυτό που συμβαίνει. Εσείς μιλάτε για κάτι όμως, ε, για μια δράση, για μια ενεργή δράση. Τώρα το πώς σκοπεύετε να το κάνετε, εντάξει, μπορεί να μην συμφωνούμε 100%. Αλλά η ιδέα είναι μια πολύ καλή ιδέα. Εγώ προέρχομαι από την Ιρλανδία. Μια χώρα που ημωράγησε για εκατοντάδες χρόνια. 19 στους 20 από την οικογένειά μου πήγαν στο Λονδίνο και στο παρελθόν εκατομμύρια άνθρωποι έφυγαν από το νησί μας και δεν έφυγαν επειδή δεν τους άρεσε ε, το τοπίο και ο καιρός στην Ιρλανδία οι γείτονές τους έφυγαν γιατί δεν είχαν καμία επιλογή και αν τα πράγματα βελτιωθούν ε, βελτιωνόντουσαν στην Ιρλανδία θα γύριζαν. Τώρα ας πούμε μένουν. Το ίδιο ισχύει για την Αφρική. Αυτή είναι η λύση. Αυτό που με ανησυχεί όμως είναι ότι ενώ έχουμε με τόσο σημαντική παρουσίαση βρίσκονται εδώ μόνο τρεις ευρωβουλευτές. Δεν υπάρχει κάποιο σύστημα απαρτίας εδώ για να εξασφαλίζουμε να... Ε, ότι οι άνθρωποι θα είναι εδώ, οι βουλευτές. Ε, είναι λάθο. είναι πραγματικά λάθος το που συμβαίνει. Πού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα πρέπει να είναι εδώ σήμερα αυτή τη στιγμή. Κύριε Βουλευτά. Οφ, ίσως καλό θα είναι αποφεύγουμε τέτοια σχόλια, γιατί είναι πέμπτη απόγευμα, πολλοί έχουν προγραμματίσει ταξίδια και ούτω καθεξής. Ο κύριος Μπόγκοβιτς. Και εγώ θα προτιμούσα να είναι πιο γεμάτη η αίθουσα, αλλά ελπίζω ότι, αν μη τι άλλο, μας παρακολουθούν από το γραφείο τους οι συνάδελφοι. Γιατί συζητάμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και αντιμετωπίζουμε πολλοί άριθμες προκλήσεις. Μιλούμε για την Αφρική, μία ήπειρο, όπου έχει διπλάσιο πληθυσμό και μάλιστα ο πληθυσμός αυτός θα διπλασιαστεί μέχρι το 2060 ε, θα διπλασιαστεί στην Αφρική και θα τετραπλασιαστεί ο αφρικανικός πληθυσμός σε σχέση με τον ευρωπαϊκό. Οπότε θα είναι σημαντική η επίδραση της Αφρικής ε, και στον παγκόσμιο πληθυσμό, στην παγκόσμια κατάσταση. Νομίζω ότι έχουμε το καθήκον να βοηθήσουμε την Αφρική που είναι πολύ ζορισμένη σήμερα και αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Και δεν θέλω να επιστρέψουμε ως απεικιοκρατικές δυνάμεις όπως κάναμε για πολλούς αιώνες μέχρι τον περασμένο αιώνα. Θα πρέπει να στηρίζουμε συστηματικά και να επικορούμε ε, εκείνους που θέλουν να αναπτύξουν ε, την Αφρικανική Ήπειρο. Να βοηθήσουμε ε, τέτοιες δυνάμεις αναπτυξιακές. Ε, να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη, τη γεωργία, την συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου Μόνο έτσι θα ανταποκριθούμε στις ε, προκλήσεις της Αφρικής που είναι και περιβαλλοντικές, κλιματικές, οικονομικές, αλλά ε, και η μεταναστευτική κρίση που πλήττει και άλλες περιοχές του κόσμου. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια σφαιρική προσέγγιση και να εγκρίνουμε πολιτικές που θα τονώσουν την ανάπτυξη και στην Αφρική. Πιστεύω ότι έτσι η εξωτερική μας πολιτική θα είναι αρκετά σοφή και στοχευμένη ώστε ο πολιτικός μας ρόλος στην Αφρική να είναι αντάξιος της οικονομικής μας συμμετοχής στην αναπτυξιακή βοήθεια. Γιατί είναι σωστό για την Ευρώπη να παρέχει βιώσιμη αρρωγή στην Αφρική, αλλά να ασκήσει και κάποιο πολιτικό ρόλο για να εξασφαλίσει αηφόρο ανάπτυξη και στο μέλλον για την Ήπειρο αυτή. Την Παγκόσμια ημέρα τροφίμων, που ήταν 16 Οκτωβρίου, με πρωτοβουλία της ΦΑΟ, και ο Πάπας Φραγκίσκος μίλησε για το πώς θα πρέπει να εμπλέξουμε και τους πρόσφυγες και μετανάστες στην οικονομική ανάπτυξη, να εξασφαλίσουμε πρόσβαση στο πόσιμο ε, είδος, στα τρόφιμα, αλλά και γενικώ στις υποδομές, γιατί αυτό αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε. Γιατί πολύ συχνά εμείς ως υπέρμαχοι και ε, πρωτεργάτες της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής. Κατηγορούμαστε γιατί η κοινή γεωρική πολιτική που σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους Ευρωπαίους αγρότες επηρεάζει παρόλα αυτά αρνητικά τους αγρότες άλλων χωρών και δι τους αγρότες της Αφρικής. Δεν είναι αυτός φυσικά ο στόχος ούτε θα θέλαμε τέτοια αποτελέσματα της κοινής γεωρικής πολιτικής. Και η βοήθεια που προσφέρουμε στην Αφρική θα πρέπει στο μέτρο του δυνατού να ενισχύει την παραγωγή και να δημιουργεί προϋποθέσεις ε, για καλύτερη παιδεία, καλύτερη κατάρτιση. Ε, γιατί είναι αυτό το γνωστό, αν θα πρέπει να δώσουμε ψάρι, να δώσουμε αγκίστρι για να ψαρεύει ο κόσμος. Αναφέρθηκαν τα προβλήματα πρόσβασης το πόσιμο είδωρα, ε, στα τρόφιμα, αλλά και αντιμετώπιση ε, ασθενειών ή επιβλαβών οργανισμών. Και εκεί θα πρέπει ανεπιφύλακτα να προσφέρουμε τη βοήθειά μας στην Αφρική ε, και να τη βοηθήσουμε στον αγώνα της ε, για την προστασία του περιβάλλοντος. Πολλές προκλήσεις ε, στα πλαίσια και της παγκοσμιοποίησης των παγκόσμιων συναλλαγών και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους παγκόσμιους οργανισμούς που παρέχουν ε, την πιο δαψιλή βοήθεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Σίγουρα θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό. Και αν θέλετε μπορώ να σας ξαναδώσω το λόγο για να ασχολιάσετε. Ε, Παρακαλώ, κύριε Δευθυντές, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Τρία σύντομα σχόλια. Ο ελέφαντας στην αίθουσα είναι η μετανάστευση και η επιρροή της ΚΑΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες. Δίκαιο έχετε ότι είναι κάτι που δεν το αντιμετωπίζουμε άμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως φαντάζομαι ότι είναι αρνητικό το αποτύπωμα που αφήνει η κινέζικη γεωργία στην Αφρική. Ε, βέβαια, ο κινέζικος ιδιωτικός τομέας είναι ιδιαίτερα παρόν εκεί ε, και μέσως και ο κινέζικος κρατικός παράγοντας. Μερικές επενδύσεις βέβαια είναι ευνοϊκές για τις ενδιαφερόμενες χώρες γιατί ε, προσφέρει υποδομές, σιδηροδρομικές συνδέσεις, ε, κατασκευάζει λιμάνια, πολλές υποδομές δηλαδή κατασκευάζει Κίνα στην Αφρική που ωφελούν τις ε, χώρες αποδέκτες, αλλά μερικές από τις επενδύσεις αυτές, η κινέζικη παρουσία γενικώ στην Αφρική, σε πολλές περιπτώσεις είναι επιζήμια. Γιατί πρόκειται για μεγάλες κλίμακος α, ε, γεωργία και κυρίω ε, κυρίως στόχο έχει τις ε, εξαγωγές που θέλουν να διασφαλίσουν την επιστηστική ασφάλεια της Κίνας και όχι της Αφρικής και είναι περισσότερο το προϊόν πολιτικής μόχλευσης ε, και επιρροής που έχει μια ισχυρή χώρα σε πιο δύναμες χώρες. Πάντως προσπαθούμε ε, και με τις χώρες της ε, G7 και την Κίνα να καταλήξουμε σε συμφωνία προκειμένου να έχουμε υπεύθυνε επενδύσεις στην Αφρική. Γιατί υπάρχουν κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές και από τον ΩΣΑ και από άλλες οργανώσεις που προβλέπουν τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Και ε, η Κίνα υποσχέθηκε ότι θα ελέγξει ε, τους επενδυτές γιατί έχει προσυπογράψει αυτές τις κατευθυντήρες γραμμές και όταν ο Σιτζιπίνκ πήγε πριν από δύο χρόνια στην Αφρική ε, απολογήθηκε, ζήτησε συγγνώμη για την αρπακτική συμπεριφορά ε, άπληστη συμπεριφορά τα κάποιων ε, κινέζικων επιχειρήσεων στην Αφρική και ότι θα το διορθώσει. Δεν ξέρω αν τήρησε βέβαια την, την υπόσχεσή του. Σε ό,τι αφορά τις ε, σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής, έχουμε και τη σχέση μας με την Αφρικανική Ένωση και αυτό θα το διασφαλίσουμε και στην επόμενη διάσκεψη κορυφής. Ε, θεσπίζουμε ένα, μια δέσμη κατευθυντηρίων γραμμών που θα υπογραφούν και από τις κυβερνήσεις και από τον ιδιωτικό τομέα. Για το τι εστί ε, υπεύθυνη προσέγγιση στις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και τι ε, προϋποθέσεις διακυβέρνηση θα πρέπει να προσφέρουν οι αφρικανικές χώρες για να προσελκύουν τις σωστές επενδύσεις. Και με αυτό το βήμα πρόοδο πιστεύω ότι θα αποδείξουμε και εμπράκτος ότι είναι προς όφελος και των Αφρικανών εταίρων μας να ενθαρρύνουν υπεύθυνε επενδύσεις και όχι μόνο ε, επιβλαβείς ε, κινέζικες επενδύσεις από κάποιες αραβικές χώρες του κόλπου. Πάντως και το θέμα των επενδύσεων ε, θα συζητηθεί στη διάσκεψη κορυφής. Και σίγουρα ένα τρόπο για να άρουμε τα κίνητρα για οικονομική και παράτυπη μετανάστευση είναι δημιουργώντας θέσει απασχόλησης και στην ύπεθρο. Και σίγουρα ο αγροτροφικός κλάδος είναι ο μόνος κλάδος που είναι κλάδος έντασης εργασία στην Αφρική και είναι ο μόνος κλάδος που μπορεί να δημιουργήσει αρκετές θέσεις εργασία για να αναχαιτήσει τις μεταναστευτικές ροές και την μεταναστευτική έξοδο από την Αφρική. Και μάλιστα πέρυσι στη διάσκεψη κορυφής της Βαλέτας δημιουργήσαμε ένα πλαίσιο στο οποίο είπαμε ότι η γεωργία και ο αγροτροφικός κλάδος είναι σημαντική Με την Ιγυρία, με το κέρας της Αφρικής ε, πρέπει να βρούμε ε, τρόπους για να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν το μεταναστευτικό πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο της ΚΑΠ που επισημάνατε κύριε Πρόεδρε, πολλοί ακόμη και σήμερα ισχυρίζονται ότι η κοινή γεωργική πολιτική ε, καταστρέφει την ε, γεωργία συντήρησης της Αφρικής, η γεωργία βιοπορισμού επιβίωσης. Όταν πέρυσι δώσαμε εξαγωγικές ε, επιδοτήσεις στα πουλερικά, φαίνεται ότι καταστράφηκαν κάποιες εκμεταλλεύσεις στην Γκάνα και σε χώρες της Δυτικής Αφρικής. Αυτό όμως ανήκει στο παρελθόν. Ήταν πριν από 20 χρόνια, συγγνώμη, δώσαμε τέτοιε ε, ενισχύσει. Αλλά αυτό ανήκει στο παρελθόν. Ε, ο Κόφι Ανάν που γνωρίζει τα πράγματα πολύ καλά ε, είπε ότι το, η ΚΑΠ είναι τόσο διαγκωμένη που επιτρέπει σε καθέναν να ταξιδεύει πρώτη θέση σε κάθε γελάδα να ταξιδεύει πρώτη θέση ε, παγκοσμίω. Και μάλιστα ένας Αυστραλός ε, υπουργό είχε πει κάτι που έμεινε παρημεώδες, ε, κάτι αντίστοιχο, αλλά αυτό είναι ανοησίες. Και μάλιστα ο κύριος Δεσίλβα από τη ΦΑΟ σε μια πρόσφατη ομιλία του είπε πόσο επιζήμια είναι η ΚΑΠ για την ανάπτυξη και χρειάστηκε να τον διορθώσουμε σε αυτή τη δήλωση. Χρειάστηκε τελικά να ανακαλέσει και να πει ότι παρεξηγήθηκαν τα λεγόμενά του. Όλα αυτά για να σας πω ότι η ισχύουσα ΚΑΠ όχι μόνο δεν έχει αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά αντίθετα έχει ευνοϊκό αποτέλεσμα. Γιατί ένα τμήμα της ΚΑΠ αφορά την εισαγωγή προϊόντων από την Αφρική. Και μπορεί να σας εκπλήσει αυτό, αλλά η ΚΑΠ είναι ε, παράδειγμα προς μίμηση για πολλές χώρες ό,τι αφορά το γεωργικό μοντέλο που θα επιλέγουν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμφωνήσω απόλυτα με αυτό που είπε ο Τζον. Όχι επειδή πριν από 10 χρόνια μου στη Τζιάγκρη, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα σε επίπεδο επικοινωνία. Υπάρχει ένα σκεπτικισμό σε κάποιες ε, περιοχές ε, της Αφρικής είναι σημαντικό αυτό διότι έχει αλλάξει η δυναμική τα τελευταία χρόνια ο ρόλος ε, της εξαγωγής των εξαγωγών από την Ασία από τη Βραζιλία ουσιαστικά μετατοπίζουν κάποιες τοπικές παραγωγές δίνει την εντύπωση ότι είναι Ευρωπαϊκή. τα ευρωπαϊκά πρέπει να το κάνουν αυτό και η κοινή πολιτική αλλά δεν είναι έτσι ε, χρειάζεται λοιπόν μια σωστή αφήγηση σε επίπεδο επικοινωνία συστηματικά και όχι αμυντικά. Αυτά ε, σε ό,τι αφορά την ατζέντα για την πολιτική ανάπτυξη. Τώρα, μόλι πριν από μια εβδομάδα ήρθα από το Μαπούτο, επειδή είπατε για την Κίνα. Οι, Κίνοι, Κινέζοι φτιάχνουν μια γέφυρα που θα συνδέει το Μαπούτο που κοστίζει 800 εκατομμύρια δολάρια. Είναι βεβαίω σαφής ε, εκεί η παρουσία τους. Έχουν βάλει που έχουν πατήσει πόδι. Και αν δείτε, είναι 181 από τις 190 χώρες στο δίκτυο ανάπτυξης, 10 ε, πιο φτωχές χώρες στον κόσμο αυτοί 800 εκατομμύρια ευρώ για μια γέφυρα, ε, αν σκεφτείτε ε, ποιες είναι οι της Μοζαμβίκης που έχει με τεράστια ακτή, 2.400 χιλιόμετρα, μεγάλες δυνατότητες, τίποτα σε επίπεδο βιομηχανοποιημένης γεωργίας, ε, γεωργία επιβίωσης. Ε, οι Κινέζοι, ναι, βρίσκονται στη Μοσαμβίκη. Εμείς θέλουμε όμως να δείξουμε προς ένα μοντέλο, ένα μοντέλο που να είναι συμπεριληπτικό και όχι απαραίτητα αυτό που προσπαθούν να προωθήσουν και να πουλήσουν στην Αφρικανική Ήπειρο οι Κινέζοι. Ένα μοντέλο το οποίο να, δίνει, να σου δίνει το δικαίωμα, να σου δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείς τη γη σου, να υπάρχουν κοινωνικές προϋποθέσεις, περιβαλλοντικές προδιαγραφές και αυτό είναι το δίλημα που έχουμε πάντα. Έγινε μια συζήτηση ε, με τους Ευρωπαίους ενδιάμεσους, οικονομικούς ενδιάμεσους, αυτοί δηλαδή που βρίσκονται μεταξύ ημών ε, και αυτών που θα οικοδομήσουν τη γέφυρα για να οδηγηθούν σε project, σε project τα οποία να είναι βιώσιμα. Εάν θέλετε, μας είπαν, ψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, είναι δύσκολο να βρεθούν projects στην Αφρική ε, τα οποία να συγκεντρώσουν χρηματοδότηση, διότι θα, είναι, θα είστε πολύ απαιτητικοί, θα ζητάτε μικρούς, κοινότητες με μικρούς ιδιοκτήτες, ε, ενώ άλλοι πουλάνε άλλα μοντέλα. Αυτό όμως είναι το δικό μας. Ε, βεβαίως μπορούμε να κάνουμε κάποιες προσαρμογές, αλλά όχι ε, κάνοντας dumping ή εν πάση περιπτώσει κάνοντας έκπτωση σε κάποιες αρχές και σε κάποιες, κάποια πρότυπα τα οποία είναι σημαντικά για μας. Το μόνο φόρουμ που μπορούμε με τους Κινέζους να συναντηθούμε όταν ήμουν στη Μοζαμβίκη ε, οι χώρες που βρίσκονται εκεί δεν είναι τόσο οι ευρωπαϊκές, είναι η Κίνα, η Τουρκία και η Ινδία. Αυτές είναι οι αυτοί είναι τρεις πέκτες κλειδιά, όχι μόνο στον τομέα της γεωργίας, ε, γενικότερα σε επίπεδο ε, κατασκευών, ανάπτυξης κτλ. Αυτό που θα πρέπει να γίνει λοιπόν είναι ε, στα πλαίσια του G20 πιο συστηματικά να το θέτουμε το θέμα με τους Κινέζους, με τους Τούρκους, με τους Ινδούς, ε, όσον αφορά το ποια είναι η συμπεριφορά τους, ποιες είναι οι αρχές που πρέπει να διέπουν ε, τις παρεμβάσεις μας εκεί και να συζητούμε βεβαίως και με την Αφρικανική Ένωση για να δούμε ε, ποιο μοντέλο είναι το πλέον κατάλληλο για την Αφρική για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Τώρα για τις ε, ρίζες του κακού. Ε, βεβαίως υπάρχουν πολλές αναλύσεις για το τι οδηγεί στην μετατόπιση των πληθυσμών, ποιες είναι οι οικονομικές μεταναστευτικές ροές, οι περισσότερες μετακινήσεις στην νότια, Αφρική ας πούμε, πάνε προς την χώρα την Νότια Αφρική από τις αγροκοινωνικές χώρες. Λίγοι πάνε προς τη Μεσόγειο ε, σε ποσοστά. Υπάρχει πολλή μετανάστευση από τον νότο προς τον νότο δηλαδή. Πρέπει όμως να τους δώσουμε τη δυνατότητα να μείνουν κοντά στην κοινότητά τους αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε αυτές τις συμπράξεις που είναι ένα πρώτο βήμα αλλά θα χρειάζεται και ισχυρή διακυβέρνηση, ισχυρούς ηγέτες, ε, ισχυρά παραδείγματα, ε, υποδείγματα που δεν υπάρχουν απαραίτητα για τους νέους ανθρώπους στις χώρες αυτές. Και κάτι που δεν ανέφερα είναι το θέμα της διατροφής. Δεν μπορούμε να έχουμε μια, μια εργατική τάξη που είναι ευημερή εφόσον δεν υπάρχει ισχυρή υγεία και πολιτική διατροφής από τις πρώτες χίλιες μέρες ε, ζωής ενός παιδιού. Εμείς δεσμευόμαστε στον τομέα της ε, διατροφής 3,5 ε, δις για την περίοδο 2015-2020 είναι η δέσμευσή μας και έχουμε ένα μηχανισμό παρακολούθησης ό,τι αφορά διατροφή. Έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά standing επίσης, 40-45% πρέπει να τα μειώσουμε. Θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα λοιπόν στην περιοχή, στην πολιτική διατροφή, ώστε τα παιδιά να μεγαλώνουν όπως πρέπει και σε συνθήκες υγιής. διότι έχουμε και φαινόμενα ανανισμού πολύ σημαντικά στην Ήπειρο. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τακτικά την Επιτροπή αυτό και πολύ συχνά μιλούμε για την ανάπτυξη αυτής της περιοχής και να εξασφαλίσουμε και την υλοποίηση των δικών μας στόχων ανάπτυξης με τη διαφύλαξη φυσικά κάποιων αξιών και χωρίς διακρίσεις. Νομίζω ότι αυτό το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι παράδειγμα προς και παγκοσμίω. Και στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου και στο στην συνάντηση του Buenos Aires θα λάβει μέρος, ε, εκ μέρους της Επιτροπής μας η κυρία Μαγκίνες. Οπότε έχουμε πολλά θέματα προς συζήτηση. Δεν πρόκειται να τα διεκπαιρεώσουμε με την σημερινή μέρα. Και μερικές φορές ακούγονται επικρίσεις ε, ε, κατά της κοινής γεωρικής πολιτικής αλλά όπως είπε και ο κύριος Κλάρκ, η κοινή γεωρική πολιτική σε καμία περίπτωση δεν είναι αντιαφρικανική πολιτική, ούτε έχει δυσμενή αποτελέσματα για την Αφρική, παρά την ε, ε, γνώμη που δημιουργήθηκε κάποιες φορές. Πρόεδρε, θα ήθελα να πω το εξής, ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να ε, συνεργαστούμε κυρίως εκεί όπου πολλοί ισχυρίζονται ότι η γεωρική πολιτική προκαλεί προβλήματα στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ε, έχουμε μειώσει τις επιστροφές των εξαγωγών. Εγώ επισκέπτηκα πάρα πολλές χώρες όταν πραγματικά προκαλούσε ζημιά και νομίζω ότι θα πρέπει κάπως και εμείς να ανταμυφθούμε για τις μεταρρυθμίσεις που μεταξύ εφαρμόζονται. ευχαριστώ λοιπόν πολύ που το επισημάνατε. Ναι. Πολύ σωστά και ήταν καλό το σχόλιο για να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ τους δύο διευθυντές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως κρατήσαμε σημειώσεις από τη συζήτηση και θα τις διαβάσουμε προς τους υπόλοιπους συναδέλφους. Συνήθως δεν έχουμε πρόβλημα με την παρουσία στην Επιτροπή μας πάντως δεν διατυπώθηκαν παρατηρήσει για τις αποφάσεις των συντονιστών και αν μέχρι την γνωστή διορία δεν υποβληθούν παρατηρήσεις θα θεωρηθούν ως συγκεκριμένες οι αποφάσεις των συντονιστών. Και μην ξεχνάτε ότι Τετάρτη το απόγευμα στις 7 θα έχουμε έκτακτη συνάντηση με τον Επίτροπο Χόγκαν όπου θα μας παρουσιάσει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2020. Αυτή είναι η παρουσίαση της ανακοίνωσης. Στη συνέχεια θα έχουμε συζήτηση για τη διαμόρφωση των ε, ε, απόψεών μας. Και φυσικά θα ακολουθήσουν και δημοσιονομικές προτάσεις στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των δημοσιονομικών προοπτικών. Πάντως, η μέρα Τετάρτη 29 του μηνός, σε 7 το απόγευμα, θα έχουμε την έκτακτη συνάντηση. Ε, γίνονται δεκτές και οι αποφάσεις των συντονιστών. Πολύ σωστά μου το υπενθύμησε και ο Γενικός μας Γραμματέας. Σας εύχομαι καλό μεσημέρι, καλή επάνωδο στις πατρίδες σας, στα σπίτια σας. Ε, πέμπτη είναι, ουσιαστικά ολοκληρώνεται η εργάσιμη εβδομάδα. Ε, και εις το επανειδήν.